Welcome everybody. Καλώς ήρθατε. Καθίστε παρακαλώ και θα έρθουν και άλλοι βουλευτές. Ξέρω πως ε, είναι δύσκολο Δευτέρα πρωί να έρθουν ε, οι συνάδελφοι από τις πιο απομακρυσμένες γωνίες της Ένωσης. Θα δούμε λοιπόν τα τυπικά. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Υποθέτω πως εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στο σημείο 2, ανακοινώσεις της Προέδρου και υπάρχουν κάποιες. Πρώτα απ' όλα για την συναπόφαση μετά την ψηφοφορία στις 13 Απριλίου για την Οδηγία 97-9 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την αποζημίωση των επενδυτών ο εισηγητής είπε πως θα πάει σε διαπραγματεύσεις για μια πιθανή συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση επί του φακέλου αυτού που αποτελεί προτεραιότητα της Επιτροπής μας. Σύμφωνα λοιπόν με τις διαδικασίες μας θα έχουμε ως διαπραγματευτική εντολή την έκθεση και βεβαίως η διαπραγματευτική ομάδα θα είναι η πρόεδρος, ο εισηγητής και οι σκιώδεις εισηγητές όπως γίνεται συνήθως. Κατόπιν ο άτυπος τριμερής διάλογος για το short selling στις 13 ε, Απριλίου. Η διαπραγματευτική ομάδα μας ζήτησε άτυπο διάλογο με την Ουγγρική Προεδρία για να συζητήσουμε τα επόμενα διαδικαστικά βήματα για μια συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Η διαπραγματευτική ομάδα συμφώνησε μετά να περιμένουμε μέχρι το Συμβούλιο Κοφήν της 17ης Μαΐου έτσι ώστε η Προεδρία να μπορέσει να βρει μια συμφωνία στο Συμβούλιο και να συγκληθεί η επόμενη τριμερή συνάντηση στις 23 Μαΐου. Βεβαίως, εάν δεν υπάρξει συμφωνία, μπορεί να ακολουθήσουν διαφορετική πορεία τα πράγματα. Για το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης ε, και το αποτέλεσμα της πρώτης ε, συνεδρίασης ε, της 20ης Απριλίου, εξήγησα στο Συμβούλιο την εντολή που είχε δώσει η Επιτροπή οι εισηγητέ και σκιώδη εισηγητέ εξήγησαν πώ θα αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά ω πακέτο και επιπλέον είπαμε πω το Συμβούλιο θα πρέπει να είναι δημιουργικό στην αναζήτηση λύσεων και αναμένουμε να κινηθεί πρώτα το Συμβούλιο σε κάποια ζητήματα. Συμβούλιο και Κομισιόν τόνισαν τη σημασία των νομοθετικών προτάσεων και εξέφρασαν το ότι θέλουν να εργαστούν σκληρά για να βρουν συμβασμούς με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνήσαμε όλοι να ξεκινήσουν οι ουσιαστικές συζητήσεις ε, στα οριζόντια, επί οριζόντιων ζητημάτων στην επόμενη συνεδρίαση που θα λάβει χώρα αύριο 3 Μαΐου 9 με 12 και μετά Τετάρτη 4 Μαΐου από τις 3 ε, μέχρι τις 6. Οπότε αυτές είναι οι ανακοινώσεις όσον αφορά τους τριμερείς ε, διαλόγους και τώρα είναι μεγάλη μου χαρά το ότι περνάμε σημείο 3, δημόσια ακρόαση με τον Μέρβιν Κίνγκ και τον Ανδρέα Ενρία, αντιπροέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συστημικού Κινδύνου. Η ακρόαση αυτή λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το άρθρο 5.4 του κανονισμού και οι αντιπρόεδροι πρέπει να παρουσιάσουν στην Επιτροπή μας το πώς σκοπεύουν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τον κανονισμό. Η ακρόαση θα γίνει ως εξής. Θα γίνουν κάποιες αγωγικές παρατηρήσεις πρώτα απ' όλα από τον πρώτο αντιπρόεδρο, τον κύριο Μέρβιν Κίνγκ για 5 λεπτά, μετά εισαγωγικές παρατηρήσεις από τον δεύτερο αντιπρόεδρο, τον κύριο Ενερία για 5 λεπτά και μετά θα περάσουμε σε μια σειρά ερωτήσεων τρεις στον κύριο Κίνγκ και τρεις στον κύριο Ανρία και ούτω καθεξής. Σαν την ε, διαδικασία νομισματικού διαλόγου. Να σας υπενθυμίσω λοιπόν πως αν ξεπεράσετε το ένα λεπτό ε, θα έχουμε λιγότερο χρόνο για τις απαντήσεις. Οπότε σας παρακαλώ μην θέτετε πολλαπλές ερωτήσεις που είναι αδύνατο να απαντηθούν εντός του χρόνου. Και αν το κάνετε αυτό τότε θεωρώ πως σωστό είναι οι ερωτήσεις αυτές να μην απαντηθούν. Καλώς ήρθατε, λοιπόν, κύριε Κίνγκ, και έχετε τον λόγο για 5 λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που έχω να στην Επιτροπή σας απόψε και να κάνω μια σύντομη εισαγωγική δήλωση. Η πρόσφατη τραπεζική και χρηματοπιστωτική κρίση είχε συντριπτικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή οικονομία. Το συνολικό ΑΕΠ είναι 5 με 10% χαμηλότερο από αυτό το οποίο θα ήταν εάν ακολουθούσε τις τάσεις πρώτης κρίσης και το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα εξακολουθεί να χρειάζεται ακόμα περαιτέρω επισκευές. Η μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και στη δομή και στους κανονισμούς είναι ουσιαστική για να αποφύγουμε περαιτέρω κρίσεις. Ένα αποτελεσματικό, ένας αποτελεσματικός και ανταγωνιστικός τέτοιος τομέας είναι βασικό συστατικό μιας επιτυχούς οικονομίας. Αλλά ένα από τα βασικά διδάγματα της κρίσης είναι πως ε, οι ισολογισμοί του τραπεζικού συστήματος επεκτάθηκαν μέχρι του σημείου ώστε να αποτελέσουν σημείο ε, αστάθειας στην ευρύτερη οικονομία. Οπότε, μία από τις αποστολές του νέου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ε, Συστημικών Κινδύνων είναι να δούμε τους κινδύνους στο ευρύτερο σύστημα. Το... Η Επιτροπή μας λοιπόν έχει κάνει κάποια σημαντικά πρώτα όπως ξέρετε. Ήδη έχει συνεδριάσει το Γενικό Συμβούλιο δύο φορές φέτος και θα συνεδριάσει και τον επόμενο μήνα. Η ΔΕ Ρυθμιστική Επιτροπή, στην οποία βρίσκομαι και εγώ, ε, συνεδριάζει και παρουσιάζει το έργο της στο Γενικό Συμβούλιο. Υπάρχει άρα και η Τεχνική Συμβουλευτική Επιτροπή που μας βοηθά στο έργο μας και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής έχουν ήδη οριστεί. Στο μέλλον η Επιτροπή μας έχει τρεις κυρίες προκλήσεις. Πρώτα απ' όλα να εξετάσουμε και αν χρειαστεί να προβούμε σε Προειδοποιήσει και συστάσεις. Υπάρχουν ακόμη πάρα πολλοί κίνδυνοι στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η κρίση δημοσίου χρέου και οι ανισορροπίε σχετίζονται με αυτό εντό της ευρωπαϊκής οικονομίας και η ζήτηση η οποία πλέον δεν μπορεί να διατηρηθεί καθώς προκύπτει από πάρα πολύ χαμηλά πραγματικά επιτόκια. Είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα. Είμαι πεπισμένος λοιπόν πως η Επιτροπή μας δεν θα αποφύγει αυτά τα προβλήματα και εξεπλάγει από την θετική αποφασιστικότητα πολλών ανθρώπων που λαμβάνουν τις αποφάσεις που μέχρι στιγμής έχει επιδειχθεί συνεδριάσεις. Κατόπιν, τα μέσα πολιτικής της Επιτροπής μας πρέπει να οριστούν. Εφόσον δεν έχουμε κάποιες δεσμευτικές εξουσίες, η ανάλυση και τα επιχειρήματα που θα αναπτύσσει πρέπει να είναι του υψηλότερου επίπεδου εάν η αρχή που ακολουθούμε, δηλαδή θα πρέπει να συμμορφώνονται ή να μας εξηγούν, ε, είναι να εφαρμοστεί. Βεβαίω ε, εμείς ε, δεν περιοριζόμαστε όσον αφορά τις στάσεις μας στις εθνικές αρχές. Σας πάρουμε ένα παράδειγμα σύμφωνα με τον κανονισμό κεφαλαϊκής ε, επάρκειας, η maximum εναρμόνιση δεν θα περιόριζε μόνο τα αντικυκλικά αυτά μέτρα, αλλά και τα μέσα που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Σε κάποιες περιπτώσεις, τέτοια περιορισμένα μέσα θα μπορούσαν να είναι πάρα πολύ περιοριστικά και αδύναμα για να μην υπάρχει υπερβολική συσσόρευση κινδύνου και μόχλευσης. Θα ήταν περίεργο εάν ένας ευρωπαϊκός φορέας άθελά του εμπόδιζε κάποιον άλλον να εκπληρώσει το καθήκον του. Τρίτον, η Επιτροπή μας θα πρέπει να συνεργαστεί στενά με τις τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και ο συναδελφός μου, ο Ανδρέα Ανρία, θα μας πει περισσότερα από αυτού. Οπότε, να συνοψίσω λέγοντας πως στον ρόλο μου ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής σκοπεύουμε να αξιολογήσουμε τους κινδύνους στην ε, ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική σταθερότητα και, ακόμη σημαντικότερο, να δράσουμε. Και είμαι στη διάθεσή σας σήμερα για να απαντήσω τυχόν ερωτήσεις για το έργο της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Thank you very Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν πολύ αποτελεσματικός. Περνάμε στην επόμενη παρουσίαση του Ανδρέα Ενρία, ο οποίος πρέπει να έχει βαρεθεί να με βλέπει, γιατί είναι η τέταρτη, τέταρτη φορά σε λιγότερα από τέσσερις εβδομάδες. Ανδρέα, λοιπόν, έχετε τον λόγο. Dear Madam Chair, dear... Ευχαριστώ πολύ, αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί ε, βουλευτές. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου προσφέρετε να Έλθω στην Επιτροπή σας ως δεύτερος αντιπρόεδρος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συστημικού Κινδύνου. Ο ρόλος μου στην Ευρωεπιτροπή μας προέρχεται από τη θέση μου ως ε, Προέδρου της Κοινής Επιτροπής ε, της Ευρωπαϊκής, των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και θα επικεντρώσω λοιπόν τις παρατηρήσεις μου στην ανάγκη να υπάρχει μια ομαλή διασύνδεση μεταξύ μικροπροληπτικής και μακροπροληπτικής ε, τραπεζικής εποπτείας. Σημαντική, κάτι σημαντικό που πρέπει να αντλήσουμε από όλα αυτά ενώ δεν υπήρξαμε αρκετά αποτελεσματικοί για να εντοπίσουμε νέους νέες πηγές συστημικού κινδύνου και να αντιδράσουμε. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η μακροπολιτική εποπτεία δεν ωφελήθηκε παρκώς από τη συνεισφορά των υποπτικών αρχών. Έχουμε με την υποστήριξη των τραπεζικών ελεγκτών κάνει διάφορες ε, συλλογές δεδομένων, αλλά μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Η μακροπροληπτική ανάλυση επίσης θα πρέπει να βασίζεται και σε στοιχεία τα οποία συλλέγουμε μέσω των ε, τακτικών ε, αξιολογήσεων κινδύνου που γίνονται από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και από τη συλλογή διαφόρων πληροφοριών και από άλλες ε, πηγές. Πρόσφατα, οι εποπτικές αρχές συμμετείχαν σε κάποιες αξιολογήσεις κινδύνου ιδίω εντό διασυνοριακών ομάδων, αλλά πρέπει να γίνει μεγαλύτερη πρόοδο ώστε τα στοιχεία αυτά να έχουν κάποια σημασία στη μακροπολιτική ανάλυση για να δούμε ποια είναι τα τροτά σημεία και ποιοι είναι οι δυνητικοί κίνδυνοι για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Το νέο λοιπόν Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτική Εποπτεία αντιμετωπίζει το θέμα αυτό. Βλέπουμε ότι το, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου έχει μια ευρεία σύνθεση. Γι' αυτό θέλουμε να έχουμε έναν επικοδομητικό, επικοδομητικό αμφίδρομο διάλογο με τι κεντρικέ τράπεζε και τι εποπτικέ αρχέ και η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή θα συνεισφέρει και αυτή στον εντοπισμό και την ανάλυση κινδύνων. Πρέπει λοιπόν να, να σας πω ότι υπάρχουν και σαφείς διατάξεις για να υπάρχει μια ομαλή ανταλλαγή πιστευτικών πληροφοριών και επίσης οι ε, μεμονωμένοι οργανισμοί κατόπιν ετοίμως μπορεί να δώσουν τα στοιχεία τους ε, στην Επιτροπή μας. Υπάρχουν πάντως και προκλήσεις. Πρώτα απ' όλα οι ελεγκτέ έχουν ε, τι άμεσε επαφέ με του χρηματοπιστωτικού οργανισμού, αλλά μπορεί να μην έχουν την μακροπροληπτική προοπτική για να υπάρχουν τα κατάλληλα στοιχεία, οι κατάλληλε συνεισφορέ. Και επίση τα αιτήματα για εποπτικέ πληροφορίε μπορεί να επιβαρύνουν την όλη εποπτική διαδικασία και να δοθεί έτσι εντύπωση ότι η μακροπροληπτική ανάλυση τελικά ε, έρχεται σε αντίθεση με τις τακτικές εποπτικές δραστηριότητες και δεν τις υποστηρίζει. Δεύτερη έλλειψη είναι ότι δεν υπάρχουν μηχανισμοί επιβολής. Ε, ναι, ε, έχουν οριστεί οι κίνδυνοι για χρηματοοικονομική σταθερότητα, παρόλα αυτά δεν υπήρχαν, είδαμε το, τα μέσα για να υπάρξει έγκυρη πολιτική δράση. Επίσης, το νέο θεσμικό πλαίσιο ε, δίνεται σωστή απάντηση και σε αυτή την περίπτωση. Οι κανονισμοί που θεσπίζουν και την Ευρωπαϊκή Χρηματοστοπτική Αρχή και το, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου προβλέπουν και ένα μηχανισμό παρακολούθησης των προειδοποιήσεων και των συστάσεων της ε, Επιτροπής μας. Και η ΕΣΑ επίσης δραματίζει ένα σημαντικό ρόλο για την ε, διατύπωση κάποιων μέτρων και για τη διαδικασία της παρακολούθησης. Για να έχουμε λοιπόν ομαλή αλληλεπίδραση μεταξύ μακροπροληπτικής, μικροπροληπτικής διάστασης ε, ε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε διάφορες ε, προκλήσεις. Είναι σημαντικό να συμμετάσχουν οι ελεγκτές στις αποφάσεις, να στηρίξουν την, τις διαδικασίες διατύπωσης προειδοποιήσεων και συστάσεων, ώστε να δοθεί απαραίτητη απάντηση και να ληφθούν τα μέτρα για την αποτελεσματική επιβολή. Βέβαια το σημαντικό είναι οι μηχανισμοί ε, δράσης ή εξήγησης, actor explain, να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και να έχουμε ακόμη και δημόσιες αναγγελίες ή δηλώσεις των νομολόγων για να ασκηθεί πίεση. Τρίτη έλλειψη που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι η συστημική κίνδυνη εκτός του ρυθμισμένου τομέα. Και σε αυτή την περίπτωση και η Ευρωπαϊκή Χρηματοπιστική Αρχή αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου έχουν αντιμετωπίσει σημαντικέ προκλήσει. Πρώτα απ' όλα, διαθεσιμότητα δεδομένων. Πολύ λίγα δεδομένα. Αλλά ακόμα και αν υπάρχουν δεδομένα, είναι δύσκολο να ε, μπορέσει να διευρυνθεί το πεδίο ρύθμισης και βέβαια θα πρέπει να είναι γρήγορη η χρηματοπιστωτική καινοτομία όταν έχουμε δηλαδή πέρασμα κινδύνων σε μια μη ρυθμισμένη, σε ένα μη ρυθμισμένο τομέα, να επεκτείνεται η ρυθμιστική κάλυψη. Η αποτελεσματική λειτουργία του ε, μακροπολιτικού ελέγχου είναι πολύ σημαντικό εγχείρημα και βέβαια για να στεφτεί με επιτυχία θα πρέπει να υπάρχει ομαλή αλληλεπίδραση με τις εμποπτικές αρχές. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Uh, σας ευχαριστώ και οι δυο σας στηρίσατε το χρόνο. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Και τώρα θα περάσουμε σε ένα γύρο ερωταπαντήσεων. Ένα λεπτό η κάθε ερώτηση και τέσσερα λεπτά οι απαντήσεις. Πρώτη ερώτηση από τον Ζαν Πολ Γκοζές, από το ΕΛΚΑ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς ε, να σας καλωσορίσω γιατί είναι η πρώτη φορά που με την ιδιότητά σας έρχεστε εδώ να θυσιαστείτε εντό αγωγικών μπροστά στους ευρωβουλευτές και να απαντήσετε στις ερωτήσεις τους που ελπίζω να είναι εύστοχες ε, κατά το δυνατόν. Σε σχέση με τα όσα είπατε και οι δύο και σε ό,τι αφορά τις κανονιστικές διατάξεις και σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις που θα πρέπει να διορθωθούν τα επόμενα χρόνια, θέλω να σας θέσω ένα πολύ απλό ερώτημα και συγκεκριμένα αν σήμερα θεωρείτε ότι έχετε στη διάθεσή σας τα απαιτούμενα μέσα σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό και τον προπολογισμό ώστε να φέρετε σε πέρα στην αποστολή που μας περιγράψατε. Σας ευχαριστώ. Θα μου επιτρέψετε να απαντήσω στα αγγλικά γιατί αυτή είναι η επίσημη γλώσσα τη επιτροπή μας και φαντάζομαι και οι συνάδελφοι μου θα ακούνε πολύ προσεκτικά αυτά τα οποία λέω. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε τις απαραίτητε δυνατότητε. Η πραγματική πρόκληση που αντιμετωπίζουμε δεν είναι τόσο το μέγεθος του προπολογισμού ή του ανθρώπινου δυναμικού, γιατί έχουμε ε, ε, επαρκείς ε, ιδιαίτερα ικανούς ε, συνεργάτες 25 ε, ε, συγκεκριμένα απαρτίζουν τη γραμματεία. Κατά την άποψή μου, το μεγαλύτερο πρόβλημα, η πρόκληση γενικά για την εποπτεία είναι η ποιότητα των απόψεων που εκφράζεται. Το θέμα δεν είναι κατά πόσο υπάρχουν όλες τις λεπτομέρειες και αυτό γίνεται, αλλά στη τελική ανάλυση αυτό που μετράει είναι κατά πόσον για να έχουμε σωστή απόφαση υπάρχει βούληση, η αποφασιστικότητα και η ανάλυση. Κατά δική μου λοιπόν άποψη το ατού της ε, Επιτροπής μας ε, είναι ότι συγκεντρώνει, συναθρίζει όλους ε, τους προέδρους κεντρικών τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλοι αυτοί ως ομάδα καλούνται να καταλήξουν σε μια κοινή απόφαση. Εάν λοιπόν δεν κατορθώσουμε να καταλήξουμε σε μια απόφαση, σε μια αξιολόγηση, αυτό λέει πάρα πολλά για την ε, ανεπάρκεια των αποφάσεων που λαμβάνουν μεμονωμένα άτομα στις, ευρωπαϊκές, στην κεντρική, στις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών. Θέλω λοιπόν να υπογραμμίσω ότι δεν πρόκειται για θέμα χρημάτων ή αριθμό ατόμων, δεν παίζεται εκεί το παιχνίδι, αλλά η ποιότητα της αξιολόγησης. Η αποφασιστικότητα επίσης όταν προκύπτει μια αξιολόγηση αυτή να μεταφράζεται στην πράξη. Και εδώ χρειαζόμαστε την υποστήριξή σα, γιατί μερικέ φορές η Επιτροπή μας ε, καταλήγει σε αποφάσεις ε, που δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε την υποστήριξη του Κοινοβουλίου που θα μας δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε ορισμένους ε, τομείς που ξέρετε πολύ καλά ότι πολύ συχνά εκεί έχουμε να αντιμετωπίσουμε τεράστιες αντιστάσεις από ομάδες πίεσης και εκεί ακριβώς χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Φαντάζομαι, Πολ, είστε ευχαριστημένος με την απάντηση. Κατόπιν τούτου, Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Δεν βλέπω την Πρεβάνς, τον Πίτερ βλέπω. Εκ μέρους ε, της ομάδας S&D από τον κύριο Σκίνερ, τους σοσιαλιστές και οι δυο σας ε, είσαστε τραπεζίτες, προφανές αυτό. Έχετε ε, τρεις αρχές ε, τις ασφαλιστικές αγορές ε, ε, τράπεζες ε, και έχετε και 25 ιδιαίτερα ικανούς συνεργάτες στη γραμματεία. Και θα καταλάβετε τώρα προς τα πού θέλω να κατευθύνω την ερώτησή μου. Εμείς που είμαστε στο Κοινοβούλιο και πολλοί ξέρουν ότι εγώ ασχολούμαι τα ασφαλιστικά, γι' αυτό χαμογελούν. Από εμά περιμένετε πληροφορίες ε, που πολλές φορές ε, ε, προκύπτει και κάποια επικάλυψη των πληροφοριών αυτών. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται πολλές φορές ίσως να αντιφάσκουν σε τελική ανάλυση. Έχετε σκεφτεί πώς ακριβώς θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο η Κοινή Επιτροπή. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει καμία σύγκρουση. Διότι κατά την άποψή μου ένα από τα μεγάλα προβλήματα που υπήρχε πριν προκύψει η χρηματοπιστωτική κρίση ήταν ότι η νομισματική ένωση είχε μόνο ένα εργαλείο, τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια, για να αντιμετωπίσει τη σταθερότητα των τιμών αλλά και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματο. Και δεν γινόταν να αντιμετωπιστούν και τα δύο προβλήματα με ένα μόνο εργαλείο. Ναι για την ε, σταθερότητα των τιμών, όχι όμω για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνο και η μόχλευση στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι τα μικροπροληπτικά προληπτικά εργαλεία ε, που προτείνονται από την Επιτροπή μας και θα εφαρμοστούν από τις Εθνικές Αρχές αποτελούν προσθήκη ε, της βεντάλιας των εργαλείων. Και δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υπάρχει σύγκρουση. Μάλιστα πριν από την κρίση, αν υπήρχε ένα ε, οπλοστάσιο ε, μικροπροληπτικών εργαλείων, ε, τότε ε, δεν θα υπήρχε αυτή η υπερβολική επέκταση των τραπεζών, η έκθεσή τους και αυτό θα ήταν ευπρόσδεκτο από πλευρά νομισματική. Όσον αφορά τι ασφάλειες, διαφέρουν πολύ από τις τράπεζες, Ίσως κατά καιρού να υπάρχουν συστημικοί κινδυνοί, καμία σχέση οι ασφάλειες ε, με τις τράπεζες, γι' αυτό και δεν πρέπει να συγχαίονται. Και πάλι δεν βλέπω να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την έννοια ότι οι ελεγκτές και όσοι βρίσκονται στην ε, δική μας την Επιτροπή γνωρίζουν πολύ καλά τις ε, διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις τράπεζες και τις ασφάλειες και τους συστημικούς κινδύνους που μπορούν να προκαλέσουν αυτοί οι δύο τομείς. I think Πάμε επόμενη, στον επόμενο γύρο των ερωτήσεων. Ε, αν δεν θέλετε να την υποβάλλετε τώρα την ερώτησή θα την συγκρατήσετε για αργότερα, για να μην την ξεχάσετε. Επόμενη λοιπόν ερώτηση, ε, Σιλβί Κούνατ, εκ μέρους των Φιλελευθέρων. Η Σιλβί παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. θα μιλήσω γαλλικά γιατί ναι μεν είναι η γλώσσα εργασίας της Επιτροπής σας ε, τα αγγλικά, αλλά ο εισηγητής μας ήταν ε, Γάλλος. Λοιπόν, ε, μια ευρωπαϊκή πτυχή των καθηκόντων σας. Όταν διαπραγματευτήκαμε με το Συμβούλιο, είχαμε να αντιμετωπίσουμε τις κυβερνήσεις απέναντί μας, οι οποίες σε σχέση με το κείμενο της Κομισιόν και τη βούληση του κυρίου Ντελαροσιέρ, ήθελα να μπει η ρήτρα διασφάλισης για την περίπτωση που θα προέκυπτε ότι αποφάσεις που λαμβάνονται από τις ευρωπαϊκές αρχές θα μπορούσαν να οδηγήσουν ένα κράτος μέλος να λάβει μέτρα που θα επηρεάσουν τον προπολογισμό του. Θέλω να σας θέσω λοιπόν το εξής ερώτημα. Προφανώς ε, βρισκόμαστε σε μια κρίση όπου η κατάσταση των τραπεζών και των δημόσιου χρέους αλληλοτρέφονται και δημιουργούν αυτό το πρόβλημα στο το οποίο αντιμετωπίζουμε. Εάν κληθείτε από συστημική πλευράς να διαπιστώσετε ότι οι δοκιμές κόπωσης, τα stress test ζητούν επανακεφαλαιοποίηση. Άρα, μιλάμε για δημόσια χρήματα. Τι θα κάνετε εσείς ο Αντιπρόεδρος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συστημικού Κινδύνου. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Νομίζω ότι δύο απαντήσεις μπορώ να δώσω σε αυτή την ερώτηση. Η πρώτη απάντηση είναι ποιος είναι ο ρόλος ε, της Επιτροπής μας στις δοκιμές αντοχής, αυτά τα stress test που θα συμμετέχουμε, πρέπει να σας πω σίγουρα, ε, και στην ε, αξιολόγηση από ομοτήμου στο peer review. Θα συμβουλευτούμε τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες για αυτές τις δοκιμές αντοχής και ο Αντρέα θα σας πει και τα αποτελέσματα ε, των δοκιμών αυτών αργότερα. Πάντως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα αποτελέσματα των ε, stress test και να δούμε ε, κατά πόσον έχουμε αυτά τα προβλήματα στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Το δεύτερο στοιχείο απάντησης αφορά την επανακεφαλαιοποίηση. Το έχουμε ξαναπεί και σε προηγούμενες συνέντευξεις τύπου, ότι εάν, και τονίζω τη λέξη εάν, χρειαστεί επανακεφαλαιοποίηση κάποια τράπεζα στην Ευρώπη, τότε πρέπει η αρμόδια εθνική αρχή να είναι έτοιμη όταν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του stress test να έχει ένα σχέδιο για το πώ είτε οι τράπεζε είτε οι εθνικέ αρχέ θα προβούν σε αυτή την επανακεφαλαιοποίηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα ήταν όλο ατυχέ να έχουμε ένα stress test και μετά να υπάρχει κενό μεταξύ ανακοίνωση του αποτελέσματο και διατύπωση του σχεδίου για την αντιμετώπιση των σημαντικών προκλήσεων που θα απορρέουν από την ανάγκη επανακεφαλαιοποίηση. αλλά ε, δεν είναι δική μα αρμοδιότητα. Είναι αρμοδιότητα των εθνικών κυβερνησεών. Από πλευρά όμω στρατηγική, εμεί η Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου έχουμε πει ότι σε περίπτωση που δημοσιοποιηθούν, όπω και θα γίνει αυτό στο δεύτερο μέσο του Ιουνίου, τα αποτελέσματα των stress test, τότε θα πρέπει να είναι έτοιμε εθνικέ αρχέ να προβούν στην ανακεφαλαιοποίηση όλων των τραπεζών για τις οποίες κάτι τέτοιο θα καταστεί αναγκαίο. Και ένα σχόλιο για τα stress test που πάντοτε τα ε, παρουσιάζουν κανείς ως ε, ένα μαχαίρι μαχαίρι ή περνά κόβεσαι. Αυτό που κάνουν ουσιαστικά τα stress test είναι θέτουν ερωτήματα. What if, τι θα συμβεί εάν γίνει αυτό και εκείνο. Για σενάρια πρόκειται και με τα σενάρια αυτά και τις ερωτήσεις αυτές θέλουμε να ε, αξιολογήσουμε τις αδυναμίες των ε, τραπεζών. Δεν ξέρουμε αν τα σενάρια θα επιβεβαιωθούν. Δεν θα πρέπει λοιπόν να τα δούμε ως εξετάσεις αυτά τα stress test, περνάς ή κόβεσαι. Απλά θα δώσουν στοιχεία που είναι πάρα πολύ απαραίτητα, γιατί δεν μπορούμε να αγνοήσουμε κάποια στοιχεία. Όταν αποτύχουν κάποιες τράπεζες, αυτές οι τράπεζες ίσως χρειαστούν περισσότερο κεφάλαιο για να προχωρήσουν. Περί αυτού πρόκειται, δεν είναι ότι αποτυγχάνουν και καταραίουν. Θεωρούμε λοιπόν επίσης ότι θα είναι ε, μια ε, τακτική, ένα τακτικό τμήμα, μόνιμο τμήμα αυτής της εποπτικής διαδικασίας, ε, τα stress test. Θα πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα που κάτι θα έχουν να μας πούν για την ευαισθησία ή την τροτότητα κάποιων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και θα πρέπει να ενημερωθούν βέβαια γι' αυτό και οι ίδιες οι χρηματοπιστωτικές αγορές αλλά και οι κυβερνήσεις. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα σε ερωτήσεις ε, για τον ε, κύριο Αντρέα Η πρώτη ερώτηση και πάλι από τον Ζαν Πολ, εκτός αν θέλετε να περιμένετε να υποβάλλετε αργότερα την ερώτησή σας. Όχι, τα κάνω όλα σήμερα κυρία Πρόεδρε. Καλό είναι αυτό λοιπόν. Ουσιαστικά το ερώτημα αφορά και τους δύο αντιπροέδρους. Κάποιες φορές ε, κάνουμε κάποιες, αν θέλετε, προοπτικές μελέτες. Εγώ θέλω να μην πάμε προς το μέλλον, αλλά προς το παρελθόν. Αναδρομικά να σκεφτείτε αν η Επιτροπή σας υπήρχε πριν από δύο χρόνια. Τι θα είχατε αλλάξει, παραδείγματος χάρη, σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος. Είναι δύσκολο, αλλά ξέρετε πού καταλήξαμε σήμερα. Yes, thank you. Um, well, uh, Κοιτάξτε, το έχω σκεφτεί αυτό τι θα συνέβαινε κατά τη διάρκεια της κρίσης αν επικρατούσαν ε, νέοι κανόνες. Βέβαια το έχω σκεφτεί ομολογώ περισσότερο από την πλευρά των εποπτικών αρχών και κατά την άποψή μου υπάρχουν τα εξή θέματα. Θεωρώ ότι σε αυτή την περίπτωση θα είχαμε ίσως ε, τη δυνατότητα να έχουμε έγκαιρες προειδοποιήσεις ε, όπως ε, στον σκιώδη τραπεζικό τομέα. Θυμάμαι λοιπόν ότι υπήρξαν συζητήσεις ε, στις εποπτικές αρχές στην Κεντρική Τράπεζα ε, για το κατά πόσο είναι δυνατόν ε, να μετακυλιστούν κάποιες δραστηριότητες και ο συστημικός κίνδυνος που έχουν βέβαια άμεση σχέση με τις δραστηριότητες που αναπτύσσει η τράπεζα απέναντι στα κράτη-μέλη. Θεωρώ λοιπόν ότι τότε κρίναμε το εξής. Ίσως να υπήρχε κάποια συγκέντρωση κινδύνου, αλλά δεν το γνωρίζαμε. Και από τα στοιχεία που υπήρχαν, ίσως ε, να μπορούσε κανείς να καταλήξει ότι ο κίνδυνος είχε διαχυθεί στην ευρύτερη οικονομία και ίσως αυτό να σήμαινε κανονικά ότι τα συστήματα θα περισσότερο, θα είχαν μεγαλύτερη αντοχή γιατί θα είχε διαχυθεί περισσότερο κίνδυνος. Αυτό δεν το γνωρίζαμε τότε. Η ε, δική μας Επιτροπή ζήτησε και συγκέντρωσε περισσότερες πληροφορίες και εάν αυτό το είχαμε κάνει νωρίτερα, ίσως να είχε βοηθήσει να εντοπίσουμε καλύτερα την συγκέντρωση κινδύνου στην αγορά και βεβαίως ε, στην περίπτωση αυτή θα είχαμε εκδώσει προειδοποιήσεις για να μπορέσουμε να αλλάξουμε κάπως την κατάσταση. Μια άλλη δυνατότητα βέβαια θα ήταν να ε, ανακηρύξουμε την κατάσταση, κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τώρα η Επιτροπή μας μπορεί να ζητήσει από το Συμβούλιο να πράξει κάτι τέτοιο και στην περίπτωση αυτή οι εποπτικές αρχές θα έπαιρναν έκτακτες ε, αποφάσεις, αποφάσεις έκτακτης ανάγκης ε, που θα εφαρμόζονταν στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το ίδιο μπορεί να κάνει βέβαια και η υποπτική αρχή και μία καλή συνεργασία ανάμεσα στην Επιτροπή Συντημικού Κινδύνου και την, τις επιτροπές, της τραπεζικές αρχές θα ήταν πάρα πολύ καλή. Εκείνο που χρειάζεται δηλαδή είναι να είχαμε μία καλύτερα συντονισμένη αντίδραση ως απάντηση στην κρίση. Νομίζω ότι αυτό θα προσέφερε μεγάλη υπεραξία. Έχουμε τώρα μια σειρά ερωτήσεων και για τους δυο σας ε, για να τις απαντήσετε και επειδή ήσασταν αρκετά σύντομοι στι ομιλίε νομίζω ότι ε, τώρα μπορούμε να περάσουμε σε ερωτήσει. Αντρέα, ο Πίτερ ε, σα ρώτησε για την κοινή επιτροπή και τι ρόλο πιστεύετε ότι μπορεί να δραματίσει αυτή η κοινή επιτροπή, αν μπορείτε να μα πείτε τώρα. Πρώτα απ' όλα να σα πω ότι εγώ έχω ε, τραπεζικό υπόβαθρο, αλλά βεβαίως ως αντιπρόεδρος ε, της Επιτροπής Συστημικού Κινδύνου ε, είμαι και αντιπρόεδρος της κοινή Επιτροπής και την επόμενη χρονιά θα έρθουν άλλοι συναδελφοί μου που θα βρίσκονται στη δική μου τη θέση την πρώτη συνάντηση της ε, κοινή Επιτροπής την είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και ήδη σε κάποιο βαθμό συμβάλαμε στον πρώτο γύρο συζητήσεων ε, για τους ε, κινδύνους έχουμε μία διατομιακή έκθεση κινδύνων την οποία προσυπογράφουν και οι τρεις αρμόδιες αρχές. Παρότι λοιπόν πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι ακόμα απόλυτα ικανοποιημένος ε, για το ε, πώς ακριβώς εξελίσσεται η ε, διατομιακή αυτή έκθεση, παρόλα αυτά θεωρώ ότι προβάλλει απόψεις από πάνω προς τα κάτω αυτό που θα έπρεπε να γίνει στο τέλο να συμπληρωθούν όλε αυτέ οι απόψει και με τι απόψει των μεμονωμένων τομέων και των κλάδων. Πάντως έχει σημειωθεί κάποια πρόοδο και πράγματι κατά την πρώτη συνάντηση τη κοινή επιτροπή ε, πρέπει να συγκεντρώσουμε πληροφορίες από ανθρώπου που είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση κινδύνου σε διάφορου φορεί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη αξιολόγηση, καλύτερη σειρά αξιολογήσεων στην επόμενη συνάντηση που ε, θα λάβει η χώρα στου κόλπου τη της ε, Επιτροπής Συστημικού Κινδύνου. Μια άλλη ερώτηση τώρα προς τον κύριο Κίνκ. Δηλαδή, πριν από δύο χρόνια, ε, ποια θα ήταν η διαφορά που θα προέκυπτε σχετικά με την κρίση του δημόσιου χρέους. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το γνωρίζει κανείς και αναμφίβολα πριν από την κρίση, εάν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου, δεν θα εξετάζαμε το θέμα του δημόσιου χρέους, γιατί αυτό προέκυψε μετά την τραπεζική χρήση και όχι πριν από αυτήν. Ε, έτσι λοιπόν, εκείνο που πρέπει να πω είναι ότι θα μας απασχολούσε βέβαια αυτή η τεράστια έκθεση των τραπεζών. Και όπως είπε και ο Ανδρέα, οι κεντρικοί τραπεζίτες, ε, οι ελεγκτές ε, έκαναν πάρα πολλές ομιλίες ε, για το ότι τα πριν κινδύνου ήταν πολύ χαμηλά, ότι υπήρχαν ε, πάρα πολλά εργαλεία που επέτρεπαν ε, την αξιολόγηση με τα 3α και επίσης επανέλαβαν, ανέφεραν και πολλές φορές ότι υπήρχε υπερβολική μόχλευση. Όμως δεν ανέφεραν τις επιπτώσεις, γιατί σε όλες αυτές τις ομιλίες απλά όλοι αναφέρονταν στον χρηματοπιστωτικό τομέα και το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι αν κάποιος δεν μας άκουγε, απλά και εμείς να ξεχάσουμε τις απόψεις μας. Δεν υπήρχε κάποια αρχή που να εφαρμοστεί. Ε, νομίζω ότι η τράπεζά μας, η επιτροπή μας, ε, θα είχε δύο πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα σε σχέση με τα βουλήματα που διδάξαν τότε οι τραπεζίτες. Πρώτον, εμείς θα είχαμε το κύρος ενός πανευρωπαϊκού οργανισμού που θα μας στήριζαν όλοι οι ελεγκτές και οι τραπεζίτες ε, πίσω μας που θα έλεγαν ότι να, εδώ είναι ο κίνδυνος ή να, εδώ είναι μια σύσταση που πρέπει να λάβετε υπόψη. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερον, η αρχή της συμμόρφωσης ε, μας δίνει τη δυνατότητα ε, όχι μόνο να επιβάλλουμε να μην μας αγνοούν, αλλά και να υπεραμεινθούμε των απόψεών μας. Οι εθνικές αρχές πρέπει να μας ακούν πολύ προσεκτικά. Και νομίζω ότι αυτό θα αποτελούσε μια πολύ σημαντική βελτίωση σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε τότε. Αυτό όμως που σε τελική ανάλυση παίζει ρόλο είναι ο βαθμός πολιτικής δέσμευσης για να αντιμετωπίζει τα προβλήματα, κυρίω όταν τα πράγματα μοιάζουν να είναι καλά. Και ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε μετά την πολιτική κρίση ως συνεπακόλουθο της χρηματοπιστωτικής κρίσης είναι ότι ο τύπος, η πολιτική αλλά και οι βουλευτές θεωρούσαν ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας θα πήγαινε θαυμάσια με μεγάλη επιτυχία και δεν ήθελαν να ακούσουν προβλήματα που ενδεχομένως θα προέκυπταν αν υπήρχε τεράστια επέκταση. Έτσι λοιπόν ε, όταν η Επιτροπή επιθυμεί να εκδώσει μία προειδοποίηση, θέλουμε απαρέγκλητα την δική σας την υποστήριξη για να μας λάβουν σοβαρά υπόψη τους. Γιατί ε, ακόμα και να υπήρχε και η καλύτερη θέληση και αποφασιστικότητα στον κόσμο, αν δεν υπάρχει στήριξη δεν μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι ουσιαστικά. Παρόλα αυτά πρέπει να πω ότι η επέκταση των ισολογισμών είναι εκείνη που προκάλεσε το πρόβλημα, αλλά εκείνο που μετράει τώρα είναι να παρεμποδίσουμε την επανεμφάνιση των προβλημάτων. ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριοι Αντιπρόεδροι, το ερώτημά μου αφορά καταρχάς τον κύριο Κίνγκ, αλλά ίσως και ο κύριος Ενέρια θα μπορούσε να απαντήσει. Δύο ερωτήματα. Πρώτον, με την εγκαθίδρυση αυτής της νέας δομής, δημιουργήσαμε και αυτήν την Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή, στο πλαίσιο της οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μπορούν να παρεμβαίνουν στην όλη συζήτηση. Τι αναμένετε από τις δικές τους εργασίες, ποια, ποιες είναι οι προσδοκίες σας και πώς αντιλαμβάνεστε την οργάνωση, τη διάθρωση της Επιτροπής αυτής ώστε να αποτελέσει ένα αντίβαρο στην ε, άσκηση επιρροής από άλλους φορείς που γνωρίζουμε ότι ενίοτε με πολύ μεγάλο ταλέντο συνδυάζουν συγκρούσεις συμφερόντων, άσκηση πίεσης, ε, ε, άσκηση πίεσης κτλ. Δεύτερο ερώτημα. Βλέποντα τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η εποπτεία και αξιολογούνται οι κίνδυνοι, αντιλαμβανόμαστε ότι κυρίω το θέμα, το κριτήριο είναι η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Έχουμε όμω την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και πίσω από αυτό ε, έχουμε μακροοικονομικά αρμπιτράζ. Και δεν είναι μόνο το θέμα ο κίνδυνο χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Μα δεν μπορώ να επεκταθώ γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Ελπίζω να έχετε καταλάβει τι θέλω να πω. Εσεί απλά περιορίζεστε στο να παρακολουθείτε τη μακροοικονομική σταθερότητα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των κεφαλαίων Διότι από πίσω υπάρχουν μακροοικονομικές διαστάσεις που δεν έχουν να κάνουν μόνο με αυτό το διακύβευμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Περβάνς. Μία ερώτηση σε ένα λεπτό, όπως ξέρεις και εσύ ως Λοιπόν, Ανδρέα. Ναι, ε, βεβαίως για την εποπτεία, για την ενίσχυση της εποπτείας ε, και των κεφαλαίων αγορών. Ναι, βεβαίως υπάρχει αυτή η έμφαση στην ενίσχυση αυτή τη στιγμή της ε, ε, σταθερότητας και δικαίως γιατί είδαμε τη ζημία μπορεί να επιφέρει η πολύ σφιχτή εποπτεία στην ανάπτυξη. Το είπε αυτό ο Μέρβιν στην αρχική του τοποθέτηση. Οπότε εκεί πέρα πρέπει να στραφούμε στην ενίσχυση της στήριξης της ε, χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Και σας ευχαριστώ για το ερώτημά σας, γιατί θεωρώ πως ε, ενώ το Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο θα πρέπει τώρα να μεταφέρουν τις διεθνείς συμφωνίες σε ευρωπαϊκή, στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι να δούμε τι μπορούμε να διορθώσουμε στον τομέα της εποπτείας, να δούμε το τι δεν πήγε καλά κατά τη διάρκεια της ε, κρίσης. Και εκεί πέρα πρέπει να δοθεί περισσότερο βάρος. Όμως Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, πως βεβαίω ε, το θέμα δεν είναι μόνο χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Χρησιμεύουν και για άλλα πράγματα χρηματαγορές, αλλά νομίζω πως αυτό το έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια και βεβαίω αυτό φαίνεται και σε αυτά τα οποία λέει και, οι δύο, και αυτά που λένε και οι δύο ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές και, το, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου. Π.χ. όταν εκδίδουμε ανακοινώσει βεβαίω για τι εκτιμιστικέ πολιτικέ. Θα δούμε το τι επίπτωση έχουν και στην ανάπτυξη και στο οικονομικό σύστημα γενικότερα. Παραδείγματο χάρη όλη η δουλειά που έχει κάνει η Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου. Βασικό ε, στοιχείο αυτής της δουλειά είναι ακριβώς να να πάνε κόντρα στο ρεύμα. Αυτό το οποίο είπε και ο Μέρβιν. Δηλαδή να μπορούμε να δράσουμε όταν αυξάνεται ο κίνδυνος ενώ βρισκόμαστε σε μια ανωδική φάση του πιστοτικού κύκλου. Και όλα αυτά βεβαίως για να υποστηρίξουμε μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη. Τώρα για την Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή. Νομίζω πως ε, είναι πάρα πολύ σημαντική λόγω του εγχειρήματο που έχουμε εδώ πέρα να αντιμετωπίσουμε. Σημαντικό είναι λοιπόν το να έχουμε ανεξάρτητες ε, απόψεις και σοβαρή οικονομική ανάλυση που να υποστηρίζει το έργο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου και εγώ προσωπικά αναμένω πάρα πολλά. πήγε ο Μάρτιν Ελβίκ, ο πρόεδρος, ο πρώτος πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής μίλησε για τη συσσόρευση συστημικών κινδύνων εκτός του τραπεζικού τομέα εδώ και καιρό. Οπότε αυτό είναι πολύ πολύτιμο και θα είναι πολύτιμο βιώστο να έχουμε αυτές τις δομές και καλύτερο θα ήταν βεβαίω να τι είχαμε πρώτη ε, κρίση. Η διαδικασία επιλογής ε, των μελών της συμβουλευτική Επιστημονικής Επιτροπής ήταν πολύ εκτεταμένη και η διαδικασία λήψη αποφάσεων επίση ε, της επιτροπή Δημικού Κινδύνου πάρα πολύ λεπτή και σημαντική. Έχουμε λοιπόν αρκετούς, είχαμε αρκετές ε, αιτήσει υψηλή ε, ποιότητας και όλοι οι πανεπιστημιακοί που επελέγησαν πολύ ικανοί στην ε, χρηματοοικονομική ανάλυση και σε πολλούς τομείς, οπότε φαντάζομαι πως η συνεισφορά από την έρευνά τους θα είναι πολύτιμη για το έργο μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δύο ήταν αυτές οι ερωτήσεις και ξέρω βεβαίως πως η μία απευθύνονταν στον Μέρβιν Κίνγκ. Ίσως θα θέλατε να πείτε και εσείς κάποια πράγματα. Είμαι σύντομος. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Η εχμαλωσία αυτή των ρυθμιστικών αρχών είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει οποιοδήποτε ρυθμιστικό σύστημα προσπαθεί να υποπτεύσει κάποιους θεσμούς και βεβαίως η ισχύς αυτών των φορέων είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Γι' αυτό ακριβώ έχουμε ανθρώπου που δεν έχουν ε, συμφέροντα στον ε, κλάδο για να μπορέσουμε να έχουμε αντικειμενικές απόψεις. Εγώ ξέρω τον Μάρτιν Χέλβι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αν μου λέγατε πριν από ένα χρόνο τον... ποιον θα διάλεγα εγώ για ε, πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής θα διάλεγα αυτόν. Για ένα συνδυασμό Γνώσεις ε, του τραπεζικού τομέα, αριστεία στον πανεπιστημιακό τομέα και το σημαντικότερο για την ακαιρεότητά του. Και νομίζω πως θα συνεισφέρει πάρα πολύ. Όσον αφορά την υποπτία και τα ζητήματα που είπατε για τις ε, κεφαλαίες αγορές, θέλω να αναφέρω κάτι σύντομα. Νομίζω πως είναι λάθος να επαφιόμαστε πάρα πολύ στην εποπτεία. Υπάρχει ένα όριο στο τι μπορεί να επιτύχουν οι εποπτικές αρχές που είναι και αυτοί άνθρωποι τελικά. Δηλαδή, εάν οι άνθρωποι που διευθύνουν τη Citibank στη Νέα Υόρκη δεν αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που αναλαμβάνουν, ε, είναι απίθανο να το αντιληφθούν και οι υποπτικές αρχές. Πρέπει λοιπόν να δούμε και την δομή εξίσου με το ρυθμιστικό πλαίσιο και πρέπει να δούμε πως το τραπεζικό σύστημα το οποίο υπάρχει δίνει στους ανθρώπους και στις ε, χρηματαγορές τα σωστά κίνητρα για να συμπεριφέρονται λογικά. Μέσω της εποπτείας δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε λανθασμένες δομές που δίνουν στους ανθρώπους λάθος κίνητρα. Έτσι. Ε, δεν έχει κανένα νόημα οτιδήποτε και να κάνουμε. Οπότε ναι, είναι σημαντική εποπτεία, αλλά δεν αρκεί από μόνη της. Πρέπει να δούμε και τις δομές. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στο αρχικό μας πρόγραμμα, ε, στην ερώτηση δηλαδή από την Γκουλάτ προς τον Ανδρέα. Mr. King, thank you very much. Για τον κύριο Κίνγκ να πω ότι σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση που δώσατε, ήταν απόλυτα σαφής και ξεκάθαρη. Και έρχομαι στον κύριο Ερία. Λίγο πολύ το ίδιο ερώτημα θέλω να θέσω για τη σχέση μεταξύ ε, της κρίσης του δημόσιου χρέους και των τραπεζών. Φαντάζομαι ότι διερμηνεύω τις απόψεις πολλών συναδέλφων λέγοντας ότι εκτιμούμε τον τρόπο με τον οποίο εσείς ε, ε αντιμετωπίσατε το όλο θέμα τη οργάνωσης των stress test και ε, έχοντα μεγαλύτερε απαιτήσει από ό,τι πέρυσι. Και είπατε ότι περιμένετε από τα κράτη αυτά τα μέτρα, τα συγκεκριμένα μέτρα, έτσι, για να δοθεί συνέχεια στα αποτελέσματα των stress test. Σας ρωτώ λοιπόν πώς θα προχωρήσετε όταν θα έχετε στα χέρια σας τα αποτελέσματα γύρω στα τέλη Ιουνίου. Οπότε και θα πρέπει να έχετε ένα όραμα για το διοικητική Κίνγκ συμφωνώ ότι δεν είμαστε ε, σε μια προσέγγιση άσπρο ή μαύρο, αλλά υπάρχουν διαβαθμίσεις, υπάρχουν αποχρώσεις. Έχετε την εντύπωση ότι ορισμένα κράτη-μέλη ενδεχομένω τα μεγάλα, όπως τα αποκαλούμε κράτη-μέλη, θα διστάσουν και δεν θα θελήσουν να, επιτρέψουν σε μια ευρωπαϊκή αρχή να, να παρεμβαίνει σε σημαντικά εθνικά ζητήματα. Θα κάνετε συστάσεις, θα επιληφθεί η Επιτροπή σας και πρέπει να σας πω ότι προβλέπονται επίσης ε, και δυνατότητες ε, για το Κοινοβούλιο να ε, παρέμβει και αυτό. Λοιπόν, πώς αντιλαμβάνεστε τη συνέχεια στα stress test. Thank you Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Ακούστε, αυτές οι δοκιμές αντοχής πραγματικά με απασχολούν ε, πολύ και σε αυτά επικεντρώνομαι, σε αυτά τα ε, stress test. Τα δεδομένα σιγά σιγά έρχονται και αρχίζουμε να τα εξετάζουμε. Αν μου επιτρέπετε θα ήθελα σε αυτά τα τέσσερα λεπτά που έχω να επικεντρωθώ σε κάποια στοιχεία. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ε, συγκροτούμε μια ομάδα από εμπειρογνώμονες και από τις εθνικές αρχές και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου και από την ΕΚΤ. Θα υπάρξουν ε, συμφωνίες εμπιστευτικότητας ε, και οι επιρρογνώμενε αυτοί για ένα μήνα έως και έξι εβδομάδες θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και θα εξετάσουν τα αποτελέσματα των μεμονωμένων τραπεζών. Και αυτό είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην ε, Ευρώπη. Είναι η πρώτη φορά που οι εποπτικές αρχές μπορούν να ελέγχουν, να την παραβάλουν, να προβάλλουν και ενστάσει ενδεχομένω για τα αποτελέσματα, για τα στοιχεία κάποιων τραπεζών. Είναι κάτι καινούριο, εντελώ καινοφανέ και υπάρχει και η μεθοδολογία για να δώσει ε, πραγματικά συνεκτικά αποτελέσματα, αξιόπιστα αποτελέσματα αυτή η διαδικασία. Το ερώτημά σας είναι τι θα συμβεί αν τα αποτελέσματα δημοσιοποιηθούν πλέον και αν θα χρειαστεί να αναλυφθεί δράση, πώς θα Βεβαίω μου θα αναλυφθεί αυτή η δράση. Θα θυμάστε ίσως ότι είχαμε ζητήσει από τα κράτη-μέλη να έχουν τα λεγόμενα bank stop measures. Μπορεί να δημοσιεύουν κάποια αποτελέσματα που δείχνουν ότι ε, μία τράπεζα θα έχει πρόβλημα ρευστότητας ε, και η τράπεζα μπορεί να μην είναι σε θέση μετά να συλλέξει τα κεφάλαια τα οποία ζητούνται και κανένας δεν μπορεί να βοηθήσει την τράπεζα να συγκεντρώσει αυτά τα κεφάλαια. Οπότε τότε η τράπεζα αυτή, χωρίς να υπάρχει μια πραγματική κρίση, θα καταρρεύσει και θα την έχουμε προκαλέσει εμείς την κρίση αυτή. Αυτό φυσικά και δεν ε, πρέπει να το επιτρέψουν. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχουν αυτά τα μέτρα πριν από τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων ε, των δοκιμών αντοχής. Τι μπορούμε τώρα να αναμένουμε. Η τράπεζα ή εν λόγω μπορεί να συμφωνήσει με την αρμόδια αρχή, ε, την αρμόδια ελεγκτική αρχή, επί ενός σχεδίου ώστε οι ελλείψεις ε, οι οποίες ε, εντοπίστηκαν και επισημάθηκαν στα στρες τεστ να αντιμετωπιστούν. Βέβαια, μέχρι στιγμής δεν έχουμε συζητήσει ε, το θέμα αυτό. Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε μία εξάμηνη περίοδο, παραδείγματος χάρη, που θα μπορούσαμε να περιμένουμε τότε διορθωτικές κινήσεις. Και μετά τους έξι αυτούς μήνες, τέλος πάντων περί τα τέλη του έτους, θα πρέπει να δει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή τι ε, δράσεις ε, συμφωνήθηκαν και εφαρμόστηκαν. Και μετά θα σταθμίσουμε πολύ σοβαρά τι μέσα έχουμε εμείς στη διάθεσή μας, ώστε να ληφθούν οι απαραίτητες δράσεις αν δεν έχουν ληφθεί. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι αυτά τα μέσα που έχουμε, είπατε και εσείς, τη δυνατότητα να επιληφθεί και η Επιτροπή μας αλλά και το Κοινοβούλιο. Φυσικά και μπορούμε να εκδώσουμε συστάσεις και επίσης και άλλα μέτρα και μέσα έχουμε στη διάθεσή μας. Αλλά νομίζω ότι η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων και αξιολογήσεις θα ασκήσουν αρκετή πίεση στις τράπεζες που βλέπουμε ότι ήδη ε, συλλέγουν κεφάλαιο οι τράπεζες ε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ώστε όταν ε, δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα των stress test να έχουν ε, ήδη αν θέλετε κάνουν το καθήκον τους να έχουν ήδη κάνει το καθήκον τους σε σχέση με αυτό που χρειάζεται να γίνει για την έκδοση κεφαλαίου, νοπού κεφαλαίου. Είναι σημαντικό το θέμα και πρέπει να τονίσω ότι συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που είπε ο Μέρβιν. Δεν πρέπει να τα βλέπουμε μαύρα ή άσπρα. Ε, δεν πρόκειται περί μιας τέτοιου είδους απόφασης. Πηγαίνοντας και βλέποντας μια τράπεζα, κανείς μπορεί να αντιληφθεί ότι υπάρχουν ζητήματα ελλείψεις ε, σε κάποιες διαδικασίες μοντελοποίησης ή ε, εξέτασης και εξολόγησης της κινδύνου. Και μπορεί κάποιες τράπεζες να περάσουν, αν θέλετε, αυτή την εξέταση, αλλά παρόλα αυτά να χρειάζονται κάποιες ε, δράσεις που θα πρέπει να αναλυθούν για να διορθωθούν κάποια κενά και κάποιες αδυναμίες. Και υπάρχουν ίσως ενδεχομένως τράπεζες που δεν θα είναι πάνω από το κατόφλι, αλλά επειδή έχουμε θετήσει ε, πολύ αυστηρά ε, κριτήρια benchmarking, ίσως, ίσως κάποιες τράπεζες να έχουν ε, μια σημαντική ποσότητα αυτό που λέμε convertibles και να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Και μπορεί οι ελεγκτές να θεωρήσουν ότι μπορεί αυτό να αποτελέσει μια επαρκή απάντηση στις αδυναμίες που εντοπίστηκαν. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες και ποικίλε δράσεις. Δεν είναι μόνο η κεφαλαίου και ταχεία κεφαλαίου. Αλλά επαναλαμβάνω όλες τις δράσεις θα τις εξετάσουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Περνάμε τώρα ξανά στις ερωτήσεις προς τον Μέρβιν Κίνγκ. Πρώτος Σβέν Γκίνκολτ από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζουμε και εμείς. Ευχαριστούμε που ήρθατε και ελπίζουμε στο μέλλον να έχουμε τακτική ανταλλαγή απόψεων. Ε, έχω μία ερώτηση κλειδί. Δηλαδή, η, η Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου πώς περιλαμβάνεται στη δουλειά που παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ πιστεύω ότι πάρα πολλά ε, πάρα πολλές νομοθετικές διατάξεις ε, αφορούν μικροπροληπτικά θέματα. Βεβαίως ε, η Ευρωπαϊκή ε, Ρυθμιστική Επιτροπή ασκεί πίεση και μερικές φορές τα βρίσκουμε καλό, άλλες φορές πάλι όχι. Πάντως γνωρίζουμε ότι αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα. Τα μικροπροληπτικά θέματα περιλαμβάνονται πλήρως στο νομοθετικό έργο. Και αν πάρουμε το παράδειγμα του responsible lending, της υπεύθυνης δανειοδότησης, Ξέρουμε ότι αυτός είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες ε, που οδήγησε στο να προκύψει κρίση σε ορισμένα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Συστημικού Κινδύνου συμπεριλήφθηκε στο έργο της Κομισιόν, θα συμπεριληφθεί στο μέλλον. Και πώς μπορείτε να διασφαλίσετε να λαμβάνονται πλήρως ε, υπόψη οι δικές σας συστάσεις και πώς μπορούμε εμείς να σας βοηθήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Προφανώς λοιπόν η ε, ρυθμιστική αρχή δική μας υπάρχει μόνο εδώ και κάποιους μήνες και δεν έχουμε συμμετάσχει πολύ στο νομοθετικό έργο. Ε, θυμάστε, θα θυμάστε όμως ότι σας ανέφερα ένα παράδειγμα για το πού ακριβώς οι νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με την κεφαλαϊκή επάρκεια μπορούν να επηρεάσουν την δυνατότητα ε, της Επιτροπής μας να υποβάλει τις κατάλληλες μικροπροληπτικές προτάσεις. Αυτό το έχουμε κουβεντιάσει ε, και υπάρχουν ε, πρακτικά παραδείγματα που δείχνουν ότι εμείς ε, θέλουμε να είμαστε παρόντες στο νομοθετικό έργο για θέματα, για νομοθετήματα τα οποία επηρεάζουν τις αρμοδιότητές μας. Βεβαίως, το βασικό μας καθήκον είναι, όπως σας είπα, να εστιάσουμε ε, αποκλειστικά και μόνο στο μικροπροληπτικό στοιχείο. Αν όμως πιστεύουμε ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία της νομοθεσίας που μας δυσχεραίνουν το δικό μας το ρόλο, τότε να είστε σίγουροι ότι εμείς θα εκφράσουμε δυνατά την άποψή μας, είτε με συνεντεύξη τύπου, είτε σε συζητήσεις και γιατί όχι, και ε, στις ε, διάφορες ε, δικές σας εδώ επιτροπές, δηλαδή εφόσον ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συντημικού Κινδύνου υποτίθεται ότι θα έρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα εδώ στο Κοινοβούλιο. Πιο συγκεκριμένα θα υπάρχει συστηματική προσέγγιση για το πώς θα ερχόμαστε σε διαβουλέψεις μαζί σας. Μετά δηλαδή εδώ την παρουσία σας που είναι πάρα πολύ ευχάριστη και εκτιμώ πάρα πολύ ορισμένα που είπατε εδώ και έχετε πει και κατά παρελθόν. Νομίζω θα ήταν πολύ ενδιαφέρον για μας να ακούσουμε κατά πόσον θα έχετε κάποια συνάντηση με την Κομισιόν για να συζητήσετε το πώς σας θα διαβουλεύεστε ε, στο νομοθετικό έργο. Και στο μέλλον πώς εσείς βλέπετε αυτή τη συστηματική συνεργασία. Κοιτάξτε, ο ε, κύριος Όλι Ρεν ε, είναι στην Διευθύνουσα Επιτροπή και στο Διοικητικό Συμβούλιο της δικής μας Επιτροπής. Ε, άρα δηλαδή εκείνος μπορεί να αναφέρεται στην Επιτροπή και αυτό μέχρι τώρα λειτουργήσε ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Όμως εκείνος δεν είναι αρμόδιος για κανονισμούς χρηματοψηφιακών αγορών. Ναι, αλλά έχει στενές επαφές με εκείνους που είναι. Κοιτάξτε, δεν ανησυχώ ε, δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι ακριβώς κάνουμε. Εγώ πιστεύω ότι όταν η δική μας Επιτροπή έχει μια άποψη και θέλει να την εκφράσει, μην ανησυχείτε καθόλου, θα την εκφράσουμε ε, οπωσδήποτε. Ε, σήμερα το πρωί, μάλιστα, λέει η Πρόεδρος, ε, έλαβε χώρα μια συνέντευξη που ήταν παρόν ο Ανδρέας και δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι. Κοιτάξτε, ο κανονισμός που προέβλεψε την σύσταση της ε, Επιτροπής μας προβλέπει επίσης ότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα να καταθέτουμε συστάσεις για το νομοθετικό έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέχρι τώρα βέβαια δεν συζητήσαμε δεν έχουμε συζητήσει για την δυνατότητα να ε, συμμετέχουμε και εμείς σε κανονισμούς ή οδηγίες, ε, να, δεν ξέρω κατά πόσον είναι απαραίτητο να συμμετέχουμε με αυτή την αρμοδιότητά μας. Πάντως, μπορούμε να ελέγξουμε, να δούμε αν υπήρχαν προτάσεις που να έχουν σχέση με αυτό το θέμα. Πάντως, ε, η συζήτηση ε, είναι ενδιαφέρουσα. Είχαμε ήδη εμείς συζήτηση για τα αντικυκλικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν. Ε, μιλήσαμε για την εφαρμογή του πακέτου Βασιλεία 3 στην Ευρώπη, για το ρόλο των ρυθμιστικών αρχών, της δικής μας επιτροπής, ε, της συστημικής. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό όλοι άμεσα ενδιαφερόμενα να καταλήξουν σε μία άποψη. Και όπως ανέφερε και ο συνάδελφος, Υπάρχουν θέματα όπου η Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου ε, θεωρούμε ότι είναι αρμόδια. Υπάρχουν λοιπόν τα εργαλεία για να εκφράζουμε και εμείς την άποψή μας και να λαμβάνετε υπόψη προφανώς. Έχετε δίκιο ότι ε, πρέπει να υπάρχει ε, κάποιος οργανωμένος τρόπος να γίνονται όλα αυτά. Ακόμα δεν υπάρχει. Πάντως θεωρώ ότι πρόθεσμα θα πρέπει να μπορούμε και εμείς να εκφραζόμεθα ε, μικροπροληπτικά στην όλη διαδικασία νομοθετικού έργου. Ευχαριστώ και η Σουίνμπορν κατόπιν για τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ και τους ε, δύο που ήρθατε. Ο κύριος Ενρία το ανέφερε σε μία απάντηση στον Ζαν θα ήθελα εγώ να αναφερθώ σε με ένα πρόσφατο έγγραφο του ε, Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής ε, Σταθερότητας που είπε πως θα πρέπει να δούμε όλες τις δραστηριότητες εκτός του κανονικού ε, τραπεζικού συστήματος. Οπότε, δεδομένης ε, της Βασιλείας 3 που θα, αντιμετωπίσει, 3 που θα αντιμετωπίσει όλες αυτές τις προφανείς ελλείψεις, εσείς θεωρείτε πως θα υπάρχει ξημένος κίνδυνος ρυθμιστικού αρμπιτράζ και ειδικά εφόσον η εφαρμογή της ε, Βασιλείας 3 αυξάνει τον βαθμό της επίσημης τραπεζικής εποπτείας και ειδικά όσον αφορά αυτούς τους ομιχλώδεις ε, ενδιάμεσους ε, τους οποίους εσείς θεωρείτε πως θα πρέπει να είναι στην Επιτροπή σας. Μας τα είπε και ο Μάριο Ντράγκη σήμερα το πρωί αυτά, αλλά ε, Ανδρέα, νομίζω εσείς πρέπει να απαντήσετε. Ναι, ευχαριστώ. Νομίζω πως ο Ανδρέα είναι ο ειδικός. Ωραία λοιπόν. Κοιτάξτε αυτό το σκιώδες τραπεζικό σύστημα. Είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία απασχολούν την Επιτροπή μας και αυτή τη στιγμή με την Τεχνική Συμβουλευτική Επιτροπή που υποστηρίζει το έργο μας ε, οπωσδήποτε θα ξεκινήσουμε το τεχνικό μας έργο. Όπως είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση, το βασικό είναι να συλλέξουμε πληροφορίες για τον σκιώδη αυτόν τραπεζικό τομέα. Και όπως είπε και η πρόεδρος, το ανέφερε και ο Μάριο Ντράγκη σήμερα το πρωί πως βασικό τμήμα της δουλειάς μας είναι πως Κοιτάξτε, ο σχέδιος αυτός τραπεζικού τομέας είναι πολύ πίκυλος σε διάφορες ε, δικαιοδοσίες. Δεν είναι κάτι το οποίο λειτουργεί σε ένα ενοποιημένο πλαίσιο. Κοιτάξτε προσωπικά, ε, εγώ θέλω να γίνει δουλειά επ' αυτού και είναι νομίζω μια κοινή ευθύνη των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και της Επιτροπής μας. Για εμένα και το λέω και ενώπιον της Επιτροπής σας, ε, όταν μιλάμε για σκιώδες τραπεζικό σύστημα, ε, πρόκειται για μια αντίφαση ήδη στη διατύπωση, γιατί ε, οπωσδήποτε από πλευρά υποπτικών αρχών δεν μπορεί τίποτα το τραπεζικό να είναι σκιώδες και κρυφό και οπωσδήποτε από πλευρά κινδύνου εκτός ε, τραπεζικού στήματος, γιατί στο παρελθόν ε, ήμασταν πεπισμένοι πως ο μετασχηματισμός του κινδύνου και της ρευστότητα ήταν η βασική πηγή του κινδύνου, αλλά πλέον δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε ένα σύστημα το οποίο βλέπει μόνο ε, πως θα παρακολουθούμε μόνο τον τραπεζικό τομέα. Πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι που δημιουργούνται εκτός του τραπεζικού κλάδου. Και υπάρχουν μόνο δύο οδοί να ακολουθήσουμε πρώτη είναι οτιδήποτε δημιουργεί συστημικό κίνδυνο να μπει κάτω από την αιγίδα αυτή ή να περιορίσουμε αυτές τις δραστηριότητες που δημιουργούν συστημικό κίνδυνο σε φορείς ε, που είναι υπό αυστηρή εποπτεία. Αλλά το είπε και ο κύριος Ντράγκη σήμερα το πρωί πως είναι δύσκολη αυτή η υπόθεση, θα απαιτηθεί χρόνος γιατί δεν είναι τα πράγματα όπως το παρελθόν που έχουμε ε, λίγα ιδρύματα υψηλής μόχλευσης που δημιουργούν συστημικό κίνδυνο. Καμιά φορά υπάρχουν πολλά διαφορετικά ιδρύματα που συνδέονται και αναλαμβάνουν λειτουργίες που προσωμιάζουν με αυτές των τραπεζών και δημιουργούν συστημικό κίνδυνο. Και βεβαίως υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις σε κάθε δικαιοδοσία για το τι είναι ε, τραπεζικό σύστημα σε διάφορου ε, τομεί. Οπότε είναι δύσκολο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό η Επιτροπή μας να αναλάβει δράση για να συλλέξει εμπειρικά δεδομένα και να δούμε ποιε ε, είναι οι πιθανές πολιτικές μπορούν να ακολουθηθούν εδώ πέρα. Φαίνεται πως απάντησε τελικά ο καταλληλότερο, έστω και κατά λάθο. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση για τον Ανδρέα θεωρητικά προέρχεται από τον Φιλίπ Λάμπερτ από του πράσινου. Είστε έτοιμος. Α, Πασκάλ. Ναι, αλλάξαμε τη σειρά, αν δεν σας πειράζει. Ήθελα να είμαι ο Ήθελα να κάνω ε, δύο πολύ σύντομα ερωτήματα. Το πρώτο αφορά το κείμενο για τα παράγωγα προϊόντα με συγκεκριτή τον Βέρνερ Λάγκεν. Θα τοποθετηθείτε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου για τον τρόπο με τον οποίο το κείμενο και συγκεκριμένα διάταξη για την ανάλυση συστημικών κινδύνων στη δημιουργία κάποιων του ε, συμψηφισμού πρέπει ε, να γίνει κάπως ε, δημόσια για να εκφραστούν οι προσδοκίες που υπάρχουν και οι μελλοντικέ αυτές τις να μην ανταγωνίζεται η μία την άλλη για κάποια σημεία κλειδιά που αφορούν βέβαια το risk management όπως είναι η ποιότητα των εγγύσεων ή τα ποσά που θα απαιτούνται. Θα παρέμβετε συγκεκριμένα πάνω σε αυτό. Και δεύτερο ερώτημα, παγκόσμια μόχλευση της οικονομίας. Έχω την εντύπωση ότι μιλάτε σαν ήδη να έχει μειωθεί το επίπεδο μόχλευσης. Έχουμε μεν το δημόσιο χρέο, έχουμε και το ιδιωτικό όμω χρέο. Αν δούμε παραδείγματο χάρη την περίπτωση τη Γαλλίας, το επίπεδο ιδιωτικού χρέους συνεχίζει να αυξάνεται. Άρα δεν θέλουμε απλά να προλάβουμε κάποια μελλοντική κρίση, αλλά πρέπει να ρυθμίσουμε και σήμερα αυτό το πολύ υψηλό ιστορικά επίπεδο ιδιωτικής χρέωση ιδιωτικού χρέου. Ποια είναι τα εργαλεία και ε, μέτρα τα οποία εσεί. Ε, προτείνεται ώστε να μειωθεί, αλλά όχι με χαοτικό τρόπο, πολύ γρήγορα πάντως το ιδιωτικό χρέος. Ευχαριστώ. you want to ε? Ναι, για το πρώτο σας ερώτημα για τα παράγωγα και κατάλαβα καλά για το νομοθετικό κίνημα, ε, κείμενο μας για τους ε, μηχανισμούς αυτούς αντιστάθμισης. Υπάρχουν ε, και πάρα πολλές δουλειές για τα over the counter και τα νομοθετικά κίνητρα για να υπάρχουν κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι όπου θα γίνει η ακαθάριση Οπότε υπάρχουν νομοθετικές ε, πρωτοβουλίες που έχουν επίδραση στο συστημικό κίνδυνο και μπορεί κάλλιστα η Επιτροπή μας ε, να τοποθετηθεί και να συζητήσει. Όπως είπα έχουμε αυτές τις συζητήσεις. Όταν αυτό απαιτείται. Και θα ήθελα να τονίσω πως προσωπικά δεν θεωρώ πως η βασική δουλειά μας είναι να εξετάζουμε την ομοθεσία, αλλά σημαντικό είναι να έχουμε ένα μηχανισμό που θα διασφαλίζει πως όταν ε, συντάσσεται η νομοθεσία που θα επηρεάζει τον συστημικό κίνδυνο, τότε η Επιτροπή μας να έχει την ευκαιρία να την συζητήσει και να δούμε αν υπάρχει ανάγκη κάποιας συνεισφοράς. Συνολικά λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν βλέπω σοβαρή ανάγκη για την Επιτροπή μας να παρέμβει. Αλλά οπωσδήποτε θα υπάρξει κάποια στιγμή ε, στην οποία θα, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε το θέμα. Δεν ξέρω αν απαντάει αυτό στην ερώτησή σας. Επίσης το ζήτημα για τα όρια των εγγύσεων. Είναι σαφές πως όλοι αυτοί οι μηχανισμοί έχουν αντίκτυπο στο συστημικό κίνδυνο και είναι άρα σημαντικό όλες αυτές οι πρωτοβουλίες να λαμβάνονται με βάση στιβαρά εμπειρικά δεδομένα και τα δεδομένα τα εμπειρικά τα οποία συλλέγει η Επιτροπή μας για τον συστημικό κίνδυνο λαμβάνονται υπόψη όταν γίνονται αυτές οι πρωτοβουλίες. Οπότε όσον αφορά π.χ. την διαχείριση εγγυήσεων σε κεντρικούς ε, αντισυμβαλωμένους κτλ. Όλες οι πληροφορίες ε, που μπορεί να έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή μας ε, να χρησιμοποιούνται εάν μπορούν να συνεισφέρουν στη συζήτηση περί νομοθετικών πρωτοβουλειών. Ευχαριστώ. Νομίζω Μέρβιν και εσείς θέλετε να τοποθετηθείτε. Ναι, θα απαντήσω στην ερώτηση για τη μόχλευση, αν μου επιτρέπετε. Ε, αυτό προφανώς είναι μεγάλη πρόκληση για τον χρηματοοικονομικό τομέα. Υπήρχε μείωση της μόχλευσης. Για το δημόσιο χρέας υπήρχε σαφώς αύξηση της ε, μόχλευσης. Και τα δύο αυτά δεν είναι τελείως ασύνδετα. Και όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, αν μιλάμε για επιχειρήσεις ή για νοικοκυριά και αναλόγως τη χώρα, είτε έχει αυξηθεί, είτε έχει μειωθεί, είτε έχει παραμείνει η ίδια η μόχλευση. Συνολικά, από όταν ξεκίνησε η κρίση, το πρόβλημα της μόχλευσης και ο συνολικός όγκος χρέους στην οικονομία είναι πάρα πολύ μεγάλος και αυτό βεβαίω αποτελεί μεγάλη μακροοικονομική πρόκληση. Είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο τα επιτόκια είναι τόσο χαμηλά και γιατί οι κεντρικές τράπεζες αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις στο να ορίσουν την νομισματική πολιτική. Οι μακροοικονομικές αυτές προκλήσεις θα κρατήσουν χρόνια και θέτουν περαιτέρω συστημικούς κινδύνους υπό την έννοια πως ε, εάν ε, το κλίμα αυτό αλλάξει των πολύ χαμηλών πραγματικών ε, επιτοκίων τότε θα γίνουν σοβαρότερες οι επιπτώσεις του υψηλού επίπεδου Χρέου αυτή τη στιγμή και δεν το υποτιμώ αυτό καθόλου και δεν θεωρώ πως η υποτροπή μας έχει μέσα στην διάθεσή της για να μειώσει το επίπεδο μόχλευσης καθ' αυτό. Αλλά μπορεί να απευθύνει προειδοποιήσεις, να επιστήσει την προσοχή στα προβλήματα που προκύπτουν από αυτό το πολύ ψηλό επίπεδο μόχλευσης. Αν και για να είμαι ειλικρινής φαντάζομαι πως αυτά τα γνωρίζουν όλοι όσοι λαμβάνουν τι αποφάσει σαν την Ιφίλιο, γιατί έχουν βεβαίω τα τελευταία τέσσερα χρόνια κυριαρχήσει στι ε, ζωέ μα, Οπότε είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και είναι μέρος του λόγου για το ότι ακόμα η κρίση η οποία ξεκίνησε έχει πολλά χρόνια μπροστά της και οι συνέπειές της θα είναι αισθητέ για πολλά χρόνια στο μέλλον. Ευχαριστώ. Επανερχόμαστε σε εσά. Κέι για μια ερώτηση που θα απαντήσει, από ό,τι γράφει εδώ πέρα, ο Μέρβιν Κίνγκ. Είμαι σίγουρο πως και οι δύο είναι ικανοί να απαντήσουν. Το θέμα είναι ποιος θέλει. Καθώς προχωράμε στο νομοθετικό πρόγραμμα για την σύσταση κονδυλίων διάλυσης τραπεζών, θα ήθελα αν θέλετε να σχολιάσετε από πλευράς συστημικού κινδύνου για το εάν θα προτιμούσατε 27 ε, εθνικά ταμεία εξ αντε ή ένα ευρωπαϊκό τέτοιο ταμείο και τι, τέτοιο, τι κίνδυνο θα έχει η προχρηματοδότηση ε, ειδικά όσον αφορά τον ηθικό κίνδυνο και σε σχέση με την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Θα είμαι ε, σαφώς, σαφής όσον αφορά το θέμα αυτό, γιατί είμαι ξεκάθαρο όσον αφορά το καθεστώς resolution το, το θέμα της διάλυσης εξυγείανης τραπεζών. Κοιτάξτε, ε, είναι πολύ σημαντικό ε, να υπάρχει ενιαία λειτουργία και εδώ υπάρχει ε, ένα σαφές εμπόδιο. Πιστεύω ότι στις περισσότερες εποπτικές αρχές οι αρχές εξυγίανσης δεν, είναι, δεν γνωρίζουν τι ακριβώς επιδιώκουν. Ε, υπάρχει η εναλλακτική λύση του δικαίου χρεοκοπίας ε, όλοι οι πιστωτές ε, θα μπορούσαν ίσως να κηρύξουν χρεοκοπία αλλά αυτό θα δημιουργούσε πρόβλημα στις καταθέσεις. Εκείνο λοιπόν που έχει σημασία είναι αυτό το καθεστώς της διάλυσης, της εξυγίανσης, ε, αυτό το καθεστώς σε διεθνές επίπεδο λίγο πολύ να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Πάντως, εγώ δεν συμφωνώ να υπάρχουν αυτά τα ε, κονδύλια εξυγίανσης, είτε είναι εθνικά, είτε για μεμονωμένες περιπτώσεις. Και η απάντηση είναι απλή, ότι εγώ ανησυχώ, ε, γιατί αν υπάρχουν τέτοιου είδους κονδύλια, ε, εκεί οι τράπεζες μπορούν να πούν αυτά είναι δικά μας χρήματα, αυτά είναι για να σωθούμε εμείς αν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Τώρα, κατά πόσον θα είναι εθνικά κονδύλια ή ευρωπαϊκά κονδύλια, κοιτάξτε, τέτοιου είδου κρίση τα τελευταία 35 χρόνια δεν υπήρξε. Μετά από 35 χρόνια ε, δεν γνωρίζει κανείς σε ποιον ακριβώς ανοίγουν τα, ανήκουν τα κονδύλια. Και η πίεση για τη διάσωση των τραπεζών θα είναι τεράστια. Αυτό που έχει σημασία είναι να είμαστε προσεκτικοί, γιατί αν υπάρχει ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί στην Ευρώπη και σε διεθνές επίπεδο, είναι το πρόβλημα των τραπεζών που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κατάρρευσης δεν μπορούν να εκτεθούν τόσο πολύ οι τράπεζες γιατί αν κάτι δεν πάει καλά τότε εσείς και εγώ και όλοι μας θα πρέπει να τις διασώσουμε όπως ακριβώς συνέβη. Αυτό λοιπόν ε, που πρέπει να κάνουμε είναι να εισάγουμε σαφή καθεστώτα εξυγίανσης όπου θα είναι ξεκάθαρο ότι ε, στις απώλειες, στις ζημιές θα συμμετέχουν και επενδυτές και όχι μόνο οι απλοί φορολογούμενοι. Και αυτό να το γνωρίζουν και οι απλοί καταθέτες. Ευχαριστώ. Έχουμε κάπως τηρή στο χρονοδιάγραμμα. Hans Peter Martin ο τελευταίος, ο μιλητής Werner Langen. And Gay Mitchell. Uh, there won't be another. That will... Τέσσερις συνολικά. Ο Hans Peter Martin ο πρώτος. I will go to Hans Peter Martin next. Ja, danke, das passt gerade ganz gut. Uh, Ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κίνγκ το εξή. Επειδή αναφέρθηκε στο, στις τράπεζες και είπε ότι είναι πολύ μεγάλες για να καταρρεύσουν. Too big to fail. Και ρωτώ, εσείς λαμβάνετε υπόψη σας ε, τα εθνικά στοιχεία, ε, τη σχέση ΑΕΠ και προϋπολογισμού. Και στη δική μου τη χώρα στην Αυστρία, στην Ισλανδία, στο Βέλγιο, δεν ξέρω, διερωτώ με κατά πόσον έχουν έτσι μια εικόνα για το ποιο είναι το οριακό σημείο οι οριακές τιμές. Μετά, βάσει της ε, Συμφωνίας Βασιλεία 3, εκεί αναφέρεται ότι ε, εάν υπάρχουν αυστηρότερα κριτήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κανονισμοί, αυτό ε, δημιουργεί μειονεκτική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις ΗΠΑ. Εσείς πώς ακριβώς τοποθετήσετε επ' αυτού. Όσον... Νομίζω ότι όσον αφορά το πρώτο θέμα πρέπει νομίζω να αναγνωρίσουμε ότι σχεδόν κάθε τράπεζα μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλη για να αποτύχει, για να καταρρεύσει υπό τις σωστές συνθήκες γιατί μπορεί να ε, υπάρξει επέκταση του προβλήματος και όταν θεωρούμε ότι υπάρχει μια ανάγκη διάσωσης ε, για κάποια τράπεζα πρέπει να το κάνουμε γιατί τέλος θα υπάρξει επιμόλυνση, μετάδοση του, του προβλήματος. Όλες οι χώρες ε, έχουν υποφέρει στο πλαίσιο αυτής της χρηματοπιστωτικής κρίσης και από αυτό το πρόγραμμα της μεγάλης, πολύ μεγάλης τράπεζας. Υπάρχει εθνική και διεθνής ε, διάσταση. Νομίζω ότι το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προσπαθεί σκληρά να βρει λύση ε, σε ένα διεθνές, ε, για ένα διεθνές καθεστώς εξυγίανσης. Αλλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει μόνο ένα και νομικά έτσι, σταθερό και δεσμευτικό καθεστώς. Θα πρέπει να βασιστούμε και στους εθνικούς ε, ελεγκτές εποπτικές αρχές που θα πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν θα πρέπει οι διεθνείς τράπεζες να γίνουν τόσο πολύ μεγάλες που να θεωρήσουν ότι είναι μεγαλύτερες και πιο σημαντικές από τις ελεγκτικές αρχές και τα ίδια τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν και αυτές οι τιμές κατοφλίου. Νομίζω ότι θα πρέπει το καθεστώς που θα προτείνουμε να ισχύει για όλες τις τράπεζες. Και θα πρέπει οι τράπεζες να μπορούν με να καταρρεύσουν αλλά με τρόπους που δεν θα ε, υπονομεύουν τη σταθερότητα του συστήματος συνολικά. Και όταν έχουμε να κάνουμε με διεθνείς συμφωνίες, είναι πάρα πολύ σημαντικό στην Ευρώπη εμεί να μιλούμε με του Αμερικανού συναδέλφου και όσο το δυνατόν να προσπαθούμε να καταλήγουμε σε συμφωνίε. Και σε ό,τι αφορά τι κεφαλαϊκέ απαιτήσει, που αντιμετωπίζουν οι πάρα πολύ μεγάλες αυτές ε, τράπεζες, τα σημαντικά δηλαδή από συστημική άποψη χρηματοπιστωτικά δρήματα, τα σύφης όπως τα αποκαλούν. Και σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρώπη να μιλάμε μία φωνή. Αυτό θα κάνει πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Αυτό που πρέπει να αναγνωρίσουμε πάντως ε, σε τελική ανάλυση είναι ότι οι χώρες οι οποίες θέλουν να στηρίξουν ε, μεγάλα τραπεζικά συστήματα σε με το ε, δεν θα πρέπει να ε, παρεκτραπούν. Είδαμε πάρα πολύ ξεκάθαρα τι έγινε με την Ισλανδία και την Ιρλανδία, δύο χώρες που ανεξαρτήτως του τι έλεγαν οι διεθνείς συμφωνίες, ε, δεν ήταν καθόλου λογικό αυτό που έκαναν, να επιτρέψουν ε, σε σχέση με το ΑΕΠ τα τραπεζικά του συστήματα να διοκωθούν τόσο πολύ. Γιατί έτσι σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν να διασωθούν με χρήματα των φορολογουμένων αυτά τα τραπεζικά συστήματα και είδαμε τι έγινε στην Ιρλανδία και στην Ισλανδία, επαναλαμβάνω. Πρέπει λοιπόν να το αποφύγουμε αυτό το πρόβλημα και αυτό είναι και ένα λόγο για τον οποίο κάποιε χώρε ίσω θεωρούν ότι ακόμη ε, και σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να προσπαθήσουν να λύσουν ε, το θέμα αυτό των ε, πολύ μεγάλων για να καταρρεύσουν τραπεζών. Εάν δεν τα καταφέρουμε πάντως με αυτό το θέμα, η επόμενη κρίση όποτε και αν είναι σε 10, 20, 30 χρόνια τότε θα μας κατηγορήσει ο κόσμος και θα πει το ήξεραν 10, 20, 30 χρόνια πριν, το είχαν αντιμετωπίσει, δεν βρήκαν τρόπο και αυτό θα είναι ένα κληροδότημα, μια κληρονομιά φρικτή για να δώσουν σε επόμενες γενιές. Δεν θα πρέπει να μας ε, απογοητεύει ούτε να μας ε, αποθαρρύνει το λόμπινγκ που μπορεί να ασκηθεί. Θα πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα με τις ε, too big to fail τράπεζες. Βέρνερ, Βέρνερ Λάγκεν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άκουσα πώς απαντήθηκαν οι ερωτήσεις της κυρίας Γκουγιάρ και του κυρίου Καμφά ε, καθώς δήλωσε ο κύριος ε, Ενερία έτοιμος να τοποθετηθεί πιθανώς και στην νομοθετική διαδικασία. Η τελευταία παρατήρηση του κυρίου Κίνγκ ε, μου λέει πως μέχρι στιγμής δεν έχουμε έναν μηχανισμό που να εμποδίζει π.χ. το ότι να φτάσουν οι Ισλανδικές τράπεζες το 350% του ΑΕΠ και οι Ιρλανδικές το 250% του ΑΕΠ και βεβαίως δεν φαίνεται πως λόγω των συγχωνεύσεων δεν έχουμε μικρότερες τράπεζες αλλά μεγαλύτερες. Αν σκεφτείτε την Societe Generale που αγόρασε την Fortis και την KPC και την Commerzbank που αγόρασε την Dresdner. Ε, τέλος πάντων, μπορούμε να τα δούμε αυτά τα κριτήρια. Αλλά το ερώτημά μου είναι άλλο. Το ερώτημα είναι τι γίνεται με τα τεστ κοπόσεως αυτά, πώς θα διαμορφωθούν. Στη Βασιλεία 2 Έχουμε κάποιες χώρες που δεν την έχουν εφαρμόσει ακόμα. Για τις ε, κεφαλαιακές απαιτήσει υπάρχουν ε, δεκαετής ε, μεταβατικές ρήτρες. Και το ερώτημα λοιπόν είναι προς τον κύριο Νρία. Τώρα κάνετε εσείς αυτά τα τεστ κοπόσεως και είπατε πως θα έχουμε στο επόμενο εξάμεινο τα αποτελέσματα και ήδη για τα ίδια κεφάλαια χρησιμοποιείτε ήδη τη Βασιλεία 3 ως κριτήριο χωρίς να λάβετε υπόψη την δεκαετή προθεσμία που υπάρχει για την εφαρμογή. Πώς θα οδηγηθούμε ε, χωρίς ε, να ισχύει η σωστή νομική βάση σε μία, σε μία στρέβλωση της αγοράς. Ένα λεπτό ε, λέει η κυρία Πρόεδρος είναι η κάθε ερώτηση. Και επιμένω γιατί η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή αγνόησε και άλλαξε τις απαιτήσει περί ιδίων κεφαλαίων που ισχύουν, τις οποίες συναποφάσισε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εις βάρος κάποιων τραπεζικών ομίλων. Ε, νομίζω πως αυτή ήταν η επιπλέον ερώτηση του ΕΛΚ. Ανδρέα. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ για την ερώτησή σας, γιατί μου επιτρέπει να ξεκαθαρίσω ποια ήταν αυτή η απόφαση που έλαβε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική ε, αρχή. Κοιτάξτε, έχουμε ένα νομοθετικό ορισμό του, του κεφαλαίου που βασίζεται στο Tier 1 και ε, αυτός ο ορισμός ε, έχει ακυρωθεί γιατί πλέον οι αγορές, ε, τα αυξημένα αυτά μέσα δεν τα θεωρούν επαρκή εξασφάλιση από τις απολύσεις και μάλιστα οι υποπτικές αρχές ε, στην ε, συμφωνία των G20 Σεούλ το Νοέμβριο που πέρασε είπαν πως θα πρέπει να πάμε προς ε, κάποιες ρυθμίσεις που θα δουν όσον αφορά τον ορισμό του κεφαλαίου πολύ αυστηρότερα. Ταυτόχρονα είπατε βεβαίως πως οι G20 αποφάσισαν με βάση την πρόταση της Επιτροπής της Βασιλείας και των Ρυθμιστικών Αρχών να έχουν μια αρκετά μεγάλη μεταβατική περίοδο όσον αφορά τις ε, κεφαλαϊκές απαιτήσεις για να μην εμποδίσουμε την ισχνή ακόμα ανάκαμψη και βεβαίως δεν είναι πρόθεση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής να αντιταχθεί σε αυτήν την απόφαση. Γι' αυτό δεν ε, εφαρμόσαμε ε, τον ε, ορισμό της ε, Βασιλείας 3 για τις κοινέ μετοχές για αυτό το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε λοιπόν είναι να εξειδικεύσουμε τον ορισμό που υπάρχει στην νομοθεσία και να φτάσουμε στον αυστηρότερο ορισμό που εξπονοείται αν θέλετε στο crb που ισχύει ήδη από πρώτης πρώτου. Ε, συμφωνήσαμε ήδη πως ε, το μέτρο σύγκριση θα είναι πάρα πολύ κοντά στον ορισμό κεφαλαίου που θα τεθεί εν ισχύ ε, από 1η Πρώτου 2013 όταν το νέο πλαίσιο θα αρχίσει να ισχύει οπότε έχουμε τις μεταβατικές αυτές διατάξεις βεβαίως που ισχύουν και καθώς η περίοδος που καλύπτεται από τα τεστ όπως είναι μέχρι 31 Δεκάτου 2012, λογικό είναι οι τράπεζες να έχουν ε, το επαρκές κεφάλαιο, το οποίο θα ισχύει την ε, επόμενη μέρα από την ολοκλήρωση των τεστ. Δεν είναι λοιπόν ε, οι, τελευ... οι οριστικές αυτές απαιτήσει της Βασιλείας 3, που θα ισχύσουν μόλις το 2018 και θα είναι πολύ σκληρότερες από αυτά τα οποία εφαρμόζουμε είναι ε, κάτι άλλο το πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ε, αυτό το οποίο είναι το ότι εφαρμόζουμε αυτά τα οποία ισχύουν στη ΣΥΠΑ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την αξιοπιστία των ε, αποτελεσμάτων παγκοσμίω. Πρέπει να γνωρίζετε πως οι τράπεζες μας σε κάποιες χώρες αντιμετωπίσουν προβλήματα όσον αφορά το δημόσιο χρέος και εκεί πέρα έχουν προβλήματα στη χρηματοδότηση, στις ε, χρηματαγορές και πολύ μεγάλο μέρος αυτής της χρηματοδότησης προέρχεται από διεθνείς επενδυτές, από τη ΣΥΠΑ, οπότε πρέπει να έχουμε αξιόπιστα αποτελέσματα τα οποία θα είναι αποδεκτά και κατανοητά και από τους διεθνείς επενδυτές. Οπότε νομίζω πως κάναμε τη σωστή επιλογή και δεν είναι πλήρης ε, δεν είναι ε, η πλήρης εφαρμογή της Βασιλείας 3 του 2018 αυτή που εφαρμοστούμε. Ευχαριστώ για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο κ. Χουανγκό. Ευχαριστώ πολύ. Το ερώτημά μου είναι προς τον κύριο Κίνγκ, ο κύριος Κόνγκ. Πολλοί τραπεζίτες θεωρούν ότι υπάρχει ένα συστημικός κίνδυνος που συνδέεται με το δημόσιο χρέος. Σε ό,τι αφορά τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο, το δημόσιο χρέος είναι συγκρίσιμο με το χρέος πολλών χωρών της ζώνης του ευρώ. Και μετά από πληροφορίες γνωρίζουμε ότι η Τράπεζα της Αγγλίας παρενέβη και αγόρασε ε, κάποια ε, κρατικά ε, ομόλογα Μπορείτε να μας πείτε το ποσό και θεωρείτε ότι αυτό συνέβαλε στο να μετριαστούν οι κίνδυνοι να έχουμε κρίση δημόσιου χρέους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και βέβαια ως αντιπρόεδρος της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συστημικού Κινδύνου τι διδάγματα αντλείτε εσεί και τι θεωρείτε ότι θα πρέπει να διδαχθεί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ώστε να παρέμβει σε περίπτωση που προκύψει συστημικό κίνδυνο σε σχέση με κάποια δημόσια χρέη χωρών της Ευρωζώνης. Παραλαμβάνω. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, αγοράσαμε 200 εκατομμύρια λίρες ε, σε ομόλογα. Κάτι το οποίο βεβαίω στόχο είχε να αυξήσει την ποσότητα χρήματος στην οικονομία για να μην υπάρξει συρρήκνωση της ποσότητας χρήματος και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και εμείς θεωρήσαμε την αύξηση της ε, ποσότητας χρήματο ω σημαντικό μέρος ε, της ανάπτυξη και χωρί αυτό βεβαίω θα είχαμε ε, σφιχτή νομισματική πολιτική χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Επίσης δεν θεωρώ πως το κατά πόσο εμείς ανησυχούσαμε είχε κάποια διαφορά όσον αφορά τον κίνδυνο του δημοσίου χρέους του Ηνωμένου Βασίλειου. Αυτό επηρεάστηκε από τις δράσεις των κυβερνήσεων πριν και μετά τις εκλογές που ε, βεβαίως έπρεπε να καταθέσουν ένα ρεαλιστικό σχέδιο για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της ε, οικονομικής κρίσης και αυτό ήταν το οποίο επηρέασε οι δράσεις των κυβερνήσεων και όχι οι δράσεις των κεντρικών τραπεζών. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στον Βολφ Κλίντς που επίσης θα απευθυνθεί στον Μπέρλιν Κίνγκ. Σας ευχαριστώ. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας ε, έχει αποκτήσει μια παγκοσμιοποιημένη διάσταση και αν εξετάσουμε το συστημικό κίνδυνο από την ευρωπαϊκή προοπτική, τότε ε, αποκτάμε μόνο ένα κομμάτι των απαντήσεων που αναζητάμε. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο και διαχειριστικά ε, όλα τα συμπεράσματά σας να τα συνδυάσετε με αυτά των συνεργατών σας, κυρίως αυτών από τις ΗΠΑ. Και θέλω να ρωτήσω, υπάρχει ένα είδος ε, άτυπης ή έστω επίσημης ε, συνεργασίας μεταξύ σας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά, ε, κάποιες συζητήσεις που κάνετε ή συμπεράσματα που εξάγετε, αυτά τα κοινοποιείτε στο κοινό γιατί αν δεν το κάνετε ή πριν το κάνετε ενδέχεται να υπάρξουν καταστρεπτικές συνέπειες στην αγορά. Εσείς πώς ελέγχετε αυτόν τον κίνδυνο. Να πω το εξής. Καταρχήν δείτε κάτι πολύ σημαντικό ότι ο χρηματοψηφιακός τομέας είναι πλέον παγκοσμιοποιημένος και νομίζω τα αίτια τα υπολαμβάνοντα αίτια της κρίσης ε, προφανώς είναι και αυτά παγκοσμιοποιημένα. Δηλαδή από το κεφάλαιο, από χώρες αποταμίευσης, ε, εισέρευσε σε χώρες με, ε, από μεγάλη αποταμίευση σε χώρες με χαμηλή αποταμίευση. Έχετε λοιπόν δίκιο ότι στην τράπεζά μας, στην επιτροπή μας, εμείς δεν μπορούμε να προσφύγουμε ότι αγνοούμε τον υπόλοιπο κόσμο και υπάρχει μια κουρτίνα που μας χωρίζει εδώ στην Ευρώπη. Στην αρχική μου παρέμβαση ανέφερα κάποιους κινδύνους και ένας εξ αυτών είναι πόσο θα ισχύσουν τα μακροπρόθεσμα χαμηλά επιτόκια και κατά πόσο ενδέχεται να αυξηθούν λόγω παρεμβάσεων στην Ασία ε, από πάντως εκτός Ευρώπης και πώς ε, θα αποδειχτεί, πόσο θα πειράσουν το χρηματοψηφιακό ε, σύστημα. Εγώ δεν νομίζω ότι έχει νόημα να δημιουργήσουμε άλλον ένα μηχανισμό επίσημο, γιατί έχουμε αρκετές επιτροπές που συστήθηκαν μετά από αυτή την κρίση. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι οι εμπλεκόμενοι να μιλάνε ανοιχτά, έστω και κατηδίαν, πάντως να είναι ειλικρινείς μεταξύ τους και να θέλουν να λάβουν δράση. Τόσο ο κύριος Ζαν Κλώτρισε, όσο και εγώ, συναντιόμαστε συχνά με τους ε, ε, ομολόγους μας ε, στο πλαίσιο της G20 και στη Βασιλεία και στους ε, κόλπους στη G7 και στους, ε, στις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές ευκαιρίες και οι αναπληρωτές μας συναντιόνται στο ε, Συμβούλιο Χρηματοψηφικής Σταθερότητας. Πάντως, εκείνο που παίζει ρόλο είναι να έχει κανείς ε, κατά νου ε, τους κινδύνους που υφίστανται και δράση μπορούμε να λάβουμε μόνο εφόσον γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Ευρώπη είναι μια ψηφίδα ενός ευρύτερου μοσαϊκού. Κατά τα άλλα, αναφερθήκατε στην δυνατότητα οι δικές μας οι διαβουλεύσεις να δημοσιοποιούνται πριν εμείς το αποφασίσουμε. Κοιτάξτε, η, η άποψή μου είναι ότι οι ε, κεντρικοί τραπεζίτες δεν αφήνουν να, διαρρεύσει, να διαρρεύσουν πράγματα ούτε στη Βασιλεία ούτε και αλλού που συναντιόμαστε. Δεν το κάνουν αυτό οι ε, κεντρικοί τραπεζίτες. Είναι αλήθεια ότι μερικές φορές οι πολιτικοί το κάνουν αυτό, αλλά πολύ σπάνια οι κεντρικοί τραπεζίτες. Γι' αυτό λοιπόν ε, όταν συναντιόμαστε θεωρώ ότι οι συνάδελφοί μου τα απόρριτα θέματα τα φυλάτουν απόρριτα. Τουλάχιστον ε, μέχρι σήμερα έτσι έχουν τα πράγματα. Υπάρχει ε, βέβαια και το θέμα ε, των εμπιστευτικών, της εμπιστευτικής ενημέρωσης στο Προεδρείο αυτής της ε, Επιτροπής και όσων ε, είναι παρόντες. Αυτό ίσως πρέπει να το έχουμε κατά νου όσον αφορά τις ε, ερωταπαντήσεις. Ερώτηση από τον Γκέι Μίτσελ. Θεωρητικά είναι για τον κύριο Αντρέα Ρία, αλλά θα δούμε σε ποιον κατ' ουσίαν απευθύνεται η ερώτηση. θα ήθελα να ρωτήσω τον πρόεδρο Ανρία το εξής. Η αρχή συστημικού κινδύνου μπορεί να δράσει. Μήπως υπάρχουν πάρα πολλοί ε, και τελικά μπερδεύονται πάρα πολύ. Και κύριε Κίνγκ, θα ήθελα να σα ρωτήσω το εξή. Άκουσα αυτό που είπατε ότι οι τράπεζε δεν μπορούν να διασωθούν από τον Ιρλανδό ε, φορολογούμενο. Έχει αυξηθεί στο 120% ε, το χρέος μας από την άλλη, ξέρετε ότι δεν έχουμε έσοδα από την ιδιοκτησία, γι' αυτό το έλλειμμα του προπολογισμού είναι πολύ ψηλό. Εμείς όμως αναλάβαμε να το αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Υπάρχει και ένα άλλο, η ε, κεφαλαϊκή επάρκεια των τραπεζών και εμπιστοσύνη στις τράπεζες. Πολλοί αφαίρεσαν, πήραν τις καταθέσεις τους και μερικοί είπαν ότι αν είχαν εμπιστοσύνη θα επανέφεραν τις καταθέσεις τους. Η ερώτηση είναι η εξής. Νομίζω 130 δις ε, είναι το ποσό ε, της ε, Κεντρικής Τράπεζας που θα διατεθεί για μας και κατά την άποψη αν διατεθεί αυτό ε, θα δημιουργούσε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη εάν ένα κομμάτι αυτού του ποσού ήταν βραχυπρόθεσμα, δηλαδή από 6 μέχρι 12 μήνες, έτσι ώστε να έβλεπαν οι Ιρλανδοί φορολογούμενοι ότι δεν καλούνται να κάνουν τα πάντα και μόνο μιας και ότι υπάρχει μια διάτεξη όχι βραχυπρόθεσμη αλλά και μακροπρόθεσμη. Ανδρέα. Ίσως μπορείτε να απαντήσετε στο πρώτο κομμάτι της ερώτησης. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Ε, μάλλον, υπάρχουν πάρα πολλοί πράγματι που εμπλέκονται στην ε, Ρυθμιστική Επιτροπή, αλλά και αυτό είναι και το ατού μας, το ότι ε, συμμετέχουν όλοι όσοι ασχολούνται με τα μικροπροληπτικά. Εμείς ε, τώρα αυτό που είπατε το κατά πόσο θα πρέπει να αποφύγαμε να είμαστε μια λέσκη συζητήσεων. Κοιτάξτε, νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί με το να εντοπίζουμε κινδύνους ε, και να λαμβάνουμε μέτρα ή να λέμε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα. Στους ε, πρώτους μήνες της ζωής μας ακολουθούμε αυτή την κατεύθυνση. Η Διευθύνουσα Επιτροπή είναι ένα σημαντικό όργανο το οποίο προσφέρει την, ε, την κατεύθυνση, το, τη στρατηγική, τις συζητήσεις ε, για ε, θέματα σε μικρότερες ομάδες και κατόπιν αυτό που έχει σημασία είναι και οι τεχνικές ομάδες να λειτουργούν και αυτές έτσι ώστε και αυτές να μπορούν να προσφέρουν στην ε, Ρυθμιστική Επιτροπή, στην Επιτροπή ε, Ρυθμιστικού Κινδύνου. Σημασία έχει επίσης να έρχονται και παρεμβάσεις και προτάσεις από άλλες επιτροπές προς την κατεύθυνση της ανάληψης ενεργειών. Θεωρώ λοιπόν ότι ένα από τα σημαντικότερα ελλείμματα που είχαμε κατά τη διάρκεια της κρίσης και μετά ήταν ότι δεν υπάρχει και δεν υπήρχε ένας χώρος όπου να λάβει η χώρα ειλικρινή συζήτηση, απόρριτη, εμπιστευτική, ανάμεσα σε όλους όσοι εμπλέκονται σε θέματα κρηματοψηφιακής σταθερότητας. Τώρα όμως υπάρχει αυτή η δυνατότητα και είναι πολύ καλό που εμπλέκει και πάρα πολλούς σε αυτές τις συζητήσεις. Να, να αναφέρω κάτι για αυτό το ερώτημα. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι υπέρ των μεγάλων εκεί συνεδριάσεων ή και των μικρών συνεδριάσεων. Αν είναι να απορροφήσουν όλο το χρόνο μας και να μπορούμε να σκεφτούμε. Καλύτερο θα ήταν σε αυτή την κρίση να έχουμε περισσότερο χρόνο να σκεφτούμε και όχι να είμαστε συνέχεια σε συναντήσεις. Αλλά αυτό το οποίο με εντυπωσίασε στο Συμβούλιο αυτό είναι πως ε, οι συνομιλητές μου είναι αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν τις αποφάσεις και ε, είδαν αυτή τη διαδικασία ε, πάρα πολύ σοβαρά δεδομένου των απαιτήσεων από το χρόνο τους. Οπότε έχουμε επενδύσει πραγματικά πολύ χρόνο και προσπάθεια, γιατί και οι ίδιοι είδαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια τις ε, προκλήσεις και τα προβλήματα που προέκυψαν από την απουσία ακριβώς ενός τέτοιου φόρουμ. Δεν θέλω τώρα να παρέμβω στην τρομερά δύσκολη συζήτηση μεταξύ Ιρλανδικών αρχών και Ευρωπαϊκών αρχών. Σαφώς η Ιρλανδική κυβέρνηση και ο Ιρλανδικός λαός αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις. Και είναι θέμα αυτή της διμερούς ε, συζήτησης να βρεθεί η το, λύση. Βεβαίω, εάν ε, επιμηκυνθεί η λήξη του χρέου ε, είναι ευκολότερο να εξοφληθεί αυτό. Είναι βεβαίω το μάθημα του δημοσίου χρέους εδώ και πολλές δεκαετίες και γι' αυτό ακριβώς το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πάντα δημόσιο χρέο, με πάρα πολύ μεγάλο χρόνο λήξη, κάτι το οποίο μα εξυπηρέτησε σε αυτή την κρίση και είναι ακριβώς το μήνυμα που δίνουμε στον τραπεζικό τομέα και οι ίδιες οι τράπεζες πρέπει να βασίζονται λιγότερο σε βραχυπρόθεσμα κεφάλαια και περισσότερο στην έκδοση χρέους μεγαλύτερου χρόνου λήξης. Δεν βγάζει βεβαίως ε, κανείς περισσότερο χρήμα με αυτόν τον τρόπο και έχουν μάθει οι τράπεζες να δανείζονται βραχυπρόθεσμα και να δανείζουν μακροπρόθεσμα, αλλά μετά το αποτέλεσμα είναι να ζητάς διάσωση από την Κεντρική Τράπεζα και το φορολογούμενο και αυτό βεβαίως ε, είναι κάτι στο οποίο εμείς πρέπει να απαντήσουμε όχι. Δεν είμαστε εκεί απλά για να βγάζουν κέρδη οι τράπεζες και να τους στηρίζουμε εμείς. Οπότε, αυτό βεβαίως είναι κάτι το οποίο θα θέλουν να κάνουν τώρα όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το δράμα που ζούμε το χρηματοπιστωτικό. Δηλαδή η επιμήκυνση της λήξης του χρέους είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστώ πολύ. Θεωρητικά θα έπρεπε να έχουμε μία ακόμη ερώτηση το Έλκαλα ο Βέρνερ, Μπερβάνς, μίλησαν και οι δύο για πάνω από δύο λεπτά, άρα θεωρώ ότι ήταν σαν να κάναν δύο ερωτήσεις. Και δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να ζητήσω συγγνώμη από τους, τις ομάδες της δύο που εκπροσωπούν δύο συνάδελφοι, που τους έκοψα δύο ερωτήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τους αντιπροέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συστημικού Κινδύνου, Πάντοτε η συζήτηση όσο περνάει η ώρα γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρουσα, έτσι ζεσθενόμαστε σιγά σιγά. Ε, ίσως αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου και να σας έχουμε μαζί μας για περισσότερη ώρα την επόμενη φορά. Ευχαριστώ. Uh, Θα περάσουμε στο επόμενο θέμα με τη συνέκταση της ΚΕΙ μετά από κανένα δύο-τρία λεπτά. Okay, if everybody... Λοιπόν, αν γυρίσατε όλοι, περνάμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Έκθεση K. Swinburne για την ελεγκτική πολιτική και διδάγματα που αντλήθηκαν από την κλίση. Θα εξετάσουμε τις ε, τροπολογίες, βεβαίως η ε, κατά κύριο λόγο αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή των Okay. Είμαι πάρα πολύ σύντομη σήμερα κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι ήδη ήταν πάρα πολύ μικρό το χρονοδιάγραμμα που είχαμε λόγω και των πασχαλινών διακοπών και κάποιοι είτε πριν τις διακοπές είτε τώρα δεν ήταν διαθέσιμοι. Το κείμενο το συμβαστικό λοιπόν μόλις τώρα σας το προτείνω και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Βέβαια προσπάθησα να είμαι σε επαφή με τους ε, περισσότερους κοιόδης ε, και με την ομάδα από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Αν, βλέπ, Όπω βλέπετε από τι που έχουν κατατεθεί και από την ΕΚΟΝ και από την ε, Γιούρη, είναι ευρύτατε οι απόψει ε, σε ό,τι αφορά το μέλλον του λογιστικού ελέγχου, τόσο στην δική μα επιτροπή όσο και στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Θα πρότεινα λοιπόν όλες οι, όλα τα αιτήματα του Κοινοβουλίου μας ε, στην Επιτροπή την Ευρωπαϊκή να στηρίζονται πάντα και να τεκμηριώνονται από πολύ καλές εκτιμήσεις ε, ε, επιπτώσεων, ώστε όταν έχουμε την τελική νομοθετική πρόταση αυτή να βασίζεται σε στέρεα βάση. Και νομίζω ότι το βασικό στοιχείο κάθε τροπολογίας είναι ο στόχος να έχουμε υψηλή ποιότητα λογιστικού ελέγχου σε όλους τους τομείς. Και νομίζω ότι εξίσου σημαντικό είναι να υπάρχει ένα σειρμός σε όλες τις τροπολογίες, δηλαδή με τον ένα τον άλλο τρόπο να αυξηθούν οι συμμετέχοντες που προσφέρουν ε, υπηρεσίες λογιστικού ελέγχου και ιδίως από το κατσατικό προβλεπόμενο εξωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ώστε οποιαδήποτε ωφέλη από την αύξηση του αριθμού των ελεγκτών να μην οδηγήσει σε δυσανάλογη αύξηση του κόστους του καταστατικώς προβλεπόμενου έλεγχου για τις ευρωπαϊκές εταιρείε. Μετά από πολλές συζητήσεις και από την ανάγνωση πολλών τροπολογιών πλέον νομίζω ότι είμαι σε θέση να μπορώ να δεχθώ ότι το πρότυπο, το λογιστικό, πρέπει να παραμείνει σε όλους τους τομείς και ίσως να κάνουμε ε, μια διακριτική μεταχείριση, μάλλον η πρόβληψη για μια διακριτική μεταχείριση του, χρημα, του χρηματοπιστωτικού τομέα να είναι ένα βήμα ε, υπερβολικό, νομίζω. Επίσης, νομίζω ότι ένα από τα κοινά θέματα είναι ότι ο λογιστικός έλεγχος συμβαδίζει με την εταιρική διακυβέρνηση. Οι ελεγκτές μπορούν να κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά πρέπει να υπάρχουν ε, για την αναφορά και την ε, συμπεριφορά και για τις ε, εταιρείε. Άρα υπάρχουν κάποια κοινά θέματα που διατρέχουν στις ε, τα είδαμε και τα ακούσαμε και στις συζητήσεις, τα είδαμε ε, την, με τον κύριο Μάση Πιθάλγο και με τους Σκιώδης και θα σας θα δώσω μάλλον στους κοιόδες ηγητές απόψε το τελευταίο, ε, την τελευταία εκδοχή του συμβαστικού κειμένου. Ζητώ για μια ακόμη φορά συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι σε καμιά δύο ημέρες θα είμαστε πλέον έτοιμοι. Έτσι λέει Η Άστρη Λούλινγκ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η έκθεση Σουίνμπερ ευτυχώς προσανατολίζεται προς θέσεις ε, λιγότερο ακαμπτές από αυτές που έχει η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων για ορισμένα θέματα και νομίζω ότι σέβεται το ρόλο που έχουμε στην Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων που πραγματικά κατά προτεραιότητα και κυρίως μας ανησυχούν οι πρακτικές επιπτώσεις που θα, έχει, που οργανώσει μας. Και δεν είμαστε τόσο πολύ λεπτολόγοι στα δικανικά και νομικά θέματα. Νομίζω ότι εύκολο, ε, εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι κάποιες διατάξεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη και θα πρέπει να καταλήξει ο ίδιος ο τομέας και ο κλάδος λογιστικού ελέγχου σε κάποια ε, συμπεράσματα. Υπάρχουν μεταρρυθμίσεις, υπάρχουν μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν ούτως ώστε να έχουμε μια καλύτερη διακυβέρνηση για να μην έχουμε συστημικές κρίσεις σαν αυτή την οποία βιώσαμε. Έχω καταθέσει μια τροπολογία που ζητεί μεταρρύθμιση του λογιστικού ελέγχου να ενταχθεί στο γενικό πλαίσιο της εταιρική διακυβέρνησης. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι εάν αντιμετωπίσουμε απομονωμένα τα προβλήματα, χωρίς να φροντίσουμε να υπάρχει συνέπεια και συνεκτικότητα, θα κάνουμε λάθος. Και είναι σημαντικό να έχουμε μια καλή συνολική εικόνα του όλου προβλήματος, της καλής εταιρικής διακυβέρνησης υπό το πρίσμα των εμπειριών των τελευταίων ετών και γι' αυτό ζητώ να έχουμε μια συνολική εικόνα και όχι μια πάρα πολύ λεπτομεριακή ανάλυση δευτερο, δευτερόντων ε, ζητημάτων. Ελπίζω να ληφθεί υπόψη η τροπολογία μου από την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Okay, that was a slight uh, mistake there because uh, Marcus is actually speaking on behalf of Otto. Μάλιστα, ε, ήταν κάποιο μικρό, μικρό λαθάκι αυτό βεβαίως στη σειρά. Με συγχωρείτε λέει η κυρία Λούλε. Μάρκους, ε, θέλετε να λάβετε τώρα τον λόγο. Εάν, εάν σβήσει το μικρόφωνο και η κυρία Λούλινγκ, θα είναι όλα καλύτερα. Ο κύριος Κάρας μου ζήτησε να πω λίγα λόγια γιατί αναρώνει αυτή τη στιγμή και σύντομα θα είναι στην διάθεσή μας και βεβαίω ξέρετε πως έχει καταθέσει και τις σχετικές ε, προτάσεις του. Βεβαίω πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε το εάν υπήρξε κάποια συνεισφορά ή μη στην ε, κρίση. Κάτι το οποίο βεβαίω δεν απαντάτε τόσο ξεκάθαρα από την αξιολόγηση επιπτώσεων και θα πρέπει να το δούμε αυτό πριν ε, περάσουμε σε τυχόν ρυθμίσεις. Ε, αν έχουμε εδώ πέρα την αίσθηση πως οι ελεγκτές και η ποιότητα του ελέγχου είναι αυτή η οποία έφταιγε, δεν ξέρω και δεν απαντάει εδώ πέρα νομίζω και το έγγραφο το εάν υπάρχει όντως μια τέτοια αιτιώδης σχέση. Κατόπιν η Κομισιόν ασκεί κριτική στο ότι υπάρχουν τέσσερις μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες αλλά από την άλλη όλες οι διαδικασίες οι οποίες περιγράφονται εδώ πέρα και προκήρυξης ε, διαγωνισμού ε, μάλλον ε, θα διώξουν και θα οθήσουν εκτός αγοράς τις μικρομεσαίες εταιρείες και θα μείνουν ακόμη λιγότερες. Οπότε δεν ξέρω εάν είναι αυτή η σωστή προσέγγιση προκήρυξης διαγωνισμών και αλλαγή δηλαδή. Πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό και οπωσδήποτε θα το κάνει ο συνάδελφος ο κύριος Κάρα στις διαπραγματεύσεις με την κυρία Σουίνμπορν, την οποία ευχαριστώ επί τη ευκαιρία. Δεύτερον, υποχρεωτικές τέτοιες ε, ε, πέραν του ζητήματος της ποιότητας του ελέγχου και θα πρέπει βεβαίως να δούμε αν θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο ή αν μπορούν να υπάρχουν ε, και άλλες επαρκείς ε, διαδικασίες ε, διαφανείς που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν περισσότερη διαφάνεια στην αγορά. Και τελευταίο θέμα για τον έλεγχο. Τον κοινό έλεγχο. Υπάρχουν εδώ πέρα κάποιες εμπειρίες και δεν ξέρουμε εάν θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την οδό. Νομίζω πως η κυρία Σουίνμπερν έχει κάνει κάποιες παρατηρήσεις ε, στην ε, έκθεσή της ε, πολύ επιφυλακτικές. γιατί δεν νομίζω πως επαρκούν τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε για να μιλήσουμε για κάποια βελτίωση της κατάστασης. Οπότε θα μπορέσουμε νομίζω να καταλήξουμε σε μια γνωμοδότηση που θα δώσουμε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και βεβαίως το βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι το εάν συνεισέφερε ε, στην κρίση η πολιτική ελέγχου ναι ή όχι και αν δεν συνεισέφερε δεν χρειάζεται να καταλήξουμε σε πάρα πολύ μεγάλες ε, και σοβαρές ρυθμίσεις εδώ πέρα, κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι η ε, πρόθεση εδώ πέρα. Και θα πρέπει βεβαίως ε, να δούμε το πώς θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να μην μείνουν, όπως σας είπα, μόνο οι τέσσερις μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες. Και ξέρετε πως με, τις αλλαγές αυτές, ε, με την αλλαγή αυτή κάθε τέσσερα χρόνια από ό,τι φαίνεται οδηγούμαστε σε μία αύξηση της ε, ποιότητας. Δεν ξέρω αν είναι βελτίωση αυτή της ε, κατάστασης όσον αφορά τα αποτελέσματα του ελέγχου. Οπότε εμείς θα έπρεπε να ζητήσουμε να ελέγξουμε και τους υπό έλεγχο και να μην έχουν τη δυνατότητα οι ελεγκτές να, να επανεπεξεργάζονται συνεχώς τα πράγματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. σου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγητριά μας γιατί έχει υποβάλει συμβιβαστικές τροπολογίες που θα μας επιτρέψουν να ξεκινήσουμε τη συζήτηση διευρύνοντας ίσως και το πεδίο, την εμβέλεια σε σχέση με αυτή που ίδια θα ήθελα αρχικά ίσως να δοθεί σε αυτή τη γνωμοδότηση. Παρεμβαίνω μετά τον ε, Βέρνερ. Θα ήθελα πάντως να μιλήσω λίγο για την διάτρωση μεταξύ της πράσινης αυτής βίβλου και της κρίσης. Η λογιστική έλεγχη δεν είναι υπεύθυνη για την κρίση, αλλά τα γραφεία των ελεγκτών, ε, τι στόχο και ρόλο μάλλον έχουν, να ελέγχουν τις επιχειρήσεις και βέβαια θα πρέπει ε, η χρηματοδότηση να είναι υγιής. Δεν ήταν και δεν έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου οι εταιρείε ε, λογιστικού ελέγχου. Αν λοιπόν δεν ελέγχουν ε, σωστά τους λογαριασμούς των επιχειρήσεων, εκ των οποίων πολλές είναι και μεγάλες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, για να το πω έτσι μαλακά, ήταν ελληματική η λειτουργία αυτών των γραφείων. Δεν λέω ότι φταίνει για την κρίση, αλλά συνεισέφεραν δεν άσκησαν το σωστό κοινωνικό ρόλο υπό την έννοια της διάθρωσης της κοινωνίας που ήταν να προειδοποιήσουν σε σχέση με την κατάσταση των λογαριασμών και τον τρόπο χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και νομίζω ότι αυτό ε, είναι κάτι που πρέπει να μας βρει σύμφωνος εδώ στην Επιτροπή μας. Δεν λέω ότι είμαστε μετά την, ε, την επαύριο της Ένρων, αλλά είμαστε την επαύριο μιας κρίσης παρόλα αυτά. Και Ξέρουμε τι έγινε με τα subprimes. Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις ε, πριν να ε, σχολιάσω τις συμβαστικές προτάσεις που προτείνει η Σίγητρε. Πρώτο, πρέπει να κουβεντιάσουμε το πεδίο εφαρμογή πράσινη βίβλου. Γιατί αρχικά η εισηγήτριά μα μας είχε προτείνει να κάνουμε λόγο μόνο για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σημαντικά από συστημική άποψη. Σύφη. τέλο πάντων που έχουν συστημικού κινδύνου. Υπήρχαν πολλέ τροπολογίε διεύνηση του πεδίου ώστε να συμπεριλάβει γενικώ ε, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αλλά δεν διακυβεύεται αυτό με την πράσινη βίβλο. Εδώ μιλάμε για όλε τι επιχειρήσει. Όλε οι επιχειρήσει που προσφεύγουν, που καταφεύγουν στον έλεγχο, στο λογιστικό έλεγχο. Εμεί είμαστε όχι Χρηματοπιστωτική Επιτροπή, είμαστε Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή. Πρέπει να δούμε την οικονομική διάσταση επομένω. Και όλε οι επιχειρήσει όταν πρέπει να επαληθεύσουν την κατάσταση των λογαριασμών του, και είχαμε και την 8η οδηγία με τον Wolf Klintz γιατί τότε, δεν είδαμε όλου του χρηματοπιστωτικού οργανισμού. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναδούμε τις διατυπώσεις και υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ακόμη ειδικότερο ζήτημα για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες της Ένωσης. Αλλά ειλικρινά ελπίζω να μην περιορίσουμε τη γνωμοδότησή μα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να καταφέρουν στο λογιστικό έλεγχο και εμείς πρέπει όλες τις επιχειρήσεις να τι εξετάσουμε και ιδίω τις εισηγμένες. Ελπίζω να εμβαθύνουμε λοιπόν στη συζήτηση. Τώρα, η συγγήτρια μα έχει παρουσιάσει μια συμβαστική πρόταση. Αλλά τι άποψη έχετε για τι τροπολογίε που δεν καλύπτονται από τι συμβαστικέ, κυρία Σούμπορν, δεν μα είπατε. Εμεί από πλευρά των Δημοκρατών έχουμε υποβάλει κάποιε τροπολογίε, των οποίων δύο μου φαίνονται σημαντικέ και θα ήθελα να ακούσω την άποψη τη συγγήτρια. Πρώτα απ' όλα, τροπολογία 6, που μιλά για τον κίνδυνο που θα αντιπροσώπευε η χρεοκοπία μίας από τις μεγάλες τέσσερις τράπεζες. Νομίζω ότι έτσι μπορούμε να θέσουμε και το ζήτημα της συγκέντρωσης και το τι κίνδυνο συνεπάγεται αυτό για το όλο σύστημα. Και δεύτερον, η τροπολογία 80. Φαντάζομαι ότι είναι μια πιο πολύπλοκη τροπολογία να τη συζητήσουμε εδώ μεταξύ μας, αλλά θεωρώ ότι είναι τροπολογία πολύ σημαντική. Όχι μέσω αυτής της νομοθεσίας να επιβάλλουμε στους ελεγκτές την ε, ανάγκη να επιβάλλουν την, ε, εταιρική και, την κοινωνική και περιβαλλοντική εταιρική ευθύνη. Αλλά, όπως είχαμε πει, να γίνει μια συζήτηση για αυτό το σημείο. Ανησύχησε η κυρία Λούλινγκ. Είπε ότι μήπως δούμε αυτό το θέμα παράλληλα με θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Ακούστε. Μέσω από της τροπολογίας 80 αυτό που μπορεί να γίνει είναι αυτά τα δύο στοιχεία να τα συνδέσουμε κάπως. Και αφού αναφέρεται και στην πράσινη βίβλο αυτό το θέμα, γιατί να μην το αναφέρουμε. Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι είναι αρμοδιότητα καταρχά τη Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Δεν απαγορεύεται όμω στην Επιτροπή μα να δούμε το θέμα τη κοινωνική και περιβαλλοντική εταιρική ευθύνη. Και, και άλλε φορέ έχουμε ασκήσει τα προνομιά μας και τις, ε, τα δικαιώματά μας. Τώρα, στην τροπολογία είναι το σαν σε πρεσέδο. Λείπει το τελευταίο τμήμα της τροπολογίας, που όμως νομίζω ότι θα έπρεπε να συμπεριληφθεί. Συμβιβαστική 2. Πάλι, τι εμβέλεια, τι βελνικές θέλουμε να έχει η πρόταση γνωμοδότησή μας. Εντάξει, δεν το... Δεν ξαναλέω αυτά που είπα πριν. Τώρα τροπολογία 4 στην τροπολογία 37 υπάρχει ένα τμήμα δική μα τροπολογία εννοώ 37 που δεν το συμπεριλαμβάνει συμβαστική 4. Η ποιότητα του ελέγχου είναι σημαντική γιατί επαναλαμβάνετε την ιδέα ότι πρόκειται για ένα κοινωνικό, ε, σημαντικό κοινωνικό λειτουργήμα. Αλλά εγώ σας προτείνω να κάνετε να το δείτε λίγο πιο αναλυτικά. Γιατί λέμε είναι σημαντικό, γιατί επιτρέπεται η πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. αν υπάρχει καλός έλεγχος ε, των λογαριασμών, υπάρχει καλύτερη δυνατότητα προσέλκυσης χρηματοδότησης ε, και από τις τράπεζες. Και το στοιχείο της εταιρικής διακυβέρνησης όχι γιατί πρέπει να κολλησιεργήσουμε και να πούμε ότι μόνο στο πλαίσιο του τη ε, εταιρική διακυβέρνηση θα το συστήσουμε, αλλά την επαύριο αυτή τη κρίση και ακριβώ αυτά τα στοιχεία τη εταιρική διακυβέρνηση, άρα τη ποιότητα των εγγράφων βάσει των οποίων μπορεί να γίνει κοινωνικό διάλογο, ε, μπορεί να. Ε, συνδεθούν και τα στοιχεία της εταιρική διακυβέρνησης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας προτείνω λοιπόν να το πείτε πιο ρητά. Συμβαστική 5. Σε σχέση με εσωτερικούς εξωτερικούς ελεγκτές, νομίζω ότι πρέπει να το διατυπώσετε λίγο πιο τολμηρά. Συμβαστική 6 είναι λίγο αδύναμη και ελπίζω να μπορέσουμε να την ξανασυζητήσουμε. Συμβαστική 7, μια πολύ καλή βάση συζήτηση νομίζω και σας ευχαριστώ γιατί δείξατε πολύ ανοιχτό πνεύμα και λάβατε υπόψη κάποιες από τις προτάσεις μας. Βέβαια, εξακολουθεί να υπάρχει εδώ το ζήτημα του ελληνικού της νομοδότησης. Περιοριζόμαστε στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή πάμε πιο πέρα. Συμβαστική 8. Νομίζω ότι υπάρχει ένα τυπογραφικό. Proportionate way πρέπει να λέει. Και μιλάω τώρα για την τροπολογία 102 της ε, Προέδρου μας, Σάρον που μας καλεί να εξετάσουμε αυτό το θέμα της αναλογικότητας. Η διατύπωση που σας πρότεινα, δηλαδή να ενδιαφερθούμε απλά για τις επιχειρήσεις της διασυνορικές cross-border, λύνει το πρόβλημα. Ε, νομίζω ότι ορίζει καλύτερα το πεδίο που θέλουμε να καλύψουμε. Συμβαστική 11. Νομίζω ότι υπάρχει μια διαπραγματευτική βάση, υπάρχουν κάποιες αντιπροτάσεις που θα ήθελα να σας υποβάλω για να ενισχύσουμε λίγο την πρότασή μας. Και σε ό,τι αφορά τη συμβαστική 12, με αρχή το κείμενο της κυρίας Λούλινγκ που δυστυχώς έφυγε από την αίθουσα, δεν έχω πρόβλημα εγώ να πούμε ότι όλα πρέπει να είναι παντού, αλλά δεν θα συμφωνήσω αν αυτό οδηγήσει σε καθυστερήσεις και μία επίτευξη πρόοδου. Εγώ θα ήθελα να το βάλουμε μαζί με την εταιρική διακυβέρνηση. Αλλά επαναλαμβάνω όχι να γίνει λόγο για να μην προχωρήσουμε μέσα στο θέμα του λογιστικού ελέγχου. Ναι, δυστυχώ δεν έχω αντίγραφο των συμβαστικών τροπολογιών, τουλάχιστον αυτών στι οποίε αναφερόταν η υπέρβανος. Βολφ Κλίντς. Ευχαριστώ. Θα μου επιτρέψετε να επισημάνω ορισμένα πράγματα. συμφωνώ με αυτά που λέξαν ότι ο έλεγχο είναι έλεγχο και δεν θα πρέπει εδώ να κάνουμε διαχωρισμό ε, σε τομεί, γιατί τότε θα είναι λάθο η προσπάθειά μα. Και εγώ θεωρώ ότι πράγματι ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να συμβαδίζει με την corporate governance. Και επιτρέψτε μου και κάποια σύντομα σχόλια. Όσον αφορά τώρα τις, ε, την παροχή συμβουλών, δηλαδή όχι την, τον κλασικό έλεγχο, αλλά την παροχή πλησίων σε όλους τους τομείς, εκεί πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι τόσο επικριτικός όσο η Κέιτ στην συμβατική της τροπολογία υπαρτιμών 5. Εγώ θεωρώ ότι οποτεδήποτε ε, παρέχονται υπηρεσίες ε, που ξεπερνούν τον καθαρό έλεγχο, είναι όμως υπηρεσίες που είναι απαραίτητο να προσφερθούν όπως οι ε, φορολογικές υπηρεσίες. Αν πραγματικά υπάρχει ενδιαφέρον, τότε εδώ θα πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός. Όμως καταρχήν πιστεύω ότι θα πρέπει ε, να παραμείνει αυτή η παροχή υπηρεσιών στους ελεγκτές, αλλά την ε, εντολή δεν θα πρέπει να τη δίνουν τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, γιατί πράγματι στην περίπτωση αυτή ελοχεύει ο κίνδυνο, η παροχή υπηρεσιών να είναι κομμένη και ραμμένη στα δικά τους τα μέτρα. Αυτό θα πρέπει να γίνεται περισσότερο από μια ε, επιτροπή ελέγχου. Η, ε, τα συμβόλαια που συνδέονται με παροχή υπηρεσιών θα πρέπει να συντάσσονται από την Επιτροπή Ελέγχων, δηλαδή από τα non-executive board members και όχι από την εκτελεστική επιτροπή. Συμβαστική 6. Αν δεν πω τίποτα για κάποια συμβαστική πρόταση, αυτό σημαίνει ότι συμφωνώ. Πάω τώρα στην 6 την συμβαστική πρόταση 6, όπου γίνεται λόγος για της δημοπρασίας, τους δημόσιους διαγωνισμούς. Εκεί συμφωνώ με τον συνάδελφο κύριο Φέιμπερτο ε, κατά πόσον ε, εδώ δεν καταβάλουμε προσπάθεια να σταθεροποιήσουμε περαιτέρω τους μεγάλους, δεν το ξέρω, είμαι λίγο επιφυλακτικό. Νομίζω η λύση που βρήκαμε το 2006 ότι... Ε, να αν υπάρχει μια εσωτερική εναλλαγή, αυτό για μένα αρκεί όχι μόνο στην εταιρεία, αλλά στον εσωτερικό έλεγχο. Η 11 αφορά τις, τους κοινούς ελέγχους joint audits. Εκεί πρέπει να πω ότι είναι αλήθεια, ισχύει. Στη Γαλλία έχουμε μεικτή εμπειρία με τον ε, υποχρεωτικό κοινό έλεγχο. Εγώ από δική μου εμπειρία ως ε, για πολλά χρόνια ε, πρόεδρος μιας εταιρείας που είχε σχέση με ελέγχους, όπου είχαμε κοινούς ελέγχους, αυτό όλες τις φορές αποδείχτηκε ιδιαίτερα ε, αποδοτικό, παραγωγικό. Γι' αυτό είχαμε συνέχεια κοινού ελέγχου και γι' αυτό λοιπόν για μένα αυτή είναι η μόνη δυνατότητα για εταιρείε που έχουν τη δυνατότητα να αυξηθούν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορούν να είναι ανταγωνιστικέ οι εταιρείε αυτέ να κάνουν κοινού ελέγχου. Και έχω συγκεκριμένο παράδειγμα η εταιρεία BDO ε, στη Γερμανία. Παλαιότερα ήταν περιφερειακή εμβέλεια και σήμερα η εταιρεία αυτή έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο έτσι ώστε να μπορεί να σταθεί αυτή στα της και σε διεθνές επίπεδο. Ευχαριστώ. Σβέν, κατόπιν. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και ειδικά την ΚΕΙ για το σχέδιο έκθεσης και αναμένω την συζήτηση αυτών των ζητημάτων. Θα ήθελα όμως να αναφέρω κάποια ζητήματα τα οποία μας ανησυχούν και σας ευχαριστώ που συμπεριλάβατε και κάποιες ιδέες μας. Πρώτα απ' όλα, το θέμα της ευθύνη για την κρίση. Εξαπλάγει λίγο από τις παρατηρήσεις ε, του Μάρκους, ε, γιατί είναι σαφές. Νομίζω πως υπήρχε πρόβλημα. Υπήρχε πρόβλημα καθώς σοβαροί κίνδυνοι δεν ε, έγιναν αντιληπτοί και αυτό οδήγησε σε λάθος επενδύσεις και συνεισέφερε στην κρίση. Οπότε πρέπει να το λάβουμε αυτό σοβαρά υπόψη. Και αυτό δεν ήταν τόσο πολύ το σχόλιο της ε, ΚΕΙ, αλλά νομίζω πως η έκθεση πρέπει να το αναφέρει. Ε, το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να πω, το οποίο είναι σημαντικό για εμάς, ποιος επιλέγει τον ελεκτή. Σαφώς υπάρχει κίνδυνος ε, πιθανών αντικρώμενων συμφερόντων, γι' αυτό προτείναμε να υπάρχει ένας δεύτερος υποχρεωτικό έλεγχος που δεν θα, ε, ε, και ελεγκτής που δεν θα επιλέγει η εταιρεία αλλά κάποιος τρίτος. Μία παρόμοια συζήτηση είχαμε για τις υπηρεσίες ε, αξιολόγησης. Η καθαρότερη λύση είναι αυτή λοιπόν για να αποφύγουμε το ότι ο ελεγκτής θα είναι ελαστικός γιατί γνωρίζει πως ε, το επίπεδο διαφάνειας ε, θα αποτελέσει κριτήριο για την επόμενη πρόσφορα. Οπότε το σαφές αντικρουόμενο συμφέρον που είναι εγγενές στο σύστημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια τέτοια λύση. Εμεί προτείναμε μια λύση, δεν βλέπουμε αυτή τη λύση μέχρι στιγμή στο σχέδιο έκθεσης. Δεύτερον, θα θέλαμε να δούμε ισχυρότερο ρόλο για τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, ειδικά όσον αφορά τις μεγάλες εταιρείες. Εκεί πέρα θα πρέπει βεβαίως να επανέλθουμε στη συζήτηση επιπλέον. Και είδα και παρόμοιες παρατηρήσεις και από κάποιους συναδέλφους από τον Wolf Κλίντς για το θέμα της ευθύνης. Η ευθύνη η αστική ευθύνη είναι πάρα πολύ σημαντική σε όλες τις οικονομίες της αγοράς για να υπάρχουν τα κατάλληλα κίνητρα. Πρέπει να είμαστε λοιπόν σαφείς στο ζήτημα της ευθύνη και ίσως και κάπως πιο ε, έντονη από η πρόταση όσο έχει αυτή τη στιγμή. Επιπλέον έχω κάποιο ζήτημα με την θέση που ανέφερε μόλις ο Βόλφ για την σύνδεση μεταξύ υπηρεσιών άλλων και ελέγχων. Είναι σαφές πως υπάρχει εδώ πέρα ο κίνδυνος της συμφερόντων και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτό το οποίο είπε ο Μάρκους για τον κίνδυνο για τις μικρότερες εταιρείες που θα κινδυνεύσουν από κάποιες από τις ε, ρυθμιστικές δομές είναι πολύ σοβαρό αυτό πράγματι και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί η λύση που προτείνουμε να υπάρχουν τρίτη, κάποιος τρίτος ο οποίος θα διασφαλίσει δεύτερο υποχρεωτικό έλεγχο που ελπίζουμε να μην είναι κάποιοι από τις μεγάλες τέσσερις εταιρείες θα βοηθήσει ειδικά τις ε, μικρομεσαίες και αναμένω την απάντησή σας εδώ πέρα και τη γνώμη σας. Και τέλος, δεν έχω δει δεν ξέρω, ίσως να μην το διάβασα κιόλας γιατί το έλαβα πολύ αργά. Ζητήσαμε να μας πει η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού τι γίνεται με τη δομή της αγοράς και καλό θα ήταν νομίζω να ζητήσουμε από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού να κάνει μια πλήρη έρευνα και αξιολόγηση της αγοράς αυτής. Ευχαριστώ πάρα πολύ και αναμένω τη συζήτησή μας you. Uh, Now, Diego Feio. Muito obrigado. Muito obrigado, Sharon. Eu queria começar por cumprimentar a Kay, bem como os... Ήθελα να ξεκινήσω δίνοντας συγχαρητήρια στην ΚΕΙ για την γνωμοδότησή της, για τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι στιγμής και θα ήθελα να πω πως προφανώς ένας γενικός στόχος που συμμεριζόμαστε όλοι στην Επιτροπή μας είναι να έχουμε καλύτερες έλεκτικες υπηρεσίες. Επίσης συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε ο Μάρκους Φέμπερ για την κρίση και τη σχέση ε, κρίσης και του ζητήματος που μας απασχολεί τώρα εδώ πέρα. Δεν θεωρώ πως αν υπάρχει μια κρίση πρέπει αυτομάτως να αλλάξουν τα πάντα. Να υπάρχει ένα γενικό πρόβλημα το οποίο θα ήθελα να φίξω. το οποίο είναι το αν έχει περάσει αρκετός χρόνος από την εφαρμογή της 8ης οδηγίας για να βγάλουμε συμπεράσματα. Μόλις πρόσφατα κάποια κράτη-μέλη μετέφεραν στην εθνική τους νομοθεσία την 8 οδηγία και πρέπει να δούμε πρώτα απ' όλα τα αποτελέσματα. Γι' αυτό θεωρώ πως δεν πρέπει να βιαστούμε. Και υπάρχουν ε, και κάποια συγκεκριμένα ζητήματα που ούτως ή άλλως θα αποτελέσουν αντικείμενο προσοχής της Επιτροπής μας. Το θέμα των ελεγκτικών εταιριών και της εναλλαγής τους, αν θα πρέπει να εναλλάσσονται εταιρείε ή αρκεί να εναλλάσσεται ο ελεγκτής. Μετά υπάρχει το ζήτημα του αποκλεισμού λοιπόν υπηρεσιών πλην ε, των ελεγκτικών και κατόπιν ο ρόλος των ελεγκτών και σε σχέση με την κρίση που ε, ζούμε το Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε με περισσότερη διαφάνεια, με περισσότερο διάλογο μεταξύ έλεγκτων και ρυθμιστικών αρχών και βεβαίως περισσότερο βάρος πρέπει να δοθεί στις ε, ελεγκτικές επιτροπές. Αυτά τα ζητήματα πρέπει να δούμε, γι' αυτό θα ήθελα πάλι να συγχαρώ την ε, εισηγήτρια για τις κατευθύνσεις που έδωσε στην συζήτηση, συζήτηση βεβαίω η οποία θα μας απασχολήσει. Βέρνερ Λάγκεν. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι δεν πρέπει να κάνει κανείς το λάθος ε, και να αναθέσει, ε, να μετακυλήσει στις ελεκτικές εταιρείες ε, την ευθύνη για την κρίση. Γιατί εκεί ήταν οι οίκοι αξιολόγηση που έκαναν την αξιολόγηση χωρίς όμως να προβλέψουν στάθμιση των κινδύνων και οι εποπτικές αρχές υιοθέτησαν αυτές τις απόψεις ε, χωρίς να κάνουν δικούς ελέγχους. Άρα δηλαδή να μην πετάξουμε και το νερό το μωρό με τα πόνερα. Αυτό που έχει σημασία είναι να κάνουμε έναν καλό απολογισμό με που βάλουν σωστά ερωτήματα και εγώ συμφωνώ με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι Φέμπερ και Κλίντς. Δηλαδή πρώτον, όσον αφορά ε, τους δημόσιους διαγωνισμούς, το θέμα των τεσσάρων μεγαλύτερων ελεγκτικών εταιριών, ε, να ε, διαχωρίζεται το θέμα του ελέγχου ε, και της ανάθεσης εντολής, αυτά είναι θετικά πράγματα με τα οποία μπορούμε να επιτύχουμε πολλούς ε, στόχους ε, ε, στον ανταγωνισμό που αναφέρεται ότι κάθε κάποια οκτώ χρόνια θα πρέπει να γίνεται κάποιος δημόσιος ανταγωνισμός. Οι μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επεκταθούν. Από την άλλη βέβαια η άλλη λύση είναι να καταστρέψουμε τις μεγάλες εταιρείες αλλά και αυτό κανείς δεν το θέλει. Γι' αυτό θεωρώ ότι εδώ δεν θα πρέπει να συγχαίουμε ποιο φέρει την ευθύνη. Κυρίως θα πρέπει να επιτρέπουμε τους κοινού ελέγχους, να μην τους απαγορεύουμε δουλεύουμε στο μέλλον, γιατί με τον τρόπο αυτό προσφέρεται η δυνατότητα ε, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συνενώνονται και να ε, δημιουργούν ένα μέγεθος έτσι ώστε να μπορούν να ελέγχουν μια εταιρεία. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το σημαντικό και θεωρώ ότι ως έχουν τα πράγματα, εμείς ε, έτσι κι αλλιώς ως Οικονομική Επιτροπή ε, καλούμεθα να έχουμε κατά νου τα συμφέροντα του κλάδου ε, και να μην αποδίδουμε σε λάθους αποδέκτες τα αίτια και την ευθύνη της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Έχω κάποιες τροπολογίες δεν θα πρέπει να εκπλαγείτε με αυτές, γιατί υπάρχουν αρκετά που έχουν ήδη γίνει στο corporate governance. Καταρχήν, ε, θέλω να κάνω κάποιες σχόλια. Σε απάντηση αυτών που είπε ο Βέρνερ, νομίζω ότι οι ε, επόπτες ε, την έβγαλαν ε, αυρόχης ποσή από την κρίση. Δεν θέλουμε να πετάξουμε το νερό με τα πόνερα, αλλά εγώ θεωρώ ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο διάλογος μεταξύ ε, ελεγκτού και επιθεωρητού είναι επαρκής ε, για να εξοβελιστούν οποιασδήποτε υποψίες. Αυτό είναι κάτι δύσκολο. Είναι δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Σε πολλά κράτη-μέλη Υπήρχε κάτι τέτοιο. Ας πούμε υπήρχε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, και ακούσατε και προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν. Άλλες πάλι φορές ε, έχετε επίσης δίκιο ότι ε, συνεχίζουν τα προβλήματα. Τώρα όμως ζούμε σε μια εποχή όπου όλα είναι συνδεμένα μεταξύ τους. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τη δυνατότητα ε, να γίνουμε λίγο πιο συστηματικοί και αυτό έχει σχέση με την διασύνδεση και με την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή, οι αρχές. Εγώ δεν θέλω να αποκλειστεί τίποτα που να έχει σχέση με όλα αυτά και που να έχει σχέση ε, με τις χρηματοψηφιωτικές υπηρεσίες. Εγώ συμφωνώ, έλεγχος είναι απλά έλεγχος και δεν θέλουμε να έχουμε δύο διαφορετικούς δρόμους. Υπάρχουν και πράγματα ε, που πρέπει να γίνουν στον τομέα των χρηματοψηφιστικών εταιριών, ε, στους ε, επίπλαστους, στους ψευδεπίγραφους ε, διαγωνισμούς. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε το θέμα και στον Αμένο Βασίλειο και στον Βέλιο. Και πρέπει να πω ότι μερικές φορές δημιουργούνται μερικές ομάδες και διαρωτώνται τι νοσή είναι να υποβάλει έναν λογικό, μια λογική προσφορά σε ε, διαγωνισμό. Εγώ ε, οποτεδήποτε συμμετείχα σε κάτι δεν ήταν ψευδεπίγραφος ο διαγωνισμός. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εξετάσουμε και να δουλέψουμε περισσότερο πάνω σε αυτό. Πρέπει να σας πω ότι δεν μου αρέσει να περιορίζονται οι ελεγκτές να κάνουν μόνο ελέγχους. Γιατί αν κάνει κανείς μόνο ελέγχους, τότε δεν θα ασχοληθούν με το θέμα αυτό οι ε, καλύτεροι, πιο ικανοί υπάλληλοι. Θα πρέπει να είναι εκείνοι οι οποίοι ασχολούνται με παροχή συμβουλών για να καταλάβουν και άλλες πλευρές ε, του κλάδου. Αυτό βέβαια δεν θα σημαίνει ότι θα πρέπει ο ίδιος να κάνει και τον έλεγχο και την παροχή συμβουλών. Ε, θα πρέπει να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Πάντως ε, να μην γίνονται και μόνο έλεγχοι γιατί και αυτό δεν δουλεύει καλά. Και εγώ προτείνω σε αυτές τις τέσσερις μεγάλες εταιρείες ότι πρέπει να δούμε λιγάκι το θέμα των κρατικών προμηθειών. Ε, στο Κοινοβούλιο καταθέσαμε προτάσεις, είπαμε ε, στις ε, διαγωνισμούς κρατικών προμηθειών να χρησιμοποιούνται περισσότερο μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, και γιατί να μην κάνουμε το ίδιο και με τους ελέγχους. Δεν είναι καλό να πούμε ότι πρέπει να τους ενθαρρύνουμε, τις μικρομεσαίες κυρίως, και μετά να ανακαλύπτουμε ότι όλοι τελικά πάνε μόνο στις τέσσερις μεγάλες εταιρείες ελέγχου. Εγώ ε, δεν θέλω να φτάσω να πούμε ότι ε, επιβάλλεται δεσμετικά να καταφεύγει κανείς στις μικρομεσές. Να υπάρχει περισσότερο ένα, ε, ένα κριτήριο σύγκρισης για να μπορούμε να διαπιστώσουμε αν έχει υπάρξει βελτίωση. Και αν δεν έχει υπάρξει βελτίωση, τότε εντάξει πρέπει να δούμε ποιο είναι το επόμενο βήμα. Αυτό είναι το πνεύμα των τροπολογιών που κατέθεσα εγώ. Και ελπίζω να τις εγκρίνουν οι συνάδελφοι. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, είναι απασχολημένοι σε τριμερείς συζητήσεις και δεν είναι τόσο να ε, εμπλακούν στις δικές μου όσο θα το επιθυμούσα. Κυρία Σόιμπον, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν αναφέρθηκα στο συμβαστικό κείμενο γιατί ήταν διαθέσιμο ένα, μία ώρα μόλις πριν ξεκινήσει η συνεδρίασή μας και φαντάστηκα ότι κάποιοι συνάδελφοι δεν θα το δουν καν γιατί θα έρχονταν κατευθείαν στην αίθουσα και δεν θα περνούσαν από τα γραφεία τους, άρα ουσιαστικά σκοπίμως δεν το ανέφερα αυτό το συμβαστικό κείμενο, δεν το σχολίασα. Σίγουρα είναι λίγο διαφορετική η κατάσταση σε σχέση με αυτήν που περίμενα, διότι κάπως ε, επισπεύσαμε τα πράγματα. Αύριο θα έχουμε και την συνάντηση με τους ε, Σκιόδης Όπως σας είπα, το κείμενο αυτή τη στιγμή είναι ένα πρώτο σχέδιο. Ε, πράγματι οι διάφορες πολιτικές ομάδες έχουν ε, αρκετές ε, διαφωνίες ό,τι αφορά κάποια από τα μείζωνα ζητήματα, ειδικότερα σε ό,τι αφορά εναλλαγή εσωτερικών εξωτερικών ελεγκτών, ε, τις διαγωνισμούς, αύξηση ανταγωνισμού με, κοινές, με κοινούς ελέγχους ή όχι. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρη και έχω ακούσει πολλοί ισχυρές φωνές να μου λένε ότι η καλύτερη λύση είναι η κοινή έλεγχη και άλλοι να μου λένε το ακριβώς το αντίθετο. Λοιπόν, έχουμε 48 ώρες για να καταλήξουμε κάπου, αλλά πρέπει να σας πω ότι έχω ε, μόλις διανύμει αυτό το συμβιβαστικό κείμενο. Η Περβάνς Μπερές έκανε αναφορά στις τροπολίες που δεν καλύπτονται από το συμβιβαστικό κείμενο. Αυτές θα ψηφιστούν χωριστά. Νομίζω ε, μιλάμε για 25 ξεχωριστές ψηφοφορίες περίπου. Η συγκεκριμένα αναφέρθηκε στις δικές της τροπολογίες, ε, καταρχάς την 6. Εγώ τη δέχομαι την ε, τροπολογία 6, αλλά σε ό,τι αφορά την 80 που επίσης ανέφερες, ε, αυτήν δεν μπορώ να τη δεχθώ, γιατί νομίζω ότι είναι καλύτερα αυτό το ζήτημα να μπει στο πακέτο εταιρική διακυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά την συμβιβαστική 12 την προτιμώ, γιατί αφήνει οι αποφάσεις να γίνουν από κοινού, δίπλα-δίπλα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εταιρική διακυβέρνηση. Πάντως η Επιτροπή μας και η δημοκρατία εν τέλει είναι αυτή η οποία θα καταλήξει στο πώ θα, θα προχωρήσουμε. Νομίζω ότι τις επόμενε 48 ώρες, όπως είπα, ο ρόλος μου είναι να εξισορροπήσω τις απόψεις των ε, πολιτικών ομάδων για τα ζητήματα αυτά που σας είπα. Εγώ προσωπικά δεν έχω ε, πιστεί σε ό,τι αφορά τους κοινού ελέγχους. Δεν θεωρώ ότι εξωτερική αναλλαγή είναι απαραίτητη δεδομένου το ότι έχουμε και την οδηγία ε, την 8η, η οποία είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Η συμβιβαστική μου πρόταση είναι για υποχρεωτικό διαγωνισμό, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση επιπτώσεων οπωσδήποτε. Και δεν θέλουμε να υπάρξει επιπρόσθετο κόστος αθέλητο, αλλά αντίθετα θέλουμε υψηλής ποιότητας λογιστικό έλεγχο χωρίς να επιβαρυνθούν υπερβολικά οι επιχειρήσεις μας. Κάποιοι από εσάς αναφέρατε τις ελεγκτικές υπηρεσίες, το κατά πόσο θα πρέπει να περιορίζουμε τις διάφορες υπηρεσίες και πόσο. Εγώ σε καμιά περίπτωση δεν θα ήθελα να δημιουργούμε ελεγκτικές εταιρείε, αποκλειστικά και μόνο δηλαδή για έλεγχο, αλλά δεν υπάρχει απέτηση για καμία εταιρεία να διαχειρίζεται σύγκρουση συμφερόντων. Δεν θα πρέπει να κάνει τίποτα το οποίο θα απαιτεί ε, το να υπάρχει ένα ολόκληρο κινέζικο τείχος. Θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πολλές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες, πολλές υπηρεσίες και δεν νομίζω ότι περιορίζουμε κανενός την επιλογή λέγοντας ότι δεν μπορείτε να έχετε ένα κινέζικο τείχος όποιος λειτουργεί ε, σε ένα ίδρυμα με κινέζικους τείχους, εκεί θα δει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να ε, υπάρξει μια σωστή διαδικασία και υπάρχουν τελικά διαρροές. Άρα γιατί να γίνει αυτό και γιατί να επιτρέπουμε τέτοιες καταστάσεις. Φυσικά και δεν θέλουμε να μειώσουμε την αξία της εμπειρογνωμοσύνης. Υπάρχουν πολλοί γραμματοπιστωτικοί οργανισμοί, άρα μπορούν διαφορετικές εταιρείε να κάνουν λογιστικό έλεγχο σε διαφορετικά, διαφορετικές δραστηριότητες, διαφορετικά τμήματα. Και έτσι μπορούμε νομίζω να καταλήξουμε σε μια ισορροπημένη εκδοχή του κειμένου. Προσπάθησα κάποιες ατερόκλητες απόψεις να τις συμβιβάσω στο κείμενο το οποίο θα σας ε, διανύμω. Και δεν θέλω αντί για άλογο ε, που ε, αποσκοπούσα να σχεδιάσω να καταλήξει να είναι μια καμήλα. Θα ξεκινήσει λοιπόν ε, η συζήτηση. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων βέβαια είναι η καθήλυνα αρμόδια για, για κάποια ζητήματα. Σε ό,τι αφορά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουμε τον ηγετικό ρόλο εμείς, αλλά και σε ό,τι αφορά την αλληλεπίδραση μεταξύ των ελεκτών που είναι δική μας αρμοδιότητα και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Σε ό,τι αφορά τις ε, τροπολογίες, νομίζω ότι έχουμε υπερβεί αρκετά το πεδίο αρμοδιοτήτων που εγώ θεωρώ ότι πρέπει να έχει η Επιτροπή μας. Η Γιούρη κοιτάζει πάρα πολύ προσεκτικά το πόσο πολύ έχουμε υπερβεί και έχουμε μπει σε ξαναχωράφια. Αλλά θέλω να σας πω ότι Νομίζω ότι μεταξύ των δύο επιτροπών, έτσι λίγο από τις συζητήσεις που είχαμε μέχρι τώρα, μπορούμε να συμβιβαστούμε και να έχουμε έτσι μια εντολή για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στις μελικές διαπραγματεύσεις. Εάν τώρα έχετε σχόλια και αν δεν είστε βέβαια αλλά παρόλα αυτά θέλετε να σχολιάσετε κάτι, ευχαρίστως ε, να λάβω υπόψη οποιασδήποτε παρατηρήσει διαβιβάσετε στο γραφείο μου και θα έχουμε ένα αξιοπρεπές έγγραφο, πιστεύω, την επόμενη εβδομάδα για να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. 9 Μαΐου θα... 9 Μαΐου θα ψηφίσουμε, 24 Μαΐου ψηφίζει η Επιτροπή Γιούρη και πηγαίνουμε για την Ολομέλεια Ιουνίου, Ιουνίου 2, τη δεύτερη Ολομέλεια του Ιουνίου για την Ολομέλεια όπως είπα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν αυτό το σημείο και θέλω τώρα να δώσω το λόγο στον αντιπρόεδρο της ΕΚΤ γιατί θα έχουμε στη συνέχεια την ετήσια έκθεση ΕΚΤ 2010 σε λίγο.

Right, thank you everybody um, and uh, welcome to Victor Constantio. Yet another... Καλώς ήρθατε. Άλλος ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βαρεθεί να με βλέπει τις τελευταίες εβδομάδες. Φαίνεται πως συναντιόμαστε σε διάφορα μέρη. Σήμερα λοιπόν χαίρομαι που καλωσορίζω τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να παρουσιάσει την ετήσια έκθεση για το 2010. Έχετε τυπωμένα αντίγραφα εντός αίθουσας και τα έχετε, ε, ναι, εδώ μπροστά σας, έχω το δικό μου αντίγραφο εδώ πέρα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λοιπόν θα μας πει για την νομισματική πολιτική του 2010 και τις λοιπές δραστηριότητες της, δηλαδή λειτουργίες Κεντρικής Τράπεζας, ε, δημοσιονομική σταθερότητα κτλ. Και μετά την παρουσίαση του Αντιπροέδρου θα δώσω τον λόγο για ερωτήσεις. Δεν έχουμε ορίσει ακόμα εισηγητή για την ετήσια έκθεση καθώς αποτελεί τμήμα του πακέτου διορισμών που θα συζητήσουν οι συντονιστές στις 10 Μαΐου στο Στρασβούργο. Οπότε θα περάσουμε στους ε, συντονιστές, καθώς δεν υπάρχει συγητής για ερωτήσεις. Καλώς ήρθατε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, κυρίες ε, και κύριοι βουλευτές ε, της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Είναι ευχαριστησή σήμερα να σας παρουσιάζω την ετήσια έκθεση του 2010 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που βεβαίω αποτελεί τμήμα της, ε, του τη λογοδοσία μας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι η πρώτη φορά που είμαι ενώπιον τη Επιτροπή μας, Επιτροπής σας υπό την ιδιότητα του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πρώτα απ' όλα θα αναφέρω τις ε, οικονομικές εξελίξεις του τελευταίου έτους, να εξηγήσω τις αποφάσεις μας και θα συνοψίσω την αξιολόγησή μας για τις ε, μακροοικονομικές προοπτικές και ζητώ κατανόηση για το ότι οι παρατηρήσεις μου για αυτό το τελευταίο θέμα δεν θα πρέπει να θεωρηθούν πως ε, αποτελούν ε, κάποια κρίση για το ποια θα είναι η μελλοντική μας πολιτική, καθώς βρισκόμαστε σε μια περίοδο στην οποία έχουμε αποδηλώσει ακριβώς για την μελλοντική αυτή στρατηγική. Πριν καταλήξω θα ήθελα βεβαίως να αναφερθώ στο δημοσιονομικό πλαίσιο Διακυβέρνηση Ένωση, ειδικά μετά τις εκθέσεις που υιοθέτησε η Επιτροπή και την έναρξη του τριμερού διαλόγου. Η νομισματική πολιτική το 2010 και αρχές του 2011 συνέχισε να λειτουργεί σε ένα πολύπλοκο και έντονο περιβάλλον. Είχαμε εντάσεις σε κάποια τμήματα χρηματαγορών του Μάιο του 2010 που ε, δημιούργησε νέε προκλήσει για την εξαγωγή τη νομισματική πολιτική. Από τι αρχέ του 2010 η οικονομική ανάκαμψη αυξήθηκε στην Ευρωζώνη. Αυτό κυρίως οφείλονταν στην ε, ισχυρή εξωτερική ζήτηση. Ταυτόχρονα η εγχώρια ζήτηση ενισχύθηκε στην περίοδο την οποία εξετάζουμε συνολικά μετά την μείωση 4,1% του 2009%. Το ΑΕΠ της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 1,18% το 2010. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν θετικότερο από αυτό το οποίο αναμέναμε πριν από ένα έτος. Στο μέλλον αναμένουμε την ε, οικονομία της Ευρωζώνης να υποφεληθεί από την συνεχιζόμενη παγκόσμια ανάκαμψη. Ταυτόχρονα η ιδιωτική ζήτηση πρέπει να συνεχίσει να συνεισφέρει στην οικονομική ανάκαμψη καθώς θα υποφεληθεί από τα οικονομικά μέτρα και τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για να βελτιωθεί η λειτουργία του χρηματοοικονομικού ε, τομέα. Οπότε θεωρούμε πως οι κίνδυνοι που υπάρχουν είναι γενικώ ισορροπημένοι στο πλαίσιο μιας αυξημένης ε, ασφάλειας. Όσον αφορά τις τιμές, ο πληθωρισμός αυξάνεται από αρχές ε, του 2010 και αυτό αντικατοπτρίζει κυρίως τις τιμές της παγκόσμιας των πρώτων υλών. Μιλάμε για ένα μέσο πληθωρισμό που αυξήθηκε στο 1,6% το 2010 και συνέχισε να αυξάνεται τις αρχές του 2011, έφτασε 2,7 το Μάρτιο και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Eurostat υπολογίζεται στο 2,8 τον Απρίλιο. Καθώς βεβαίως οι εγχώριες πιέσεις των τιμών ε, ακόμα είναι μέτριες, ε, αναμένουμε Πιέσει από πλευράς ε, τιμών της ενέργειας, ε, έμεσης φορολογίας, ε, καθώς υπάρχει ανάγκη δημοσιονομικής εξυγείας στα επόμενα έτη. Τέλος, η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις. Ενώ η νομισματική μας ανάλυση υποδεικνύει πώς η υποκείμενη βάση της ε, επέκτασης είναι ακόμα μέτρια. Οι προβλέψεις μας δείχνουν πως ε, δεν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πληθωρισμού. Μπορεί η ε, ρευστότητα να διευκολύνει τυχόν πιέσεις που προκύπτουν από άλλους παράγοντες. Άρα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας στη συνεδρίασή του στις 7 Απριλίου 2011 αποφάσισε να αυξήσει το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης καθώς αυτό είχε παραμείνει αμετάβλητο για δύο σχεδόν έτη σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Το βήμα αυτό ήταν αναγκαίο για να αντιμετωπίσουμε τις ε, τάσεις της ε, νομισματικής πολιτικής όσον αφορά την σταθερότητα των ε, τιμών, καθώς θα πρέπει οι πρόσφατες εξελίξεις να μην οδηγήσουν σε μεγάλες πληθωριστικές πιέσεις μέσω πρόθεσμα, μέσω δεύτερογενών επιδράσεων η απόφασή μας αυτή για την αύξηση των επιτοκίων θα οδηγήσει στο να παραμείνουν οι προσδοκίες σύμφωνες με τον στόχο μας του να παραμείνει ο πληθωρισμός μεσοπρόθεσμα κάτω αλλά κοντά στο 2% και αυτό είναι προαπαιτούμενο για να συνεισφέρει η νομισματική πολιτική στην οικονομική ανάπτυξη ιστορικά. Τα επιτόκια παραμένουν σταθερά σε ολόκληρο το φάσμα λήξης. Άρα εξακολουθούμε και εμείς να στηρίζουμε με αυτόν τον τρόπο τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη. Δεδομένων δε των εντάσεων, διατηρήσαμε κάποια από τα μη συνήθεια οικονομικά μας μέτρα το 2010 και 2011, δηλαδή την πλήρη παροχή ρευστότητα σε σταθερά επιτόκια, Επιπλέον, το Μάιο του 2010 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να ξεκινήσει το πρόγραμμα αγορών αξιογράφων για να αγοράσει ιδιωτικά και κρατικά ομόλογα για να βοηθήσει την πολιτική. Άρα εδώ πέρα βοηθήσαμε πάρα πολύ μέσω επιχειρήσεων οι οποίες απορρόφησαν την ρευστότητα. Και βεβαίως όλα αυτά τα μέτρα είναι προσωρινά από τη φύση τους και θα διορθωθούν όταν παραστεί ανάγκη. Όσον αφορά τώρα τις δημοσιονομικές πολιτικές, τα ελλείμματα και ο λόγος των ελλείμματων επιδεινώθηκαν ουσιαστικά το 2008 και 2009. Το 2010 ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ σταθεροποιήθηκε σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο γύρω στο 6% ενώ το λόγος του χρέους συνεχίστηκε συνέχισε να αυξάνει και έφτασε στο 85%. Συγκεκριμένες χώρες είχαν πάρα πολύ μεγάλους ε, ρυθμούς ελλείμματος. Αν δούμε το ζήτημα ευρύτερο, ενισχύθηκαν λόγω της ύφεσης οι ανισορροπίες οι οποίες είχαν συσσωρευτεί από πριν. Συγκεκριμένα πάρα πολλές χώρες δεν μπόρεσαν να εφαρμόσουν σε καιρούς ευμάρειας σωστές οικονομικές πολιτικές, χρησιμοποιήθηκαν προσωρινά πλεονάσματα για να χρηματοδοτηθούν μόνιμες ε, αυξήσεις δαπανών και δεν ε, μπόρεσε να γίνει σημασμό των οικονομικών παρά τις ε, μακροχρόνιες περιόδους οικονομικής ανάπτυξης. Από τη θεσμική πλευρά, το πλαίσιο το οποίο είχε αναθεωρηθεί το 2005 ήταν πολύ ασθενές και δεν είχε εφαρμοστεί και επαρκώς. Ως αποτέλεσμα αυτού, οι ψαλίδες των επιτοκίων των κρατικών ομολόγων άνοιξαν πάρα πολύ, τα σπρέτς δηλαδή, και ε, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη διακύμαση σε αυτές. Ε, υπήρχε λοιπόν πρόβλημα στην Ελλάδα και την Ιρλανδία το 2010, οι οποίες ε, χρειάστηκαν στήριξη από πρόγραμμα από κοινού Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και η Πορτογαλία επίσης τον περασμένο μήνα ζήτησε βοήθεια. Στο μέλλον, λοιπόν, είναι ε, ουσιαστική σημασία στις τρεις αυτές χώρες να αναλάβουν δραστικές μεταρρυθμίσεις. Η Ιρλανδία και η Ελλάδα πρέπει να εφαρμόσουν τα προγράμματα τα οποία έχουν συμφωνηθεί και το ίδιο ισχύει και για την Πορτογαλία. Γενικότερα όλε οι κυβερνήσει τη Ευρωζώνη θα πρέπει να επιτύχουν του στόχου μείωση του χρέου, οι οποίοι ε, στόχοι θα πρέπει να ακολουθούν από συγκεκριμένα μέτρα. Οι προθεσμίε για τη μείωση του υπερβολικού ελλείμματος που συμφωνήθηκαν στο κοφίν πρέπει να γίνουν σεβαστές. Η Εστονία και το Λουξεμβούργο είναι οι μόνες χώρες της Ευρωζώνης που αυτή τη στιγμή δεν υπόκεινται σε μια δικασία υπερβολικού ελλείμματος δεδομένων των ε, πολύ μεγάλων δάπανων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί πέρα ακριβώ θα πρέπει να επικεντρωθούν τα σχέδια αυτά για να υπάρξει εμπιστοσύνη για το ότι είναι βιώσιμα τα δημόσια οικονομικά για να βελτιωθούν οι συνθήκες ανάπτυξης. Επιπλέον βεβαίως αυτό αποτελεί και τη βάση σωστών ε, οικονομικών πολιτικών, ειδικά όταν έχουμε καιρού ευμάρες. Θα έρθω σε αυτά σε λίγο. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ σύντομα σε ζητήματα χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστημικής ε, σταθερότητας και οι τρεις ε, ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές ε, ξεκίνησαν να λειτουργούν τώρα. Η Ευρωπαϊκή Αυτή του Συστημικού Κινδύνου λειτουργεί πλήρω. Το Γενικό Συμβούλιο έχει ήδη συνεδριάσει δύο φορέ και οι συμβουλευτικέ επιτροπέ έχουν συσταθεί σε σώμα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα δώσει βεβαίω την πλήρη στήριξή τη στο Συμβούλιο αυτό. Άρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να ενισχύσει τι δυνατότητε τη και τα αναλυτικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή τη για ανάλυση συστημικού κινδύνου. Στο πλαίσιο της Βασιλείας 3 υποστηρίζουμε πλήρως το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Οδηγία Κεφαλιακών Απαιτήσεων 4. Οι προτάσεις της ε, Κομισιόν μέχρι το Μάιο του 2011 όπως προβλέπετε θα δώσουν σε Συμβούλιο και Κοινοβούλιο επαρκή χρόνο να ολοκληρώσουν το πλαίσιο μέχρι το τέλος του έτους. Η έκθεσή μας ε, τονίζει την στήριξη στην πρόταση της Κομισιόν για τη διαχείριση της κρίσης και για ένα πλαίσιο για τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Σαφώς η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται καλύτερα μέσα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τα προβλήματα στο τραπεζικό τομέα. Τα εθνικά καθιστώτα θα πρέπει να εναρμονιστούν στο μέτρο του δυνατού και να υπάρχουν προβλέψεις για καλύτερο συντονισμό μεταξύ κρατών μελών σε καταστάσεις κρίσης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συμφωνεί με το γενικότερο στόχο του νέου καθεστώτος τη Ένωσης, δηλαδή να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο εντό του οποίου μπορούν να ε, αποτύχουν ευρωπαϊκά πιστοτικά ιδρύματα, διασφαλίζοντας την σταθερότητα του ιδρύματος με τις λιγότερες δυνατές ε, ζημίες. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ένα στιβαρό πλαίσιο το οποίο έχει κέρια σημασία. Και άρα θα πρέπει στο πλαίσιο αυτό να υπάρξει ένα δίκτυο εθνικών ε, ε, ταμείων εξυγίανσης που θα συνεισφέρουν σε ένα ευρωπαϊκό τέτοιο ταμείο και αυτό έχει οπωσδήποτε πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επίσης συνεισφέρει ενεργά στις συζητήσεις ε, και στους G20 για την δημιουργία συστημάτων, για τον περιορισμό του συστημικού κινδύνου, ειδικά το μιλάμε για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν παγκόσμια συστημική σημασία όσον αφορά δε τα νέα τεστ κοπόσεως που θα γίνουν υπό την αιγίδα του νέου φορέα που έχει συσταθεί για αυτό το σκοπό θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυστηρά για να είναι αξιόπιστα. Θα πρέπει να μειωθεί η αβεβαιότητα στους συμμετέχοντες στην αγορά όσον αφορά την υγεία των ευρωπαϊκών τραπεζών. Να αναφέρω ορισμένα ε, χαρακτηριστικά ότι είναι πιο ισχυρό το μακροοικονομικό σοκ. Επίσης η EBA, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, έχει προτείνει κάποια πιο αυστηρά κριτήρια. Οι απαιτήσει έχουν γίνει πιο αυστηρέ και τα κράτη-μέλη δεσμεύτηκαν σε φιλόδοξες στρατηγικές για την ενίσχυση των ευάλωτων ιδρυμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό να υπάρχουν backstops κατάλληλα για αυτές τις τράπεζες που δεν θα περάσουν αυτά τα τεστ. Θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε τα τρεστέ στην Ευρώπη, ούτω ώστε να ξεκινήσουμε ένα πιστικό εγχείρημα ανακεφαλαιοποίησης ε, του τραπεζικού τομέα στην Ευρώπη συνολικά. Εν τέλει, θα ήθελα να συγχαρώ τη δική σας Επιτροπή που πρόσφατα ψήφισε το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης. Η Επιτροπή έκανε πράγματι έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα προς ε, την απαιτούμενη ενίσχυση της χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Συγκεκριμένα χαιρετίζω ιδιαίτερα το γεγονός ε, ότι ο αυτοματισμός των διαδικασιών έχει αναβαθμιστεί επεκτάθηκε η χρήση ε, της ανεστραμμένης ειδική πλειοψηφία. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα διαδικασίες για χώρες που παραβιάζουν κάποιους κανόνες, ε, πρέπει να ενισχυθεί και ο ρόλος της Κομισιόν και όλα τα προτινόμενα στην έκθεση του Κοινοβουλίου είναι καλοδεχούμενα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέτρα τα οποία προτείνεται, είναι απαραίτητα για να υπάρχει έγκαιρη και πρόορη συμμόρφωση με το εποπτικό πλαίσιο και θα πρέπει να εφαρμόζονται και οι οικονομικέ κυρώσει εντό ε, του μακροοικονομικού ε, εποπτικού πλαισίου. Όλα αυτά είναι προ την ίδια κατεύθυνση. Επίση, στο ίδιο πλαίσιο στηρίζουμε τη σαφή διάκριση μεταξύ κρατών μελών ε, τα οποία ανήκουν και τα οποία δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν αρνητικές ανισορροπίες και θα πρέπει να υπάρχουν μεγαλύτερε απαιτήσει για τα μέλη τη Νομισματική Ένωση. Τέτοιου είδου διακρίσει, αξιοποιώντα και το νέο άρθρο 136 τη συνθήκη, πρέπει να εφαρμοστεί σε διαφορετικού ε, τομεί και θα πρέπει να συναχθούν τα κατάλληλα συμπεράσματα μετά την κρίση για τη λειτουργία τη Νομισματική Ένωση. Ε, Τέλο, ε, η συμμόρφωση των κρατών μελών με τι υποχρεώσει και με το πακέτο σταθερότητα και ανάπτυξη διευκολύνεται με το ισχυρά δημοσιονομικά πλαίσια τα οποία θέλετε να εγκαθιδρύσετε εντό τη Ευρωζώνης, προτείνοντας ε, συγκεκριμένα υποχρεωτικά χαρακτηριστικά. Η πρόταση οικονομικών κυρώσεων για, την, ε, ε, για το χειρισμό δεδομένων είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό αν θέλουμε να έχουμε έγκαιρα αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία. Ταυτόχρονα υπάρχουν κάποιες πτυχές ε, της θέσης της Επιτροπής σας για τις οποίες έχουμε κάποιες ανησυχίες. Πιο σημαντικό θέμα είναι ότι το πακέτο σταδερότητας και ανάπτυξης δεν θα πρέπει να έχει περισσότερες εξαιρέσεις και μακρύτερους καταλόγους σε αιτικών συναφών παραγόντων, κυκλικές εξελίξεις, παραδείγματο χάρη, δημο, ε, δημόσιες επενδύσεις, κρατικά μέτρα για το χρηματοπιστωτικό τομέα, τα οποία θα πρέπει να ε, μπορεί να επικαλείται κανείς ό,τι αφορά τη μη σε προς τα στοιχεία, ε, τα κριτήρια του χρέους και του ελλείμματος γιατί αυτό μπορεί να ανοίξει την ε, πόρτα σε κάποια φορολογικά μέτρα, εκεί που όμω απαιτείται δημοσιονομική εξήγηση. Ό,τι αφορά τη μακροοικονομική εποπτεία, πολλέ φορέ έχουμε τονίσει ότι για να υπάρχει αποτελεσματικότητα θα πρέπει να υπάρχει εστίαση σε έναν περιορισμένο ρυθμό δικτών που θα συλλέγουν ε, κάποιε μακροοικονομικέ ανισορροπίε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιλάμε ακριβώ στι μακροοικονομικές ανισορροπίε. Δηλαδή πρέπει να βλέπουμε αν υπάρχει σημαντική απόκληση από μια δεδομένη τάση, αν υπάρχουν ανισορροπίε οι οποίε απειλούν την ίδια τη λειτουργία τη Νομισματική Ένωση. Δεν μιλάμε τώρα να επιτευχθεί ένα δυναμικό υψηλό ανάπτυξη. Φυσικά και αυτό βέβαια είναι ευκταίο, είναι και ένα από του στόχου ε, τη στρατηγική 2020. Δεν εννοώ ότι δεν αναγνωρίζουμε την ανάγκη να υπάρχει συντονισμό μεταξύ όλων των πτυχών τη οικονομική πολιτική υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η έκθεση που εγκρίνει η Επιτροπή σας είναι πολύ θετικό μήνυμα εν ώψη του τριμερούς διαλόγου που ακολουθεί και ελπίζω να ολοκληρωθεί σύντομα το πακέτο αυτό ώστε να εγκριθεί το πακέτο οικονομικής δικυβέρνησης και να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, τα μαθήματα που έχουμε αντλήσει από τη χρηματοπιστωτική κρίση είναι αυτά τα οποία ε, οδήγησαν και στις ευρείες μεταρρυθμίσεις που έγιναν. Επικεντρωθήκαμε πέρυσι ε, στην κρίση αυτή που έδειξε ότι υπάρχει ζήτημα με το δημόσιο χρέος, ε, με το χρηματοπιστωτικό τομέα που είναι οι δύο πτυχές, οι δύο όψεις του, της κρίσης. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας ενδέχεται πολλές φορές να επηρεάσει αρνητικά τα δημόσια οικονομικά ενώ οι μακροανισορροπίες και οι δημοσιονομικές πολιτικές μπορούν επίσης να επηρεάσουν αρνητικά το χρηματοπιστωτικό τομέα. Πρέπει να επιληθούν λοιπόν και τα δύο θέματα γιατί έτσι η Ευρωζώνη θα μπορέσει να ξεκινήσει μια νέα πορεία για βιώσιμη ανάπτυξη και να αφήσει πίσω τα προβλήματα τα σημερινά. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει αποτελεσματική οικονομική διακυβέρνηση για να υπάρχει δημοσιονομική βιωσιμότητα, ανταγωνιστικότητα, ανάπτυξη θα πρέπει λοιπόν ο μόνιμος ε, μηχανισμός σταθερότητας να οριστικοποιηθεί και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά τα ευρωπαϊκά συστήματα χρηματοοικονομικής εποπτείας. Σε όλες αυτές τις προσπάθειες ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, μοιράζονται τους ίδιους στόχους, τις ίδιες αξίες και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουν να συνεργάζονται ώστε να στεφθεί με επιτυχία το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Ευχαριστώ. Thank uh, Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, έχουμε μόνο 25 λεπτά στη διάθεσή μας ε, και πρέπει να τελειώσουμε και στην ώρα μας γιατί εγώ έχω μια άλλη μεν υποχρέωση. Ε, και αυτή τη στιγμή έχω την κυρία Ποντήματα και την κυρία Φερέρα εκτός από τους συντονιστές. Δεν ξέρω αν θέλει και κάποιος άλλος να λάβει το λόγο γιατί πραγματικά πρέπει να κλείσουμε τον κατάλογο των ερωτώντων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν ξέρω αν ε, κατάλαβα καλά, αλλά ε, νομίζω ότι ουσιαστικά μας τα παρουσιάσετε αισιόδοξα τα πράγματα, τουλάχιστον δεν άκουσα να κρούεται κάποιον κόδωνα κινδύνου. Θέλω να σας θέσω δύο ερωτήματα. Πρώτον, τι γίνεται με τις έκτακτες παρεμβάσεις της ΕΚΤΑ που ε, ήταν αρκετά τρέχουσε, θα έλεγα, τον τελευταίο καιρό για στήριξη του ευρώ. Και δεύτερον, ότι πρέπει να σκεφτούμε για τις φήμες που κυκλοφορούν, ε, για ενδεχόμενη πιθανή ε, μελλοντική διάρθρωση του ελληνικού χρέους. Ευχαριστώ. θα απαντήσουμε σε την ερώτηση. Ερώτηση απάντηση καλύτερα να πηγαίνει έτσι. είναι πολύ δύσκολο. να βρει κανεί ε, το κατάλληλο ύφο ε, για να μπορούν και οι ελεγκτέ να γνωρίζουν κατά πόσο το ύφο είναι θετικό ή απεσιόδοξο. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Πρέπει να δούμε το επίπεδο των spread, το χρέος ε, πολλών κρατών, το δημόσιο χρέος και έτσι καταλήγουμε ότι όλα αυτά ήταν εκείνα που οδήγησαν στην κρίση του ε, Μαΐου. Τα μέτρα που λήφθησαν και από τις ενδιαφερόμενες χώρες ε, και από την Ευρωζώνη δεν έχουν ακόμα πείσει την αγορά ότι τα μέτρα αυτά είναι αρκετά για να αντιμετωπίσουν επιτυχώς ε, το πρόβλημα χρέους. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό γιατί ήδη έχουν ληφθεί πολύ τολμηρές αποφάσεις και αυτές οι τολμηρές αποφάσεις δεν αξιολογήθηκαν ε, σωστά, δεν εκτιμήθηκαν από τους οίκους ε, αξιολόγησης γιατί το ποσό της ε, βοήθειας που χορηγήθηκε, αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος χρέους έχει μειωθεί. Γι' αυτό χορηγήθηκε η βοήθεια. Αυτό όμω δεν εκφράζεται μέσα από την αξιολόγηση των οίκων αξιολόγηση. Κάθε άλλο, αντίθετα, αμέσως μετά την ανακοίνωση χορήγηση βοήθεια, οι χώρες υποτιμήθηκαν ακόμα περισσότερο στην κατηγορία αξιολόγησης. Οι κράσεις λοιπόν, η κρίση, η κρίση υφίσταται ακόμα και είναι πάρα πολύ σοβαρή. Όσον αφορά τώρα τα μέτρα που λάβαμε πέρυσι, τα μέτρα αυτά εκτοτε ε, χρησιμοποιήθηκαν και αντιστοιχούν περίπου στο 12% της ε, συνολικής ε, παροχής ε, ρευστότητας. Μιλάμε για μια τέτοια τάξη μεγέθους. Το πρόγραμμα δεν ενεργοποιείται εδώ και κάποιο καιρό. Το πρόγραμμα δεν έχει καταργηθεί, αλλά δεν χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή. Αυτό έχω να σας πω ως ε, μια βοήθεια, ενδεχόμενη βοήθεια εξόδου από την κρίση. Προφανώς το μέτρο από τη φύση του είναι προσωρινό και παραμένουμε σε αυτή τη θέση. Το μέτρο προφανώς παροχής βοήθειας. Και ένας από τους λόγους που δεν χρησιμοποιούμε σε αυτή τη φάση το μέτρο αυτό είναι ότι ένα κομμάτι των αυξήσεων στα spread πρόσφατα ήταν το αποτέλεσμα που αναφέρετε κι εσείς και κυκλοφορούν σχετικά με την αναδιάρθρωση του χρέους. Και ενώ οι φήμες αυτές διαψεύστηκαν από πολύ σημαντικές προσωπικότητες και κυβερνήσεις, παρόλο αυτά οι φήμες εξακολουθούν να κυκλοφορούν. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί ε, δυστυχώς ε, και μεμονωμένα άτομα και θεσμοί που επιθυμούν να διατηρήσουν την κυκλοφορία αυτών των φημών. Γιατί αν τελικά υπάρξει αναδιάρθρωση στην Ευρωζώνη, οι κύκλοι αυτοί θα υποφεληθούν, θα κερδίσουν. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει κανείς αυτές τις τελευταίες εξελίξεις. Εξάλλου, οι περισσότερο ευάλωτες χώρες, ε, είτε είναι ήδη μέσα σε ένα πρόγραμμα, είτε ζήτησαν παροχή βοήθειας, όπως η Πορτογαλία. Όσον αφορά την αναδιάρθρωση χρέους, γνωρίζετε τη θέση μας. Η θέση μας είναι ότι εφαρμόζονται προγράμματα. Τα προγράμματα ε, προβλέφτηκαν σε συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, υφίστανται πρέπει να εφαρμόζονται και να υπάρχει η απαραίτητη συμμόρφωση. Βεβαίως, ε, από τη φύση τους τα προγράμματα δεν είναι θέσφατα, ανανεώνονται και αναθεωρούνται. Πάντως πρέπει να συμμορφωνόμαστε με τα προγράμματα, να παραμένουμε πιστοί στα προγράμματα και να μην δημιουργούμε εκ των προτέρων την εντύπωση ότι τα προγράμματα θα αποτύχουν. Η Κέι είναι ο επόμενος συντονιστής που βλέπω η επόμενη Ίστρια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Ελπίζω. Αλλά αναφερθήκατε στα ταμεία εξυγένσης, resolution funds. Είχα ρωτήσει πριν τους αντιπροέδρους ε, του, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συστημικού Κινδύνου νωρίτερα αν θεωρούν ότι υπάρχει επαρκές κεφάλαιο ε, που να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε ε, αυτά τα ταμεία, να βάλουμε δηλαδή κάποια κεφάλαια κατά μέρος. Εσείς πιστεύετε ότι ισχύει, υπάρχει επαρκές κεφάλαιο το οποίο ε, υπάρχει στο σύστημα δεδομένου του σωρευτικού αποτέλεσματος όλων των ρυθμίσεων που έχουμε, ώστε να έχουμε αυτό το Ταμείο Εξυγίανσης για τα 27 κράτη-μέλη. Yes, that's precisely... Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Από τότε που άρχισε να γίνεται λόγος για την φορολόγηση στον τραπεζικό τομέα, εμείς είπαμε ότι πρέπει να επικρατήσει σύνεση με την έννοια ότι όλα πρέπει να είναι σωστά σταθμισμένα έτσι ώστε να μπορέσουμε το βάρος που προκύπτει για τον τομέα να διοχετευτεί σε πιο χρήσιμους Χρήσιμε διόδους. Όσον αφορά τώρα τα ταμεία εξυγίανσης, πολλές φορές που επιβλήθηκαν σε πολλά κράτη-μέλη θα πρέπει να αναδιοχετευτούν σε ένα τέτοιο είδος ταμείο εξυγίανσης που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο. Ένα στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό έτσι ώστε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής και τραπεζικής κρίσης στην Ευρώπη. Βεβαίως, η οικονομική κρίση και η εξυγίανση των θεσμών, κυρίως η εξυγίανση των θεσμών, είναι καθοριστικό στοιχείο της κρίσης. Και ένας βασικός στόχος είναι να μειωθούν οι ζημιές, να αποφευθεί η επιμόλυνση, να επιτευχθεί η προστασία των φορολογουμένων και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τα μη εξυγίανσης εκ των προτέρων πριν χρειαστούν. Εξάλλου αυτό το δίκτυο ταμείων εξυγίανσης ε, που θα συσταθεί με βάση την πρόταση Κομισιόν, αν βέβαια αυτή εγκριθεί, αυτό το δίκτυο των Εθνικών Ταμείων Εξυγίανσης θα μπορούσε μετά να μετεξελιχθεί σε ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξυγίανσης, το οποίο θα βοηθούσε πάρα πολύ στο να αντιμετωπιστεί αυτό το τόσο δύσκολο πρόβλημα του επιμερισμού του βάρους ε, σε περίπτωση ε, κρίσης ε, διασυνοριακής κρίσης που δεν πλήττει μόνο ένα κράτος. Ε, νομίζω ότι πρέπει το πρόβλημα να λυθεί άπαξ διαπαντός, διότι η ύπαρξη αυτού του προβλήματος παρεμποδίζει την περαιτέρω πρόοδο σε αυτό που εμείς αποκαλούμε έλεγχο, έλεγχος ο οποίος λαμβάνει υπόψη του την ευρωπαϊκή προοπτική και το ενδεχόμενο να επιμολυνθεί μια χώρα, όπως λέμε, από μια προηγούμενη. Ο Σβέν. Ευχαριστώ που μας δώσατε την ετήσια έκθεσή σας και σας ευχαριστώ που ήρθατε. Είναι πολύ σημαντικό να μελετάει κανείς το δύσκολη δουλειά σας. Δεν ξέρω αν θα ήθελα τη δουλειά σας αυτή τη στιγμή. Δύο ερωτήσεις έχω. Η πρώτη είναι η εξής η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έλαβε σκληρά μέτρα για να δώσει στις τράπεζες ε, την απαιτούμενη ρευστότητα και αποδέχτηκε ε, εγγυήσεις όχι τόσο ισχυρές σε αντάλλαγμα. Είδαμε λοιπόν τη συσσόρευση στοιχείων ε, παυτικού Στου ε, λογαριασμού τη. Επίσης παρεμβαίνει στη δευτερογενή αγορά αγοράζοντας ε, κάποια συγκεκριμένα προϊόντα. Οπότε το ερώτημά μου είναι πώς, ε, τι προβλέπετε να κάνετε για τον κίνδυνο που έχετε αναλάβει εάν δείτε το πώς αξιολογούν οι αγορές τα διάφορα αξιόγραφα τα οποία έχετε δεχτεί ως εγγύηση και αγοράστε από τη δευτερογενή αγορά. Υπάρχει ένας υπολογισμός πόσο κίνδυνο έχετε αναλάβει και πώ αντικατοπτρίζετε αυτό στους ετήσιου λογαριασμού σας. Επίσης αναρωτιέμαι, ε, δείχνετε εδώ πέρα στη σελίδα 233 της έκθεσης πως έχετε κέρδος. Ακόμα και από αυτές τις ε, συνθήκες ε, μοιράσατε κέρδη στις εθνικές κεντρικές τράπεζες και αναρωτιέμαι αυτή η διανομή κερδών πώς κολλάει με τον πιθανό κίνδυνο. Και δεύτερον, όπως εξηγήσατε, μειώσατε κατά πολύ τα επιτόκια κατά τη διάρκεια της κρίσης και τώρα κάνετε το πρώτο βήμα για να φύγετε από αυτή την κατάσταση βεβαίως και ταυτόχρονα εξηγείτε πως δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σημάδια Αύξηση ε, του βασικού πληθωρισμού, αλλά βεβαίω ε, βλέπετε πως είστε υπέρ ε, των αυξήσεων φόρων και είπατε πως θα αυξηθούν τιμές της ενέργειας και των βασικών πόρων. Εάν παρόλα αυτά αυξήσετε και τα επιτόκια που θα δυσκολεύσουν τα ασθενέστερα μέρη της Ευρωζώνης, ενώ είναι ταυτόχρονα αναγκαίο κάτι τέτοιο σε άλλα σημεία της Ευρωζώνης, μήπως αυτό αμφισβητεί τον ορισμό του πληθωρισμού που χρησιμοποιείται. Μήπως θα μπορούσατε να συμπεριλαμβάνετε και το ζήτημα των ε, τιμών των ε, πόρων ε, όσον αφορά το τι ορίζετε εσείς ως πληθωριστικές πύρες. Okay, thank you uh, for your... Σας ευχαριστώ για το ερώτημα που μου βάλατε. Ακούστε, σε ό,τι αφορά τους κινδύνους, που είναι το πρώτο σας ερώτημα, Καταρχάς, η κίνδυνη πιο σημαντική στον τομέα των αγορών. Μιλάμε για την αγορά αξιογράφων και το σχετικό πρόγραμμα. 77 δις αριθμοί αυτή τη στιγμή και το πρόγραμμα των ε, ομολόγων, καλυμμένων ομολόγων, 60 δις. Σε ό,τι αφορά τα covered bonds, η ανταπόκριση για αυτά τα ομόλογα, όχι μόνο για τα περιουσιακά στοιχεία που είναι πίσω από αυτά τα ομόλογα, αλλά και οι τράπεζες που έχουν εκδώσει τα ομόλογα και που φυσικά είναι και υπεύθυνε, και σε ό,τι αφορά τον S&P, ξέρετε ότι υπάρχουν προγράμματα για κάποιες από τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα και αυτό σημαίνει ότι βασιζόμαστε στην επιτυχή υλοποίηση των προγραμμάτων αυτό. ώστε στο τέλος αυτά τα αξιόγραφα να πληρωθούν. Αγοράστηκαν στη δευτερογενή αγορά, ήδη με μεγάλη μείωση, οφείλω να σας επισημάνω. Κάτω δηλαδή από την ονομαστική αξία και στο μεταξύ πήραμε και πολλές πληρωμές ε, επιτοκίων Μιλάμε για εκατοντάδες ε, χιλιάδες ευρώ. Τώρα, εκτός αυτού μας προστατεύει ήδη το γεγονός ότι αγοράσαμε, όπως σας είπα, αυτά τα προϊόντα στη δευτερογενή αγορά με μείωση και έχουμε λάβει και κάποια, εσπράξει κάποιους στόκους και αυξήσαμε και τις ε, γενικές μας προβλέψεις κατά πολύ για την αντιμετώπιση των κινδύνων. Όχι μόνο το κεφάλαιο της ΕΚΤ διπλασιάστηκε, αλλά χρησιμοποιήσαμε επίσης και πολλά από τα κέρδη, ακριβώς για το προηγούμενο έτος μιλάω, τα κέρδη του προηγούμενου έτος για να αυξήσουμε τις γενικές προβλέψεις κατά πάνω από 5 δις ευρώ. Άρα μιλάμε για σημαντική αύξηση των προβλέψεων, που και αυτό είναι ένα προστατευτικό δίχτυ για κινδύνους που ενδέχεται να ανακύψουν στο μέλλον. Διαπλασιασμός του κεφαλαίου επίσης είναι ένα μέτρο που κατά την άποψή μας φροντίζει να λέμε υπόψη του μελλοντικού κινδύνου. Διανύμαμε μεν τα κέρδη, αλλά σε μικρό βαθμό, γιατί το μεγαλύτερο μέρο των κερδών ουσιαστικά πήγε στην αύξηση των γενικών προβλέψεων τη ΕΚΤ. Σε ό,τι αφορά τώρα τον πληθωρισμό, και αυτό που είπατε για το βασικό πληθωρισμό και τις διαφορετικές καταστάσεις στα διαφορετικά κράτη της Ευρωζώνης. Φυσικά γνωρίζετε ότι η συνθήκη είναι σαφής σε ό,τι αφορά την πρωταρχική εντολή του συστήματος του ευρώ είναι κάτι που γνωρίζουμε και βέβαια πρέπει την εντολή μας να την σεβαστούμε και να τηρήσουμε τις διατάξεις της συνθήκης σε ό,τι αφορά το μέσο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Έτσι γίνεται σε όλες τις νομισματικές ενώσεις ανά τον κόσμο. Μιλήστε για το βασικό πληθωρισμό που είναι πράγματι είναι με, ε, υποέλεγχο, είναι λίγο πάνω από το 1%. Αν βγάλουμε έξω την ενέργεια και τα μεταποιημένα τρόφιμα, αλλά ο βασικός πληθωρισμός δεν είναι στόχος για την νομισματική μας πολιτική. Ξέρετε ότι είπα, για να σας αναφέρω ένα πολύ γνωστό παράδειγμα, χρησιμοποιεί αυτή την έννοια γιατί μπορεί οικονομετρικά να φανεί ότι στη ΣΥΠΑ ο βασικός πληθωρισμός είναι ένας καλός βασικός δείκτης για τον μελλοντικό headline inflation. Αλλά δεν έχουμε αντίστοιχη εφαρμογή αυτού του δείκτη στην Ευρώπη. Ίσως λοιπόν δεν ξέρω αν θα πρέπει να πάρουμε τον βασικό πληθωρισμό ως βασικό ε, στόχο της νοσηματικής πολιτικής. Ε, μας είπατε ότι έχουμε πρόβλεψη, σας είπα μάλλον ότι έχουμε πρόβλεψη 2,8 πληθωρισμό στις τελευταίες ε, εκτιμήσεις της Eurostat για τον Απρίλιο. Πρέπει να δούμε τι γίνεται. για να σταθεροποιηθούν οι εκτιμήσεις ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Ιστορικά τα επιτόκια συνεχίζουν να είναι πολύ χαμηλά και όπως είπε ο πρόεδρος Τρισέ στην ε, συνέντευξη τύπου όταν αποφασίσαμε να αυξήσουμε κατά 0,25% δεν αποφασίσαμε να σπεύσουμε σε άλλες ε, αυξήσεις στο μέλλον. Έχουμε μόνο 7 λεπτά η και ε, μετά θα δώσω το λόγο σε έναν ακόμα συνάδελφο. Thank Sharon, you, uh, Ευχαριστώ πολύ, Sharon. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Έχω δύο πολύ σύντομε ερωτήσει. Μία έχει σχέση με αυτό που ρώτησε ο Ζαν Πόλη σχετικά με την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους και είμαι ευγνώμων για την απάντησή σας. Είπατε ότι έχουν διαψευστεί οι φήμες αλλά είπατε ότι εξακολουθούν να κυκλοφορούν οι φήμες αυτές γιατί ε, κάποιοι κύκλοι κερδίζουν με αυτές τις φήμες. Το θέμα είναι το εξής. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γιατί δεν είναι ότι απλά υπάρχουν. Αυτές οι φήμες υπονομεύουν αυτή την ε, επώδυνη προσπάθεια του λαού και της κυβέρνησης για την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών της Ελλάδας. Μετά, αυτό που είπατε σχετικά με την απόφασή σας της 7 Απριλίου για την αύξηση των επιτοκίων της ε, Κεντρικής Τράπεζας, της ΕΚΤ. Ε, είμαι σίγουρη ότι ασκήθηκε κριτική σε αυτή την απόφαση, γιατί η ανάκαμψη δεν έχει επανέλθει πλήρως ε, και η απόφαση αυτή μπορεί να υπονομεύσει την οικονομία ορισμένων κρατών. Εξάλλου αναφέρθηκε ότι η απόφαση αυτή να αυξηθούν τα ε, βασικά επιτόκια που καθιστά το χρήμα και πάλι πιο ακριβό, η απόφαση αυτή ε, δυσχεραίνει περαιτέρω ε, τις προσπάθειες κρατών που προσπαθούν να εξηγειάνουν όπως είπαμε, τα δημόσια οικονομικά τους. Η Ελίζα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τον τρόπο ε, για τον οποίο δραστηριοποιηθήκατε στην κρίση. Η κρίση δεν έχει ακόμα ε, παρέλθει και έχω δύο ερώτησεις. μία φορά την Ελλάδα. Αναφέρθηκε ότι η κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς παρά την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η δική μου ερώτηση έχει σχέση με το εξής. διαπιστώθηκε ότι η επιδείνωση αυτή οφείλεται μεταξύ άλλων στο ότι η ανάπτυξη και μακροπρόθεσμα και μικροπρόθεσμα θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί και τα μέτρα της σταθεροποίησης αξιολογούνται μικρο, βράχι πρόθεσμα. Έχουμε τα μέτρα τα παρεμβατικά του Διεθνούς Εναμισματικού Ταμείου, ε, της Τρόικα. Πολλές φορές όμως ε, τα μέτρα αυτά σχετίζονται με μία κρίση σε μία χώρα η οποία μπορεί να αποβεί και μοιραία, μπορεί να, αποβεί, να καταλήξει τη χρεοκοπία. υπήρξαν μέτρα στήριξη από μεμονωμένες κυβερνήσει, αλλά όχι ευρωπαϊκά μέτρα. Εσείς τι πιστεύετε, τι μπορεί κανείς να μάθει από το πάθημα της Ελλάδας, τι μπορεί να, μάθει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από την Ελλάδα για αυτά που θα εφαρμόσει στην Πορτογαλία. Και τι μπορεί κανείς να μάθει από το συγκεκριμένο πακέτο μέτρων. Ήταν η πρώτη μου ερώτηση. Και η δεύτερη έχει σχέση με το εξής. Πώς πρέπει να αξιολογείτε να αξιολογούνται τα περιουσιακά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε σχέση ε, με, ε, ε, με το χρέος των κρατών. Άλλα τέσσερα λεπτά έχουμε μόνο. δεν μπορώ δυστυχώς, γιατί εγώ έχω μια άλλη υποχρέωση, πρέπει να φύγω και έχετε εσείς το λόγο. Oh, yes. Ε, the floor is mine. Α, ναι, ναι. Έχω το λόγο, ναι. Και για την αναδιάρθρωση, τις φήμες ε, και τις δυσκολίε που δημιουργούν και τι μπορεί να γίνει. Σε αυτή τη συγκυρία, αυτό το οποίο μπορεί να γίνει είναι να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε την αντίληψη αξιοπιστίας του προγράμματος που εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Υπήρξε μια σοβαρή διαρθρωτική προσαρμογή, αλλά ταυτόχρονα υπήρχαν ε, κάποιες, ε, κάποια προβλήματα που βασικά οφείλονται στα μειωμένα έσοδα και τώρα πρέπει να ε, γίνει πιο έντονο το πρόγραμμα για να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Δεύτερον, αυτά τα οποία ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση όσον αφορά τολμηρά και μεγάλα προγράμματα ιδιωτικοποίησεων πρέπει να εφαρμοστούν κιόλα. Και οι αγορές πρέπει να πιστούν πως ε, το πρόγραμμα αυτό θα εφαρμοστεί με τρόπο σοβαρό γιατί αυτό βεβαίω μπορεί να συνεισφέρει στο να μειωθεί ο λόγος χρέους τη Ελλάδας. Και αυτό από μόνο του πρέπει και θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αξιολόγηση κάνει οποιοδήποτε των δυνατοτήτων επιτυχίας ε, του προγράμματος προσαρμογής Ελλάδας. Και βεβαίως γνωρίζουμε πως η προσαρμογή αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί για, κάποιο καιρό, γιατί δεν θα γίνει σε δύο χρόνια ή σε ενάμιση και η Ελλάδα δεν έχει ακόμα επιτύχει πρωτογενές πλεόνασμα. Και άρα είναι σημαντικό και οι μεσοπρόθεσμες ε, προοπτικές που θα παρουσιάσει η ελληνική κυβέρνηση να είναι πιστικές υπό την έννοια ότι θα δείχνουν πως τα δημόσια οικονομικά πηγαίνουν προς την κατεύθυνση πλέον άσματος. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν είναι σημαντικά. Βεβαίως σημαντικό είναι να μπορούμε να σταματήσουμε τις φήμες αυτές. Αν και αυτό είναι πολύ δύσκολο, γνωρίζουμε όλοι πω κατά κάποιο τρόπο αυτά ξεκίνησαν ε, πέρυσι τον Οκτώβριο. Και το βλέπουμε αυτό και στους δείκτες της αγοράς, πως μετά από αυτό τα, πάντα ανέβηκαν. Γιατί για, για κάποιο χρονικό διάστημα υπήρχε η ερμηνεία πως τα ευρωπαϊκά προγράμματα θα ζητούσαν κάποια εκ των προτέρων συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Αυτό ξεκαθάρισε 28 ε, Οκτωβρίου από το ΕΚΟΦΗΝ και μετά εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 16 Δεκεμβρίου, αλλά παρόλα αυτά το τζιν είχε βγει από το μπουκάλι και δεν ξαναμπήκε ποτέ έκτοτε και υποφέρουμε ως αποτέλεσμα αυτού. Οπότε η ενίσχυση της αξιοπιστίας του προγράμματος και το πρόγραμμα ιδιωτικοποίησεων είναι τα στοιχεία που έχουμε τώρα στη διάθεσή μας για να αντιστρέψουμε την κατάσταση. Όσον αφορά την ε, αύξηση επιτοκίων και τις συνέπειες που αναφέρατε, όπως είπα, ε, Κοιτάξτε, εμεί λαμβάνουμε αποφάσει με βάση, όπω σα είπα, μόνο το, το μέσο όρο και εδώ περιέρχομαι στην απάντηση στη δική σα ερώτηση. Γιατί εκεί που είδατε κάποια αισιοδοξία, αυτό οφείλεται στο ότι στην πραγματικότητα η κατάσταση αυτή της κρίσης ε, που επηρεάζει κάποιες ε, χώρες μέλη δεν έχει εκτροχιάσει την ανάκαμψη στην Ευρωζώνη συνολικά. Υπάρχει μια παγκόσμια ανάκαμψη, όχι φοβερή, ήπια, αλλά υπάρχει. Και συνεχίζεται και η Ευρωζώνη συνολικά πέρσι αναπτύχθηκε περισσότερο από όσο περιμέναμε πριν από λίγους μήνες και συνεχίζει. Οπότε, από μια έννοια, βλέπουμε πως τα στοιχεία κρίσης που υπάρχουν και είναι πολύ σοβαρά δεν εκτροχιάζουν την ανάκαμψη συνολικά της Ευρωζώνης. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την πολιτική μας ε, όταν ο πληθωρισμός ε, αυξάνεται όπως αυξάνεται. Και αυτό είναι ένα στοιχείο αισιοδοξία ε, στην αξιολόγησή μου. Να μην μειώσουμε δηλαδή γενικά την κατάσταση με βάση κάποια στοιχεία κρίσης που υπάρχουν στην Ευρωζώνη. Τώρα για την ερώτηση της κυρίας Ελίζα Φερέιρα. Πάντα είναι πολύ δύσκολο να πούμε σε ένα πρόγραμμα προσαρμογή το που βρίσκεται η χρυσή τομή δηλαδή μεταξύ της υπερβολής και της απαραίτητης ε, προσαρμογής. Και πάντα βεβαίως μπορεί να κάνει λάθος κανείς και προς τη μία κατεύθυνση και προς την άλλη αλλά βεβαίως ε, αυτό είναι κάτι το οποίο η Τρόικα εξετάζει προσεκτικά. Μπορεί να σφάλουν Ο καθένας μπορεί να κάνει λάθη βεβαίως, αλλά το εξετάζουμε αυτό. Και όταν τα προγράμματα συντάσσονται, προσπαθούν να βρουν ακριβώς ε, την ισορροπία αυτή μεταξύ των διαφόρων στόχων και είδατε πως στην περίπτωση του προγράμματος ε, της Ελλάδας και της Ιρλανδίας στο τέλος των προγραμμάτων υπήρχε η πρόβλεψη πως ε, θα είχαμε ήδη θετική ανάπτυξη μετά τον αρχικό αντίκτυπο βεβαίως τον αναπόφευκτο της προσαρμογής δεδομένης της κατάστασης. Οπότε το ίδιο θα ισχύσει και στην περίπτωση της Πορτογαλίας. Και αναλαμβάνουμε βεβαίω υπόψη αυτό το γεγονός. Όσον αφορά τα τεστ αυτά κοπόσεως ή και τυχόν ε, ψαλίδισμα των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών, Κάναμε μία ανάλυση πέρσι και είπαμε πως δεν θα είναι σωστό για τις αρχές ε, να ορίσουν αυτές ποιο θα είναι το τυχόν ψαλίδισμα που θα γίνει στα στοιχεία αυτά του ενεργητικού που βεβαίως αντιβαίνει και με τη δική μας τη θέση ότι τα προγράμματα τελικά θα επιτύχουν δηλαδή. Θα εφαρμοστούν επιτυχώς και δεν θα οδηγήσουν σε ε, αναδιάρθρωση. Οπότε, ταυτόχρονα Δώσαμε στην αγορά όλες τις πληροφορίες, τις απαραίτητες για τους αναλυτές, επενδυτικές τράπεζες, επενδυτές, να κάνουν εύκολα τους υπολογισμούς. Και αυτό θα γίνει και αυτή τη φορά πολύ περισσότερο, γιατί δεν μιλάμε μόνο για την έκθεση της κάθε τράπεζας, αλλά και η λήξη της ε, έκθεσης. Ε, ο χρόνος λήξη και αυτό θα διευκολύνει βεβαίω ε, του αναλυτέ να υπολογιστούν αντίκτυπο. Σα ευχαριστώ που δώσατε τόσο ακριβείς απαντήσει στα ερωτήματα. Ευχαριστώ του ε, διερμηνεί, ε, γιατί υπέρβηκαμε λίγο το χρόνο. Αλλά ε, πρέπει να δοθούν συγκεκριμένε και ακριβείς απαντήσει. δεν μπορούσα να κόψω την απάντηση που θα δίνατε στη συμπατριώτησά σα την Ελίζα. Να σα πω ότι η επόμενη συνάντηση τη Επιτροπή μα στην Εδρίαση είναι η 9η Μαΐου, μέρα τη Ευρώπη από τις 7 ως 9 το βράδυ στο Στρασβούργο. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ.